Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich darf heute die Sitzung leiten und möchte unsere Καλώς ήρθατε και σε σχέση και με την, τον πρόεδρο και την κυρία Χρύμνε που για λόγους ε, μεταφοράς ε, κυκλοφορίας δεν μπορούν να είναι παρόντες, θα έρθουν υστερότερα. Χαιρόμαστε ότι έχουμε κάποιους φιλοξενουμένους εδώ τον κύριο Τζον Κάμινς πρώτα, τον πρόεδρο της νοτιοανατολικής Ιρλανδικής Διοίκησης που θα ενημερωθεί και θα εξοικειωθεί με τα θέματά μας. Καλώς ήρθατε. Επίσης έχουμε μια ομάδα επισκεπτών από το Περιφερειακό Κοινοβούλιο της Αξονίας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων που παρακολουθούν αυτήν. Καλώ ήρθατε όλοι οι φιλοξενούμενοι που βρίσκεστε στην Ευρωβουλή και μα έχετε επισκεφθεί. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα στη συνέχεια, διότι ο κυριότερος, η κυριότερη προσωπικότητα της σημερινής πρωινής συνεδρίασης είναι παρόν, δηλαδή ο Επίτροπος για τα Περιφερειακά Θέματα, κύριος Ιωάννης Χάν. Κύριε Χάν, καλώς ήρθατε θερμά σε αυτή τη συνεδρίασή μας σήμερα εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Έχουμε κάποια αρκετά θέματα να συζητήσουμε μαζί σας, όπου θα έλεγα ουσιοδός στα ουσιοδέστερα με τις θέσεις του Κοινοβουλίου μπορείτε να είσαστε ικανοποιημένος. Είτε πρόκειται για την έκθεση Σάνσες, είτε για την έκθεση για το μέλλον της διαρθρωτικής πολιτικής μετά το 2013. Παρ' όλα αυτά προσδοκούμε και προσβλέπουμε να δούμε και να ακούσουμε πώς εσείς τις προτάσεις του Κοινοβουλίου τις αντιμετωπίζετε. Χαιρόμαστε ήδη για τα όσα θα μας πείτε και μετά θα έχουμε κάθε ευκαιρία για συζήτηση. Κύριε Πίτροπε, έχετε τον λόγο παρακαλώ. Θα Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση σήμερα να είμαι εδώ παρόν στη συνεδρίασή σας, στην Επιτροπή σας και να τοποθετηθώ ας το πω σε μια πρώτη φάση. Και φυσικά <clears throat> για το ότι θα μπορέσουμε και να συζητήσουμε για τα θέματα του δημοσιονομικού πλαισίου για συναφή θέματα. Όμως, ακόμα είναι πρόημο θα έλεγα να κάνουμε κάτι τέτοιο. Επί της ουσίας για τις προοπτικές υπάρχει μια σειρά θεμάτων που μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις σίγουρα. Και αυτή την ευκαιρία νομίζω θα έπρεπε να την εκμεταλλευτούμε από κοινού και εσείς και εμείς. Θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές των τελευταίων μηνών που συνέταξαν εκθέσεις, αλλά κυρίως ε, εσένα Μάκους ε, για τις εκθέσεις που κατατέθηκαν για το μέλλον της περιφερειακής πολιτικής και εκφράζονται σκέψεις και προτάσεις. Τις διάβασα προσεκτικά αυτές τις υπηρεσίες και η υπηρεσία μου, οι υπάλληλοι μου διάβασαν και πρόσεξαν ιδιαίτερα αυτά τα θέματα και παρακολουθούμε και παρακολουθούν τις συζητήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο πολύ προσεκτικά. Είναι σημαντικές προτάσεις επί της, των προτάσεων της Επιτροπής και των συζητήσεων που διεξάγονται για την μετεξέλιξη της πολιτικής συνοχής και περιφερειακής πολιτικής και που σίγουρα με αυτόν τον τρόπο υπάρχει μια παράλληλη έκβαση στο work in progress, στο έργο που βρίσκεται υπό εξέλιξη, εμρευστό και μετεξελίσσεται. Την επόμενη εβδομάδα, όπως είναι γνωστό, σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχουμε τις ε, δημοσιονομικές προοπτικές ε, στο πολιετές τους πλαίσιο που θα κατατεθούν ως προτάσεις. Και μετά στις 29-30 Ιουνίου, στη συνέχεια αναμένουμε ότι σε σχέση με τα μακροοικονομικά θέματα και την κατάσταση στα κράτη-μέλη, μια και έχουμε δύσκολες διαπραγματεύσεις ε, για τα δημοσιονομικά θέματα που θα εκκρεμούν κατά τους επόμενους μήνες και ελπίζω όχι και χρόνια βέβαια, αλλά απλώς μήνες, και βασίζομαι πρέπει να πω στεναρά στην υποστήριξη του Ευρωκοινοβουλίου και αντίστροφα εσείς μπορείτε να βασιστείτε σε εμά. και βασίζομαι και στην υποστήριξη των περιφερειών. Ένα πράγμα πρέπει όμως να είναι σαφές. Αν θέλουμε να υλοποιήσουμε μια περιφερειακή πολιτική, αυθεντική πολιτική, που θα ανταποκρίνεται στις υψηλές προδιαγραφές και προσδοκίες όπως εκφράζονται και στις διαφορετικές εκθέσεις, τότε χρειαζόμαστε κάπως ε, επαρκή προϋπολογισμό και επαρκή κονδύλια για να τα κάνουμε όλα αυτά. Νωρίς το φθινόπωρο, και λέω κατά τα τέλη Σεπτεμβρίου περίπου, ανάλογα σε σχέση με το σχέδιο προϋπολογισμού που θα έχουμε, θα υποβάλουμε τις προτάσεις μας όσον αφορά τις διαφορετικές δράσεις και διατάξεις και κανονισμούς για την, για την πολιτική συνοχή ε, από το 2014. Ως Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλουμε ένα πακέτο μέτρων όσο αφορά κανονισμούς και διατάξεις που πιθανότατα τα εξή στοιχεία θα συμπεριλαμβάνει αυτό το πακέτο. Ένα γενικό κανονισμό πρώτα. Ένα κανονισμό στην συνέχεια για το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο. Κανονισμό για το Ταμείο Συνοχής ένα κανονισμό, ένα κανονιστικό πλαίσιο για το κοινωνικό ταμείο και τέλος κανονισμό για την περιφερειακή συνεργασία. Ελπίζουμε με όλα αυτά ότι με τη βοήθειά σας οι διαπραγματεύσεις θα μπορέσουν μέχρι τα τέλη 2012 ή κατά τις αρχές του 2013 να ολοκληρωθούν. Αυτό και στις εκθέσεις έτσι εκφράστηκε. Το ότι δηλαδή θα έπρεπε εμείς, ας το πω έτσι, από την τρέχουσα περίοδο να μπορέσουμε τα συμπεράσματά μας να τα συνάξουμε, να μπορέσουμε να τα διατυπώσουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε οι καθυστερήσει στην υλοποίηση του έργου όσον αφορά και τις διάφορες αυτές διαδικασίες να μην υπερβολικά καθυστερήσουν. Αυτό θα είναι όμως δυνατόν αν έγκαιρα και πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014 τα καταφέρουμε. Δηλαδή το δυνατόν νωρίτερα το 2013 να έχουμε ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες και διεργασίες ώστε με τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες τα διάφορα αυτά θέματα των εξελίξεων για τα θέματα επενδύσεων και λειτουργικών προγραμμάτων να συμφωνήσουμε αυτό το πλαίσιο οι διαπραγματεύσεις άτυπα ξεκινούν νωρίτερα κιόλα, αλλά επίσημα μπορούν να ολοκληρωθούν φυσικά μόνο όταν θα έχουμε ως βάση ένα πλήρες πλαίσιο. Δηλαδή, μια πλήρη απόφαση και που θα βασίζεται σε γνώσεις για τα νομοθετικά πλαίσια, τις νομοθετικές προϋποθέσεις και τους όρους που, στους οποίους θα κινηθούμε. Είναι σημαντικό όμως πριν από την έναρξη της νέας περίοδου να έχουμε επαρκή χρόνο για την υλοποίηση όλων αυτών, για την εφαρμογή τους. Είναι προς το συμφέρον μας με την 1η Ιανουαρίου 2014 να τα καταφέρουμε χωρίς καθυστερήσεις αν γίνεται, αμέσως να περάσουμε χωρίς καμία διακοπή στη νέα περίοδο και έτσι στις πολίτες, στους πολίτες μας και στις περιφέρειες αυτό να είναι υποφελές. Πέρα από αυτό εργαζόμαστε, συνεργαζόμαστε και με τους συναδέλφους και των άλλων υπηρεσιών ώστε από κοινού να εκπονήσουμε ένα στρατηγικό πλαίσιο που όλα τα διαρθωτικά θέματα που μέχρι τέλη του έτους θέλουμε να έχουμε ρυθμίσει θα τα λαμβάνουν υπόψη Πιστεύω και το λέω αυτό ειλικρινά και ανοιχτά, οι συζητήσεις δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί από πλευράς μας. Όμως πιστεύω παρόλα αυτά ότι αυτή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους συνομοθέτες θα πρέπει να υποβληθεί, να κατατεθεί για να ληφθεί απόφαση από αυτούς. Και νομίζω ότι δεδομένων των του ευρύτερου πλαισίου αυτού του στρατηγικού ε, πλαισίου, αυτού του στρατηγικής αυτής της στρατηγικής προσέγγισης είναι σκόπιμο και καλό οι συνομοθέτες να έχουν στη διάθεσή τους <clears throat> την δυνατότητα να εμπλακούν και να συνεξετάσουν όλα αυτά. Το κύριο μέλημα, το κύριο θέμα είναι να υλοποιηθούν οι στόχοι της στρατηγικής του 2020 για την Ευρωπαϊκή Ένωση με συγκεκριμένες προτεραιότητες ε, στις επενδύσεις και έτσι νομίζω ότι θα πρέπει με σαφήνεια να υπάρξει ε, τοποθέτηση και συντονισμός μεταξύ μας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μένα να επισημάνω ότι με την συνάδελφο Κουίν εργαζόμαστε ώστε να υπάρξει η καλύτερη συνεκτικότητα και συνάφεια μεταξύ του πλαισίου για τα διαθροτικά κονδύλια και του στρατηγικού πλαισίου, ιδιαίτερα για καινοτομία. Να διασφαλίσουμε αυτή την ε, εφαρμογή. Η έννοια αυτή να εξεταστεί σε ευρύ πλαίσιο ώστε να μπορέσει από την έρευνα, και στην περιφερειακή πολιτική να λειτουργήσει και να είναι αποτελεσματική σε σχέση με την εκμετάλλευση ιδιαίτερα ε, των δυνατοτήτων που θα προσφέρονται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ένα άλλο ξεχωριστό σημείο συζήτησης εδώ στο Κοινοβούλιο και όπου υπήρξαν και διαφορετικές απόψεις μεταξύ των ευρωβουλευτών που εκπροσωπούνται στο σώμα σας και ημών και κυρίως εμού προσωπικά, όμως παρόλα αυτά δεν είναι τίποτα τραγικό αυτή η διαφορά απόψεων, γιατί είναι μια συζήτηση αντικειμενική αυτή που διεξάγουμε. Και το θέμα του αν η πρόταση αυτή για την εισαγωγή μιας ενδιάμεσης κατηγορίας για περιφέρειες δηλαδή για περιφέρειες μεταξύ 75 και 90% transition regions, δηλαδή προσωρινή μεταβατική κατηγορία προσωρινών ε, μεταβατικών ε, περιφερειών. Νομίζω ο συμβιβασμός που βρέθηκε και βρίσκεται υπό εξέλιξη είναι σκόπιμος και καλός και μπορεί να ανταποκρίνεται στις, ε, στον προβληματισμό μας. Και πάλι, για όλα όσα βρίσκονται πίσω από αυτές τις σκέψεις, εμείς στην Ευρώπη αυτό που έχουμε είναι, νομίζω συνολικά, μέσα στο πλαίσιο των περιφερειών μας, έχουμε ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό μια θετική εξέλιξη. Αν δούμε τουλάχιστον το ΑΕΠ και χρησιμοποιήσουμε το ΑΕΠ ως πύχη, ως γνώμονα. Παρόλα αυτά όμως από την άλλη πλευρά υπάρχουν ακόμα επαρκώς πολλές αρκετές περιφερειές που πρέπει να καλύψουν την απόσταση που τις χωρίζει για να φτάσουν στις ευρωπαϊκές μέσες, στους ε, ευρωπαϊκούς μέσους όρους ε, ως ε, στοιχείο. Και μέχρι σήμερα είχαμε μια κατηγοριοποίηση ανάλογα με το, το κατόφλι του 75%, δηλαδή περιφέρειες κάτω από αυτό το ποσοστό έχουν λιγότερο καλά αναπτυχθεί όσον αφορά τη συνεκτικότητα και γι' αυτό αυτό στην χρηματοδότηση, στην κατανομή, στον επιμερισμό κονδυλίων είναι εύκολο να παρατηρηθεί γιατί έχουμε την αναλογία καταρχήν 1 προς 10. Αυτό και στο μέλλον έτσι θα συμβαίνει και νομίζω ότι μια και εμείς ήδη σήμερα έχουμε ένα phasing out ή και ένα phasing in θα μπορούσαμε να πούμε και για λόγους ε, μη υπερβολικής περιπλοκής ε, των θεμάτων δεν θα αναφερθώ σε αυτές τις λεπτομέρειες. Δημιουργούμε μια δυνατότητα μετάβασης από την ε, συνοχή και σύγκληση στην ανταγωνιστικότητα περιφερειών προς όφελος ενός soft landing, μιας ήπιας προσγείωσης, να διοργανώσουμε χωρίς προβλήματα μια τέτοια μετάβαση. Δεν αντιμετωπίζει αντιρρήσεις κάτι τέτοιο. Αν από αυτή την κατηγορία 75% κάποιος βγει από αυτήν, δεν έχει φτάσει ακόμα στον στόχο, έτσι δεν είναι. Δεν έχει υλοποιήσει τον στόχο να υλοποιείται απόλυτα ο μέσος όρος της Ευρώπης και γι' αυτό πρέπει να συνεχιστούν οι διαδικασίες υποστήριξης και πρέπει να υπάρξει μια συνέχεια και διασφάλιση όλων αυτών των ε, δράσεων στήριξης. Και υπάρχουν μετά και άλλες περιφέρειες που ποτέ δεν βρέθηκαν κάτω από το 75% ως μέσο όρο, αλλά δεν βρέθηκαν και ποτέ πάνω από το 90% και που ουσιαστικά από την, ε, ας το πω έτσι, οικονομική τους επίδοση, από το επίπεδο ευημερία των ατόμων που ζουν σε αυτές, ουσιαστικά με ίδιο τρόπο πρέπει να αντιμετωπίζονται, όπως εκείνες οι περιφέρειες που ουσιαστικά έχουν τη διαδικασία κάλυψης της απόστασης που πρέπει να καλύψουν. Μόνο που αυτή η κάλυψη της απόστασης ε, δεν είναι εξίσου ταχεία, διότι έχουμε και μία κάλυψη απόστασης όταν έχουμε και περιφέρειες του 60% που φτάνουν στο 70% ή στο 75% και που τα περαιτέρω βήματα από τα 85% στα 90% απομένουν κτλ. Όλα αυτά όμως πρέπει να υποστηρίζονται και να συνεχίζονται υποστηρικτικά ως μέτρα αρρωγής. Και έτσι για την μη διαφοροποίηση μιας περιοχής που βρίσκεται στο 82 περίπου της 100 και για να πω ένα ακραίο παράδειγμα στο, ε, στο Inner City of London στην ε, στο, στο κέντρο του Λονδίνου που βρίσκονται στο 380% και γι' αυτό πρέπει να βοηθήσουμε κάποιες περιφέρειες. Αυτές οι περιφέρειες που χρειάζονται να καλύψουν κάποια απόφαση να μπορούν να συμμετέχουν. Και αυτό γιατί, διότι εμείς στην περιφερική πολιτική έχουμε δύο κύριους στόχους που θέλουμε να υλοποιήσουμε. Και το λέω ειλικρινά αυτό. Ιδιαίτερα ο δεύτερος στόχος βρίσκεται εκτός αυτού του πλαισίου και δεν έχει υλοποιηθεί πλήρως. Ο πρώτος στόχος, οι παραδοσιακές αντιθέσεις και διαφορές που υπάρχουν μεταξύ περιφερειών να καλυφθούν και να βρούμε τρόπους για τις μεταβατικές περιφέρειες, ενδιάμεσες περιφέρειες να υποστηριχθούν όπως πρέπει. Δεύτερος στόχος, είναι εκείνο το μέσο, το εργαλείο, το tool στην Ευρώπη να βρούμε και να χρησιμοποιήσουμε ώστε τα ευρωπαϊκά προγράμματα με στοχοθέτηση αυτά τα οποία βρίσκονται στη στρατηγική της Ευρώπης 2020 να μεταφραστούν με συγκεκριμένες χειροπιαστές δράσεις. Και αυτό είναι έργο της περιφερειακής πολιτικής. Συνολικά, πανευρωπαϊκά να δράσουμε, ώστε να υπάρξουν αυτές οι προϋποθέσεις το τμήμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να αυξηθεί. Μέτρα αποδοτικότητας της ενέργειας να υποστηριχθούν, να είμαστε πιο αποδοτικοί στην εκμετάλλευση, στην χρήση ενέργειας και εδώ τα ουσιοδέστερα θεμελιώδη στοιχεία ακριβώς για αυτές τις μετανατικές περιφέρειες. Αν τα δούμε τότε σκόπιμο θα ήταν και σε αυτό το πεδίο να δράσουμε ώστε να υποστηρίξουμε, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε γιατί έχουμε περιφέρειες ανταγωνιστικότητας οι οποίες δεν παραμένουν, δεν λιμνάζουν σε κάποιο επίπεδο, μετεξελίσσονται και γι' αυτό σκόπιμο είναι και δίκαιο αυτές τις διαδικασίες να τις υποστηρίξουμε, να βοηθηθούν αυτές οι περιφέρειες. Όλους εκείνους που, θε, που θεωρούν ότι όλα αυτά συνεπάγονται πρόσθετα κόστη και δαπάνες, θέλω να πω ότι πρέπει να διαφοροποιήσουμε μεταξύ κονδυλίων δημοσιονομικά του προϋπολογισμού και πολιτικών ενιών και προσεγγίσεων ή στοχοθετήσεων. Μέσα σε αυτό το πολιτικό πλαίσιο εμείς εκπροσωπούμε την άποψη, εγώ εκπροσωπώ την άποψη, πρέπει να έχουμε αυτή την αρχιτεκτονική δομή και με μια μετάθεση των κονδυλίων να μεριμνήσουμε ώστε η χρηματοδότηση αυτών των ενδιάμεσων μεταβατικών περιφερειών να μπορεί να διασφαλιστεί η χρηματοοικονομική υποστήριξή τους ανεξάρτητα από το τι γίνεται σε σχέση με απόλυτα μεγέθη στον προϋπολογισμό στο σύνολό του, μέσα σε αυτή τη στοχοθέτηση τα κονδύλια για αυτή τη μεταβατική, τις μεταβατικές ή προσωρινές περιφέρειες ή ενδιάμεσης κατηγορίας περιφέρειες πρέπει να διασφαλιστούν και για τους βουλευτές ε, περιφερειών και χωρών που αφορώνται από αυτό Κάθε χώρα θα έπαιρνε περισσότερα κονδύλια. Αν υπήρχαν μεταβατικές τέτοιες περιφέρειες από αυτή τη χώρα, σε σχέση με το αν δεν υπήρχαν. Αυτό φυσικά εξαρτάται από την γραμμή κίνησης των κονδυλίων του προπολογισμού. Αλλά όταν υπάρχουν τέτοιες ενδιάμεση κατηγορία περιφέρειες, οι χώρε του παίρνουν περισσότερα κονδύλια για αυτέ. Και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαφοροποιούμε μεταξύ δημοσιονομικών αρχών ή αρχών που αφορούν τα κονδύλια του προπολογισμού και τη πολιτική προσέγγιση και στοχοθέτηση. Θέλουμε να υπάρξει μια αντιστάθμιση συμφερόντων, μια σωστή εξισορρόπηση εξισορρόπηση συμφερόντων για τις περιφέρειες. Και να μην αμελούμε, να μην ξεχνάμε ότι αυτό αφορά 30 εκατομμύρια πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξαρτώνται από αυτή την χρηματοδότηση και θα υποφεληθούν από αυτήν. Λοιπόν, τούτων λεχθέντων σίγουρα θα έχουμε όλες τις δυνατότητες να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Είμαι πάντα στη διάθεσή σας και όπως είπα θα ήθελα ολοκληρώνοντας παράλληλα με τον Μάρκους Πίπερ και τον συνάδελφο Σταυρακάκη να ευχαριστήσω, Βλάσακ, Νικολάτσικ και Σάντσες, να ευχαριστήσω για τις τελευταίες εκθέσεις των τελευταίων εβδομάδων και μηνών, για τις σκέψεις και προτάσεις που βρήκανε μεγάλη αποδοχή και έγκριση και που βοηθούν την ε, μετεξέλιξη της δικής μας προσέγγισης και αντιμετώπισης. Χαίρομαι ιδιαίτερα και προσβλέπω στη συζήτηση που θα διεξαχθεί εδώ σήμερα και μεθαύριο στην Ολομέλη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιωχάνες Χάν. Κύριε Επίτροπε, μια ολόκληρη σειρά θεμάτων ε, παρεμβάσεων έχουμε. Πρώτα απ' όλα οι συντονιστές έχουν ζητήσει να παρέμουν. Έκανες λόγο για το ότι πρέπει, ε, ότι ε, βρήκαμε ένα σωστό συμβιβασμό. Η ψηφοφορία την Πέμπτη στην Ολομέλεια αναμένεται να γίνει και πραγματικά αναμένω και προσβλέπω να δω ποιοι συμβιβασμοί τελικά θα είναι εκείνοι που θα κυρωθούν και θα εγκριθούν. Έχουμε έχω το ε, καθήκον να, είμαι, να προεδρεύω στη συνεδρίαση και πρέπει να είμαι συνετός. Τον λόγο έχει ο συντονιστής μας από το ΕΛΚ και μετά η κυρία Κωνσταντσε Κρέλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, να μείνουμε στα βασικά. Οι κανονισμοί αυτοί, όπως έχουν συζητηθεί και προηγουμένως, ε, δεν τα καλύπτουν όλα τα ζητήματα. Επίσης, ε, προτείνω να ε, συμπεριλάβετε αυτή την προσδοκία ότι θα χειριστούμε και το στρατηγικό πλαίσιο για τη δικασία της απόφαση. Αυτό μας χαροποιεί και η πρόεδρο μας, κυρία Χίμπνερ, σα έχει ε, γράψει μια επιστολή από αυτού. Θα ήταν καλό την πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε με τα υπόλοιπα ταμεία να καταλήξουμε σε ένα πλαίσιο το οποίο θα ελαμβάνει υπόψη και τα προγράμματα που συμπεριλαμβάνονται στρατηγική για το 2020. Και θα ήθελα να δώσω έμφαση σε αυτό το σημείο, γιατί για παράδειγμα, τώρα βλέπουμε ότι ε, αν εξετάσουμε τα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης, ε, δεν συμβαίνει αυτό. Ε, ήδη εδώ και μερικά χρόνια ε, προσπαθούμε να επιτύχουμε τους στόχους του 2020 και αυτό δεν αφορά μόνο τον τρόπο με τον οποίο ε, καθορίζουμε ε, ε, τις δαπάνες μας, αλλά και με τα συνεργασία μεταξύ των περιφερειών για την συνεχτικότητα και την αποτελεσματικότητά μας. Έτσι πρέπει τη δράση μας να διευρύνουμε και σε άλλους τομείς. Γι' αυτό και εμείς μιλήσαμε για καλές συμφωνίες εταιρικής σχέσης, partnership contracts, και αυτό θα πρέπει να το κάνουμε και στο επόμενο διάστημα. Πολύ καλά λοιπόν, αν είναι έτσι αυτοί οι κανονισμοί θα συμφωνήσουμε. Τώρα, για την συζήτηση ε, προτεραιοτήτων ε, αυτή τη, αυτή τη βδομάδα στο Κοινοβούλιο, πολύ θετικό βήμα και αυτό. Μπορούμε δηλαδή από πλευρά Κοινοβουλίου να θέσουμε τις απόψεις μας και πρέπει να πω ότι τα βλέπουμε όλα με καλό μάτι όλα αυτά τα ζητήματα. Τώρα, υπάρχουν συστήματα για τα οποία δεν έχουμε αρκετές πληροφορίες, παίρνουμε πληροφορίες δεξιά και αριστερά, αλλά δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση της Επιτροπής. Δεν έχουμε τίποτα χειροπιαστό. Και το τελευταίο διάστημα είχαμε μια συζήτηση που ξεκίνησε και από την Επιτροπή ΣΥΡ, αλλά εμείς θα προτιμούσαμε, αν ε, συζητάμε μια μορφή μετάβασης, ε, είτε τη λέμε κατηγορία, δεν ξέρω πώς ακριβώς θα το ονομάσουμε αυτό, να ξεκινάμε από μια ξεκάθαρη πρόταση. Πολύ, πολύ ξεκάθαρα τα σήμερα ο Επίτροπος, αλλά δεν το έχω δει αυτό επί χάρτου. Και αυτό μας δυσκολεύει στο να καταλήξουμε σε μια συγκεκριμένη πολιτική ή σε ένα συμβιβασμό, γιατί ο συμβιβασμός Ε, θα πρέπει να διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχουν ε, δεσμενείς επιπτώσεις. Σε αρκετά κράτη-μέλη δεν έχει ξεκινήσει καν ο στόχος 2. Και όταν ε, πάμε να εισαγάγουμε ε, μεταβατικές κατηγορίες, αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα. Βεβαίως και υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ των κρατομελών. βέβαια όχι πάντα όσο θα έπρεπε και αυτό με λυπεί, αλλά ε, λόγω αυτού του γεγονότος μπορούν ορισμένα κράτη μέλη να χάσουν τον στόχο 2. Επομένω, δεν θα πρέπει αυτοί οι μεταβατικές, αυτές οι μεταβατικές κατηγορίες να έρθουν και να λειτουργήσουν σε βάρος ε, των στόχων 1, 2 και 3. δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο που να έχουμε καταλήξει ακριβώ ε, στην κατάλληλη διαδικασία. Θα πρέπει λοιπόν να τα συζητήσουμε περαιτέρω. Πιστεύω ότι βραχυπρόθεσμα μόλις έχουμε την, απόφαση, την πρόφαση Λεβεντόσκη ε, για τα δημοσιονομικά ζητήματα θα πρέπει να, να δώσουμε έμφαση σε αυτό το τομείο γιατί σε ένα ορισμένο πλαίσιο υπάρχει αρκετό ε, πεδίο δράση για τον στόχο 2 και για κάποια ζητήματα τα οποία αποτελούν προτεραιότητε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίω υπάρχει και η συνοχή με τι μεταφορέ ή με άλλε εμβληματικέ πρωτοβουλίε ε, τη στρατηγική 2020. Με επενδύσει. Ε, Πώ θα εξετάζει αυτό το ζήτημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήταν καλό αυτό να γίνει πριν τι καλοκαιρινέ δικοπέ, αλλά αν αυτό δεν είναι δυνατόν, έστω και μετά. Τι συμβαίνει με, αυτό το, σε αυτό το πλαίσιο το δημοσιονομικό. Ε, για την συνεχιζόμενη ε, αξιολόγηση της ε, ε, πολιτικής ε, καλής γειτονίας. Εκεί βλέπουμε ότι θέλουμε να στηρίξουμε περισσότερο την, ε, τον εκδημοκρατισμό ή τις, αυτές τις ε, δυνάμεις ε, στην Βόρεια Αφρική, στην Ρωσία που θέλουν να βελτιώσουν το επίπεδο της δημοκρατίας. Όμως υπάρχουν κονδύλια τα οποία έχουμε παρκάρει εντός εισαγωγικών σε αυτήν την πολιτική γειτονία αλλά αυτό δεν είχε καλά αποτελέσματα και βλέπουμε ότι αυτό συνεχίζεται. και δεν εστιάζουμε σε άλλους τομείς που θα έπρεπε να δώσουμε την προσοχή μας. Θα πρέπει λοιπόν να παρουσιάσουμε μια καλύτερη αξιολόγηση για να δούμε αν γίνεται σωστή κατανομή των κονδυλίων ε, στο Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και αν θα πρέπει να διατηρήσουμε αυτή την, αυτή την κατανομή μας ε, στα εξωτερικά σύνορα. Εδώ πρόκειται για ουσιαστικά και θεμελιώδη ζητήματα. Και ήθελα να αναφερθώ σε αυτό, αλλά θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Κωνσταντσε Κρέλ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Μάρκους. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Επίτροπε. Οι τις δύο πιο σημαντικές υποθέσεις διεξοδικά τις καλύψατε. Ποια σχέδια κανονισμών υπάρχουν και πώς εσείς πρώτον στην Περιφερειακή Επιτροπή και στην έκθεση Γαρίγα στην Ολομία, Ολομέλεια πώς σε σχέση με τις ε, πλειοψηφίες ε, για ε, την ενδιάμεση κατηγορία μετεξελίσσεται το θέμα. Ελπίζουμε ότι την Πέμπτη θα έχουμε μια τρίτη φορά ή δεύτερη φορά επιβεβαίωση στην Ολομέλεια αυτών όλων, διότι την ενδιάμεση κατηγορία την θεωρώ πολύ σημαντική για μια ολόκληρη σειρά περιφερειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν πάση περιπτώσει θα ήθελα όμως αν γίνεται δύο άλλες πτυχές εδώ να αναφέρω και να καλύψω. Πρώτον, θα με ενδιαφέρε να ακούσω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα από πλευρά τη. Αν στο σχέδιο προπολογισμού το οποίο καταθέτει και που προτείνει, προβλέπεται ένα ταμείο επενδύσεων που θα δημιουργηθεί εκ νέου ή αν αυτή η πρότασή σας ε, έχει τεθεί στο αρχείο και δεν έχει επικαιροποιηθεί σε σχέση με την πολιτική συνοχή. Τι πρόκειται να γίνει. Δεύτερον, Διεξοδικότερα τοποθετηθήκατε για τη συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση για την Έρευνα. Δεν είπατε όμως κατά πόσον η συνεργασία και ο συντονισμός προχωρεί σε σχέση με το Ταμείο για τη Γεωργία και πόσο, κατά πόσον αυτό ε, διευκολύνθηκε και με το Ταμείο για την Αλληλεία και αν θα υπάρχει η δυνατότητα μέσα σε αυτό το κανονισμό να υπάρχει ισχυρότερη διασύνδεση αυτών των δύο τομέων, Γεωργίας και Αλίας, όσον αφορά τη συνοχή τις προσπάθειες για τη συνοχή. Υποθέτω ότι ένα τέτοιο θέμα φυσικά έχει κάποια επιρροή στα θέματα του προϋπολογισμού. Ακούω ότι ο δεύτερος πυλώνας για την γεωργική πολιτική έχει, πρόκειται να ελαχιστοποιηθεί λέει. Και αυτό το οποίο ήθελα να συνδέσουν με την αγροτική, με τη γεωργική πολιτική δημιουργεί κάποιες δυσκολίες. Έχω ανάγκη να μου απαντήσετε αυτό το ερώτημα. Μία παρόδο παρατήρηση Πρόσφατα είπα σε μια αποστολή με, στην, στο Ηνωμένο Βασίλειο και με τη συζήτηση που είχαμε με την Βαρόνι Χέμσερ που είναι αρμόδια από τη Βρετανική κυβέρνηση για το Περιφερειακό Ταμείο επεσήμανε επανειλημμένα ότι είπε ο Treasurer, ο Υπουργός Οικονομικών, ότι πρέπει το, ο υπολογισμός να περικοπεί και δεν υπάρχουν δυνατότητες περαιτέρω κατανομής κονδυλίων. Και στη δεύτερη παρέμβασή της αναφέρθηκε γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να διασφαλίζει στο μέλλον αυτές τις δύο πηγές χρηματοδότησης. Ίσως όλα αυτά θα πρέπει να τα συνεξετάσουμε, ίσως είναι θελκτικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και για τους φιλελεύθερους. Ο Μιχαήλ παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε πίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Στις εκθέσεις αυτές μια ολόκληρη σειρά θεμάτων εμπεριέχονται και αιτήματα που είναι σημαντικά για τους φιλελεύθερους. Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ κυρίως στο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά την υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και σε διασύνδεση με την μετάθεση, μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και συνεργασία με τα πανεπιστήμια βρήκαμε μία διατύπωση ότι το Ταμείο Συνοχής και από πλευρά των κονδυλίων των διαθωτικών πρέπει να διευκολυνθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης ώστε να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο και στο μέλλον η δυνατότητα για την απασχόληση. Είναι σημαντικό να υπάρχει και συνένεση από τις κοινοβουλευτικές ομάδες που με μεγάλη πλειοψηφία υποστηρίζουν αυτές τις προτάσεις. Στη σημερινή συζήτηση, όπως ο συνάδελφος Λάμπερτ Φανίστερ Ρόι προανέφερε, το θέμα της ενδιάμεσης κατηγορίας διαδραματίζει ένα ρόλο. Έστω και θεωρητικά, έστω και καθαρά θεωρητικά, στις συστηματικές συζητήσεις αυτή η πρόταση ήταν πολύ θελκτική, ας το πω έτσι, με το επιχείρημα ότι όχι μόνο εκείνοι που βρίσκονται στη φάση phasing out, που ουσιαστικά τώρα από ένα χαμηλότερο ποσοστό έφτασαν σε ένα υψηλότερο ποσοστό του ΑΕΠ, να μπορούν όχι μόνο εκείνες οι περιφέρειες να απολάβουν αυτών των κονδυλίων αλλά και οι περιφέρειες που μέσω κάποιων πληγμάτων που ε, επλήγησαν από αυτά και βρέθηκαν από υψηλότερη κατηγορία σε χαμηλότερη κατηγορία και αυτές να απολάβουν από αυτή την υποστήριξη ώστε να μπορούν να στηριχθούν από τα ε, κονδύλια αυτά υποστήριξη με σταθεροποιητικές δράσεις ε, υπό αυτό το πρίσμα μακροοικονομικά να δούμε την ενδιάμεση κατηγορία που έχει κάποιο νόημα να υπάρχει. Και για τη δική μας ομάδα διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο αυτό το επιχείρημα. Και από αυτό θα εξαρτηθεί η στάση μας στην ψηφοφορία. Πόσες περιφέρειες σε αριθμό συμπεριλαμβάνονται. Τι θα κοστίζει αυτό συγκεκριμένα ως δαπάνες και συμφωνώ με τον κύριο Φανίστερ Ρόι, θα ήταν επικοδομητικό αν είχαμε γραπτά στοιχεία, υπολογισμούς που να αποσαφηνίζουν τι γίνεται με όλα αυτά, με τις δαπάνες και τη στήριξη. Γι' αυτό συγκεκριμένη ερώτηση επίτροπε προς εμάς. Από τις 40 περιφέρειες, αληθεύει ότι περίπου 40 περιφέρειες είναι που καλύπτονται. 9 δις λέει ευρώ πρόσθετα θα απαιτηθούν όμως αυτά δεν μπόρεσα να τα επαληθεύσω εγώ ως αριθμητικά μεγέθη. Μπορείτε να μας πείτε κάτι για τα πρόσθετα κόστη που αναμένονται και πόσο μεγάλος είναι ο αριθμός των περιφερειών όσον αφορά το σημερινό τους επίπεδο σήμερα που στην παλαιά κατηγορία στόχου 1 ε, παρέμεναν. Και τώρα θα ήθελα να αναφέρω ένα άλλο σημείο πιο σύντομα. Γνωρίζετε ότι ως εισηγητής για το ποσοστό απορρόφησης, την απορροφητικότητα, εξετάζω κάποια θέματα και είχαμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Και εδώ δείχνει ο αριθμός ε, της απορροφητικότητας, ε, τα ποσοστά απορροφητικότητας ότι κάποιες περιφέρειες έχουν καλές επιδόσεις έχουμε την εντύπωση ότι κάποιες περιφέρειες και χώρες επιταχύνουν τους ρυθμούς τους. Υπάρχουν άλλες περιφέρειες και χώρες που έχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες. Ήταν δύσκολο να βρούμε ποιο είναι το ποσοστό απορροφητικότητας πραγματικά για κάποιες χώρες. Και η συνάδελφος Γκρέσλε από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού μας ανέφερε μια συζήτηση στη Νότια Ιταλία που είχε. Εκεί οι ελεγκτές, δημοσιονομικοί ελεγκτές την ενημέρωσαν την κυρία Γκρέσλε ότι η απορροφητικότητα βρισκόταν λέει κάτω από 7%. Τέτοιου είδους φήμες ή στοιχεία μπορείτε να τα υπαλληθεύσετε, γνωρίζετε αυτά τα αριθμητικά μεγέθη, αυτά τα στοιχεία. Και εμείς ως κοινοβούλιο δεν θα έπρεπε άμεσα για να ενημερωνόμαστε για την απορροφητικότητα, ώστε από πολιτική πλευράς να μπορούμε άμεσα τις δυσκολίες που υπάρχουν προφανώς εν μέρη για την υλοποίηση αυτών των προσπαθειών να τις παρακολουθούμε και να μπορούμε να δράσουμε στηρικτικά. Ευχαριστώ. Ja, ich würde jetzt ganz gerne dem... Θα ήθελα τώρα, αν γίνεται, να δώσω τον λόγο στον Επίτροπο τώρα. Η... Για λόγους ε, και τάξης ε, το θέμα της ενδιάμεσης κατηγορίας και της χρηματοδότησης των περιφερειών είχε κύριο ρόλο. Αλλά καταρχήν τώρα λοιπόν πρώτα ο Επίτροπος για αυτή τη θεματική ενότητα. Επίτροπος, σας ευχαριστώ. Με τη σειρά των παρεμβάσεων που έγιναν να απαντήσω αν γίνεται. Πρώτα, παρακαλώ να δείξετε κατανόηση για το γεγονός ότι όταν έχουμε ένα σχέδιο το οποίο θα καταθέσουμε το Σεπτέμβριο δεν μπορούμε να έχουμε και προσχέδιο. Αυτό είναι αν θέλετε, χαρακτηριστικό των σχεδίων που κατατίθενται. Κάποτε ένα πρώτο έγγραφο υποβάλλεται, κατατίθεται και μετά μπορούν κάποια πράγματα να συζητηθούν αφού έχει κατατεθεί. Αλλά η δυνατότητα είναι δεδομένη με προφορική επαφή και συζήτηση να μπορούμε να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων και μπορείτε να βασιστείτε στο ότι τα πράγματα τα οποία σας αναφέρω εγώ δεν αποσυνδέονται από το αντικείμενο προβληματισμού μας και στη συνέχεια και στο σχέδιο το οποίο θα καταθέσουμε θα ξαναβρεθούν, θα αντακλώνται σε αυτό. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι πρώτα απ' όλα καταβάλουμε και θα καταβάλουμε αυτή την προσπάθεια μέσα στο πλαίσιο αυτής της, ε, αυτού του κοινού στρατηγικού πλαισίου με τα άλλα ταμεία για την αλληλεία και τη γεωργία φυσικά. Να υπάρξει ένας συντονισμός που θα διασφαλιστεί, ώστε ακριβώς όσον αφορά τις πιο σημαντικές, τις πιο σοβαρές επενδύσεις και σχέδια, προγράμματα επενδύσεων που έχουμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο, να δούμε πώς μεταξύ των διαφορετικών ταμείων θα επιμεριστεί το έργο. Ιδιαίτερα αφορά αυτό όσον αφορά τους πολιτικούς τομείς επενδύσεων που πρέπει να κλείσουν, να συμφωνήσουμε επ' αυτού του πλαισίου και με αυτή την απόφαση να κατανείμουμε τα βάρη, να δούμε ποιος θα μεριμνήσει για ποια δράση ως κέντρο βάρους και σε σχέση με την, ε, ε, με το, και με τις περιφερειακές δράσεις. Γι' αυτό από πλευράς του Επιτρόπου Σόλος υπευλήθη αυτή η πρόταση και έτυχε άμεσα συνέχεια από εμάς. Η υπεύθυνη για τη γεωργία δεν θα μας εξέπλητε να μην ε, ε, έχουν κάποια αντίδραση. Δεν έχω κάποια επισήμαση τι γίνεται σε σχέση με την ανάπτυξη της ε, υπαίθρου, αν θα υπάρξει κάποια συμπίεση ή όχι. Το αντίθετο φαίνεται ότι υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον κιόλα από πλευράς των αρμόδιων για τη γεωργία και από, στις συζητήσεις προσπαθώ να αποσαφηνίσω ότι πρόκειται για το Ταμείο για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου και στην ανάπτυξη της υπαίθρου δεν έχουμε μόνο γεωργικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται, αλλά και άλλες επιχειρήσεις. Και από αυτό το ταμείο καλύπτονται. Και γι' αυτό είναι αναγκαίο αυτό το πλαίσιο να έχει τέτοια μορφή, ώστε η εκμετάλλευση των κονδυλίων να γίνεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πάντα. Τώρα, για το θέμα της governance, της διαχείρισης ε, η διακυβέρνηση. Έχω ήδη αναφέρει ότι από πλευρά του Φαντερ Μπράντε που και σε σχέση με το αξίωμά του ως Προέδρου της Επιτροπής Περιφερειών σε βάθος είχε ασχοληθεί με το θέμα της governance, της διακυβέρνησης και ότι με τη γνωμοδότηση αυτή και την τοποθέτηση αυτή ως σύμβουλος παρακολουθεί market level governance το θέμα αυτό στο σχέδιο κανονισμού Πάντα έλεγα ότι ελπίζω ότι θα μπορέσει να επιβιώσει στις διαπραγματεύσεις αυτή η προσέγγιση και να αντέξει πρώτη παρατήρηση. Δεύτερον, έχει και ένα χαρακτήρα Τοποθέτηση ή δήλωση αυτό αλλά αν βρεθεί και στον κανονισμό και ενταχθεί στον κανονισμό θα έχει πρόσθετη ηθική συνιστόσα ηθική δέσμευση που θα είναι δεδομένη και που θα αναπτύξει τη δραστηριότητά της και την επιρροή της υπάρχουν περιφέρειες και ε, χώρες ε, όπου πρέπει αυτή η αρχή να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη. Σε άλλες περιπτώσεις συμβαίνει ίσως κάτι διαφορετικό. Εδώ πρέπει παντού όπου χρειάζεται να δράσουμε ώστε η κατάσταση να μπορεί να βελτιωθεί. Μπορώ να βεβαιώσω αυτό που είπε η Κωνσταντσε Κρέλ. Θα υπάρξει υποστήριξη για όλες τις περιφέρειες και στην γνωμοδότηση κιόλας ακόμα του Ηνωμένου Βασιλείου αυτό το οποίο αναφέρεται ριτά ότι το δέχονται γίνεται δεκτό επειδή ο χάρτης της Μεγάλης Βρετανίας της επικράτειάς της αναφέρει και δείχνει πώς, πού υπάρχουν αυτές οι περιφέρειες και οι ανάγκες τους και αναγνώρισαν πόσο σκόπιμο και αναγκαίο είναι να υπάρχει αυτή η υποστήριξη. Και με τη στοχοθέτηση της στρατηγικής της Ευρώπης 2020 πρέπει να δράσουμε σε όλες αυτές τις περιφέρειες. Και γι' αυτό για τον Λάμπερτ Φανίστερ Ρόι θα υπάρξει αντίστοιχα μια επαρκής χρηματοδότηση και της ομάδας κατηγορίας 2. Όσον αφορά την πολιτική γεωργίας, όχι μόνο θα συνεχιστεί, αλλά εμπεριέχει και σε σχέση με το στοιχείο των, του πυλώνα όσον αφορά την πυλωνική δομή, ο, τα κονδύλια σε σχέση με την ε, αύξηση που ε, ζητείτε. Γνωρίζετε ότι τα σκανδιναβικά, χώρα, ε, τα σκανδιναβικά κράτη η, την προθυμία για επενδύσεις ε, σε αυτόν τον τομέα την έχουν περιορίσει και επειδή γνωρίζετε ότι έχουν υπάρχουν οι μεγαλύτερες περικοπές, οι πιο ευαίσθητες περικοπές σε αυτούς τους τομείς καμιά φορά ελπίζουμε ότι παρόλα αυτά θα μπορέσει να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια. Όσον αφορά τη συνεργασία με περιφέρειες ή χώρες, πέρα από το να είναι κράτη-μέλη ή την ιδιότητά τους αυτή, υπο... καταρχήν τα προγράμματα θα παραμένουν μέσα στο ίδιο πλαίσιο. Εσωτερικά θα πρέπει να διασφαλίζεται ένας καλύτερος συντονισμός στο μέτρο του εφικτού ώστε να έχουμε μια ενιαία πρόσβαση όσον αφορά τους κανονισμούς στην υποστήριξη. Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως, μέσα στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής, υιοθετείται καμιά φορά ένα διαφορετικό σύστημα από ότι η υποστήριξη εκτός του πλαισίου στήριξης ε, των ε, περιοχών της Ένωσης. Και εδώ έχουμε σπέρματι τα προβλήματα που υπάρχουν και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Όμως μόνο εν μέρη μπορούν να ξεπεραστούν, μόνο μερικά μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Μέσα στην Ένωση πρέπει να έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση με συγκεκριμένη πρικοδότηση, με συγκεκριμένα κονδύλια που θα ε, έχουμε κατανείμει και μέσα σε αυτό το πλαίσιο να προσπαθούμε να δράσουμε. Τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα δεν θα υπάρχει άλλη εναλλακτική δυνατότητα. Ταμείο επενδύσεων Εννοείται το Ταμείο Υποδομών, έτσι υποθέτω. Μάλιστα, Ταμείο για τις Υποδομές. Υποθέτω ότι θα δημιουργηθεί αυτό το Ταμείο Υποδομών, όπου τα κονδύλια που παραδοσιακά από την περιφερειακή πολιτική προήρχοντο να μην θυγούν. Θα πρόκειται όμως για μια βελτιωμένη μορφή συνεργασίας που πρέπει να πετύχουμε, ιδιαίτερα στον τομέα των μεταφορών έχουμε θεμητό αίτημα και έτσι το προσεγγίζουμε ότι τα έργα υποδομών ιδιαίτερα διασυνοριακά και για τα δίκτυα τα διασυνοριακά των μεταφορών είναι ιδιαίτερα αναγκαία και αυτό όχι μόνο στα νέα κράτη-μέλη αλλά και στα παλαιά κράτη-μέλη και γι' αυτό θα πρέπει το Ταμείο Υποδομών να ε, χρησιμοποιείται για, αυτή την, ε, για αυτές τις επενδύσεις και αυτή την δημιουργία αυτής της δικτύωσης θεματολογικά θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο συντονισμού μεταξύ μας ώστε το επόμενο, σημείο, το, ε, επόμενο βήμα που θα ακολουθεί σε σχέση με τα ε, δίκτυα μεταφορών να μπορούν να συντονιστούν οι δράσεις μας πιο αποτελεσματικά. Η πρότασή μας στοχεύει στην κατεύθυνση ότι θα πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο, ένα κατάλογο των αναγκαίων δράσεων διευρωπαϊκών δικτύων διευρωπαϊκών σχεδίων, έναν σαφή κατάλογο ώστε να αποσαφηνίζεται πώς θα χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια και με, ε, προς ποιο στόχο και με ποιο τρόπο θα γίνει ο επιμερισμός. Γιατί επέμεινα στο θέμα της έρευνας. Επέμεινα στην έρευνα επειδή για πρώτη φορά στον τομέα της έρευνας έχουμε την έννοια της καινοτομίας που είναι ιδιαίτερα ανάγλυφος και τονίζεται ιδιαίτερα και είναι σημαντικό να καταστήσουμε σαφές, να αποσαφηνίσουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές έννοιες για την καινοτομία. Δεν είναι μια αντιπαράθεση για το φύλλο των αγγέλων, δεν είναι μια θεωρητική συζήτηση, μια βυζαντινολογία. Είναι χειροπιαστό ζήτημα μέσα στο πλαίσιο της ανάπτυξης του προϋπολογισμού μας. Ε, η μέσα στο πλαίσιο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων η καινοτομία διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν σταματώ να επαναλαμβάνω ότι η καινοτομία δεν είναι μόνο τεχνολογική καινοτομία στο τέλος της αλυσίδας της εξέλιξης των δράσεων, αλλά μπορεί να είναι καινοτομία στο marketing, καινοτομία στην παροχή υπηρεσιών και τα λοιπά και τα λοιπά. Και πρόκειται για μια ευρεία έννοια στην προσέγγιση μας αυτή για τις επενδύσεις, ώστε ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και διασφαλίζουν θέσεις απασχόλησης να μπορέσουν να τονωθούν, να ενδυναμωθούν. Είναι αναγκαίο να εξευρεθεί ο η σωστή οδό συνεργασίας και συντονισμού προς αυτές τις δράσεις μεταξύ μας. Τις επόμενες ερωτήσεις όσον αφορά τις περιφέρειες από πλευράς του Ευρωβουλευτού εδώ θα ήθελα σε σχέση με αυτές τις επιφυλάξεις που υπάρχουν για την μπορεί τα πρόσφατα αυτά στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται για τη μία ή άλλη περιφέρεια, η συνολική όμως εικόνα που έχουμε είναι δεδομένη, είναι σαφής. Αναμένουμε κατά την επόμενη περίοδο 271 περιφέρειες συνολικά που έχουμε σήμερα, από αυτές 51 στην κατηγορία των μεταβατικών ή ενδιάμεσων περιφερειών. Αυτό θα ήταν 72 εκατομμύρια πολίτες ή λίγο παραπάνω από 72 εκατομμύρια. Οι παραδοσιακές phasing out περιφέρειες είναι 17. Οι νέες θα ήταν 34 που θα εντασσόντουσαν. Οι νέες αυτές περιφέρειες προέρχονται από χώρες όπως Βέλγιο, Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Φινλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Γερμανία, Ελλάδα και Αυστρία. 40 εκατομμύρια περίπου πολίτες καλύπτουν αυτές οι περιφέρειες. Τα μεγέθη που αναφέρατε δεν είναι τόσο υψηλά επειδή μέσα σε αυτόν τον αριθμό που εσείς αναφέρατε έχουμε και κόστη που συμπεριλαμβάνονται ήδη που θα έπαιρναν οι περιφέρειες αυτές αν θα ήταν περιφέρειες ανταγωνιστικές, κατηγορίας ανταγωνιστικής. Κάτι λοιπόν πρέπει εδώ να συνυπολογιστεί ώστε με τη μετάθεση που θα έχουμε, θέλω να το τονίσω αυτό, με την μετάθεση υπάρχει ένα μικρότερο από εκείνο το οποίο αναφέρθηκε από εσάς ποσό. Κάνουμε λόγο για 40 εκατομμύρια πολίτες λοιπόν που συνολικά ζουν σε αυτές τις περιφέρειες σήμερα. Έχουμε 271 περιφέρειες. Από αυτές, αυτή τη στιγμή σήμερα, 84 είναι περιοχές, περιφέρειες σύγκλησης. Υπολογίζουμε ότι στην επόμενη περίοδο ο αριθμός ε, της συνοχής των περιφερειών αυτών συνοχής θα είναι μεταξύ 64 και 80 και υπολογίζουμε ότι μέσα στο πλαίσιο των ε, περιφερειών ανταγωνισμού θα έχουμε μικρές αλλαγές, λίγες αλλαγές. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε και μπορούμε να σας δώσουμε αυτή τη στιγμή. Ποσοστό απορρόφησης, απορροφητικότητας. Ναι, έχουμε συνειδητοποιήσει τα προβλήματα που υπάρχουν σε κάποιες χώρες και κάποιες περιφέρειες. Το έχουμε συνειδητοποιήσει απόλυτα και πριν από δύο μήνες όταν ήμουν στην Νότια Ιταλία, κυρία στην Απουλία, στην Καμπανία, και στην Σικελία για να κατασταθεί σαφές για το τι συμβαίνει εκεί διακυβεύεται να χάσουν κονδύλια. Υπάρχει ο κίνδυνος να απολεστούν κονδύλια. Έχουμε commitment rules, έχουμε κανόνες για τη δέσμευση κονδυλίων και φυσικά αυτοί θα πρέπει να τηρούνται και να είναι σεβαστή. Δεν θα υπάρχουν περιθώρια ερμηνεών και διαφορετικών ερμηνεών. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιωθεί η επίδοση αυτών των περιφερειών για να μην απολέσουν κονδύλια. Για άλλους λόγους που μπορείτε να φανταστείτε έχουμε δυσκολίες στην Ελλάδα για παράδειγμα όπου ιδιαίτερα για την ιδιωτική οικονομία σε σχέση με τις δυνατότητες που υπάρχουν και περιορισμένη χρήση κονδυλίων Βουλγαρία, Ρουμανία επίσης έχουμε γνωστά προβλήματα εκεί όπου εδώ Ωστόσο, με όλες τις ε, δυσκολίες που συνδέονται, ε, σκιαγραφούνται κάποιες βελτιώσεις. Ε, έχουμε ίχνη βελτιώσεων. Έχουν κερδίσει έδαφος και μπορούν να βελτιωθούν. Ευελπιστούμε ότι το 2012 θα γίνει πιο αισθητή αυτή η βελτίωση, αυτή η κατάσταση που μπορεί να βελτιωθεί, ιδιαίτερα στη Βουλγαρία για την υλοποίηση κάποιων ε, σχεδίων προγραμμάτων και την καλύτερη απόδοση. Γνωρίζουμε όμως ε, αυτή την κατάσταση και προσφέρουμε σε όλες αυτές τις χώρες την ε, δική μας συνδρομή και υποστήριξη. Υπάρχει ένας προϋπολογισμός με κονδύλια για την τεχνική υποστήριξη, τεχνική αρρωγή δεν γίνεται χρήση όμως πολλές φορές αυτών των δυνατοτήτων. Υπάρχουν όμως αυτές οι δυνατότητες και η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και με την Παγκόσμια Τράπεζα είναι άλλες δυνατότητες αυτές να συνεισφέρουν επαΐοντες πραγματογνώμονες για την κατάρτιση σχεδίων και υλοποίησή τους αλλά δεν μπορούμε εμείς να επιβάλλουμε αυτά τα πράγματα εκ των άνω δια της βίας. Μπορούμε να προσφέρουμε αυτές τις δυνατότητες. Μπορούμε να επεξηγήσουμε ποιες δυνατότητες υπάρχουν, τι μπορεί να γίνει, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Κάποτε πρέπει οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι να πούν, μάλιστα το θέλουμε. Θέλουμε να κάνουμε χρήση αυτών των δυνατοτήτων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για τις απαντήσεις σας. Από τους Πρασίνους, Αλφόνση, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε σε αυτόν τον καθορισμό της μελλοντική πολιτικής της συνοχής νομίζω ότι διαγράφεται μια πλειοψηφία προς ένα πρόγραμμα που γενικά υποστηρίζουμε το σχέδιο, διότι αποκρίνεται σε μια φιλοδοξία να διατηρηθεί μια ισχυρή περιφερειακή πολιτική στην Ευρώπη και να δοθούν και αναγκαίοι πόροι για αυτή την πολιτική. Η αρχιτεκτονική που προτείνεται και σχεγραφείται σήμερα, αυτό το οικοδόμημα, το τετραόροφο κατά κάποιο τρόπο, στόχου 1 παραμένει ο βασικός στόχος, Εν συνεχεία έχουμε τον ενδιάμεσο στόχο. Στόχος 2 παραμένει και στόχος 3 είναι σημαντικός για μας, διότι για μας ε, στο διασυνοριακό σχέδιο ε, ε, χρειάζεται διαχείριση οικονομική και προώθηση ανταγωνιστικότητα που σημαντική για του πληθυσμού. Όλα αυτά που να Αυτή είναι η γενική προσανατολισμή. Μα βρίσκουν συμφώνου και πέρα από τις περιφέρειες που μπορεί να αφορά αυτό άμεσα, πιστεύω ότι ο στόχος των ενδιάμεσων ε, στόχων μπορεί να προσαρμόσει την πολιτική συνοχή της Ευρώπης, να της δώσει μια πραγματική διάσταση εδαφικής ε, διαμόρφωσης. Μπορεί να είναι μακροοικονομικός σταθεροποιητικός παράγων και δίνει σημαντικό εργαλείο της στην Ευρώπη για να μπορεί να διχειρίζεται καλύτερα το μέλλον της και να εξασφαλίζει την ισότητα των ευκαιριών που έχουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες που κατοικούν στις περιοχές αυτές. Εν γέννη λοιπόν αυτά θα μπούμε σε μια φάση που θα εξετάσουμε σαφέστερα τις λεπτομέρειες. Ξέρω ότι σήμερα ότι δεν μπορείτε να μας δώσετε όλα τα στοιχεία, θα τα παρουσιάσετε τον ε, επερχόμενο Σεπτέμβριο. Έχω κάποιες ερωτήσεις όμως ε, και θα σας παρακαλούσα ή δυνατόν να απαντήσετε και να μην τις δυσμονήσετε, πάση περιπτώσει. Πρώτη ερώτηση. Σε αυτή τη νέα αρχιτεκτονική, ποιο είναι το μέλλον, με ποιο τρόπο θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των περιφερειών που βγαίνουν από το άρθρο 194 συνθήκη τη Αβώνα. Νησιά, οι υπερπεριφερειακέ ζώνε, αεροκατοικημένε, ορεινέ περιοχέ. Και πέραν αυτού, τι θα γίνει με το πρόβλημα των υπερπεριφερειακών περιοχών που είναι ένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Μετά υπάρχουν νέα πλαίσια που διαφαίνονται σήμερα στο τοπίο της πολιτικής συνοχής, κυρίως στις μακροπεριφέρειες. Πώς θα βρουν τη θέση τους στο μελλοντικό, στη μελλοντική πολιτική συνοχής. Και νομίζω ότι έχει τεθεί ήδη το επόμενο ερώτημα όσον αφορά το κοινό στατικικό πλαίσιο. Πώς διαθρώνεται ε, με το Ταμείο του Δεύτερου Πυλώνα για την Αγροτική Ανάπτυξη, με το Ταμείο Αλίας κλπ. Συνεχίζεται η συζήτηση λοιπόν, εγκρίνουμε τις γενικές γραμμές που ε, απορρέουν από την τελευταία ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από τις θέσεις ε, των διαφόρων επιτροπών συμπεριλαμβανομένης αυτής, αλλά νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε πιο πέρα. Και θα πρέπει να είναι εργαλείο πολιτικής συνοχής, πολύ καλά επεξεργασμένο, που θα μπορεί να συμβάλλει στην ευμάρεια των ευρωπαϊκών περιφερειών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά για την ΙΣΙΑ ο κύριος Βλάσακ προχώρα ο Βλάσακ. πάνε κομισάρι, ε, Ευχαριστώ. Αξιότιμε κύριε Επίτροπε, χαίρομαι για το ότι συμμετέχετε στη σημερινή συζήτηση και Ευχαριστώ και για τις παρεμβάσεις και απαντήσεις σας. Εκείνο από το ότι από την ομάδα μας η σκέψη των μεταβατικών περιφερειών είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη. Θα έλεγα ότι θα ήταν αναγκαίο αυτή η σκέψη να αναπτυχθεί όσον αφορά τις ε, χρηματοοικονομικές προοπτικές και τις πηγές άντλησης, δηλαδή από πού θα υπάρξει άντληση και μετάθεση κονδυλίων να αποσαφινιστούν όλα αυτά. Ένα πρόβλημα επίσης θα ήθελα να αναφέρω που ήδη από τον κύριο Λάμπερτ Φαν Ρόι ε, παρουσιάστηκε και αυτό είναι η κοινή στοχοθέτηση, η κοινή προσέγγιση και η κοινή προσανατολισμή των προγραμμάτων και σχεδίων. Έχουμε τη διαδικασία συναπόφασης που έχουμε εισαγάγει. Θέλουμε η αρχή της εταιρικής σχέσης να εφαρμόζεται πλήρως Λυπούμε ότι από στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας αγνοούνται κάποιες περιφέρειες ε, όταν σε κρατικό επίπεδο λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις οι ίδιες οι περιφέρειες και οι ίδιες οι μικρές ε, ε, ενότητες και μονάδες να μην αγνοούνται. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι εδώ θα υπάρχει ιεράρχηση στην λήψη αποφάσεων και ιεράρχηση αντιμετώπισης προτεραιοτήτων. Ένα άλλο πρόβλημα σε αυτή τη διαδικασία και αυτό είναι προς το συμφέρον μας να δράσουμε είναι οι δραστηριότητες για τους τελικούς αποδέκτες. Πρέπει να ξεκινήσουν τέτοιες ε, διαδικασίες ώστε να έχουν οι τελικοί αποδέκτες ε, σαφείς δυνατότητες για τα κονδύλια τα οποία θα τους παρέχονται στο τέλος στη συνδιαμόρφωση αυτών των μηχανισμών. Ποιες είναι οι προοπτικές για μηχανισμούς Jeremy, Jessica και Just Funds. Ξέρουμε ότι η απορροφητικότητα σε κάποιες δράσεις από αυτές είναι πολύ χαμηλή και έχουμε πληροφορίες ότι οι τελικοί αποδέκτες, οι δήμοι και οι κοινότητες δεν, γνωστο, δεν γνωρίζουν ακριβώς πώς θα πρέπει να εφαρμόσουν κανόνες για την ε, χρήση αυτών των κονδυλίων. Και θα πρέπει οι τελικοί αποδέκτες λοιπόν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία. Ευχαριστώ. Γεια. Uh, ευχαριστώ. Θα παρακαλούσα, μια και οι συντονιστές ολοκλήρωσαν και δεν έχουμε άλλους ε, από άλλη κατηγορία, ο Επίτροπος να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις και μετά θα ακολουθήσει ο γύρος με τα μέλη της Επιτροπής μας που θα παρέμβουν Επίτροπος. Το άρθρο 272. Όπως ε, αναφέρθηκε σε σχέση για παράδειγμα για τις αρεοκατοικημένες περιοχές στην Ήπεθρο πώς θα πρέπει να διασφαλίζεται η περαιτέρω στήριξη στη συνέχεια και αυτό συμπεριλαμβάνει και τη δυνατότητα να διατηρούνται και στο μέλλον τέτοιες δυνατότητες. Δηλαδή στο μέλλον να υπάρχει ελαστικότητα που θα διασφαλίζεται σε σχέση με κάποιες περιφέρειες όσον αφορά την χρήση των κονδυλίων μπορούν οι ίδιες οι περιφέρειες να θέσουν κέντρα βάρους, προτεραιότητες και να πούν σε συγκεκριμένα τμήματα αυτής της περιφέρειας πιο έντονα θα διατίθενται για συγκεκριμένους στόχους αυτές, αυτά τα κονδύλια. Διότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ πιο πλούσιων τμήματων και λιγότερο πλουσίων τμήματων σε μια περιφέρεια. Με αυτή τη διαφοροποίηση θα πρέπει να ε, δούμε αυτή τη δυνατότητα. Θα το χαιρετίζαμε, αλλά αυτό είναι κυριαρχικό δικαίωμα των εμπλεκόμενων περιφερειών και κρατών. Μπορώ να αναφέρω για πολλές ε, χώρες και περιφέρειες ότι αυτό ήδη κάποιες το εκμεταλλεύονται και το χρησιμοποιούν. Υπάρχει και η αρχή του, της κάνουλας από την οποία ε, διατίθενται κονδύλια. Όμως για τις μακροπεριφέρειες εδώ υπάρχει σαφές δρομολόγιο που λέει ότι εφέτος θα έχουμε την πρώτη ενδιάμεση έκθεση μετά για την περιοχή της Βαλτικής, μετά για την περιοχή του Δούναβη, της λεκάνης του Δούναβη και μετά στη συνέχεια μία έκθεση για το πώς η μακροπεριφερειακή ε, συνεργασία αναπτύχθηκε και ποιες επιδόσεις είχε. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη υπάρχει μια κάποια εφορία όσον αφορά τις μακροπεριφέρειες. Έχω καμιά φορά την εντύπωση ότι όταν μια χώρα δεν συναποτελεί τμήμα μιας τέτοιας ε, ε, δράσης θεωρούν ότι είναι μια χώρα δεύτερης κατηγορίας. Κατανοώ βέβαια ότι υπάρχουν και προσφέρονται σχεδόν παντού στην Ευρώπη μακροπεριφερειακές προσεγγίσεις ή δυνατότητες προσέγγισης στη συνεργασία και ανάπτυξη. Πάντα όμως θέλω να επισημαίνω και επισημαίνω ότι και για το μέλλον εδώ δεν πρέπει να πούμε ότι θα προβλέπονται πρόσθετα ατέλειωτα κονδύλια και ότι όλες αυτές οι περιφέρειες ή αυτές οι στρατηγικές μόνο τότε θα έχουν νόημα και αποτέλεσμα όταν πραγματικά χειροπιαστά Έχουμε κοινό συμφέρον και κοινή στοχοθέτηση. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω, μέσω συνεργασίας και συντονισμού αρκετών περιφερειών και αρκετών χωρών, περισσότερων χωρών και περισσότερων περιφερειών. Η μακροπροσέγγιση δεν μπορεί να οδηγεί στο ότι προβλήματα που υπάρχουν σε μια περιφέρεια και που αυτόματα μπορούν να επιληθούν από πλευράς αυτής της περιφέρειας θα μετατίθενται ή θα μεταφέρονται στο μάκρο επίπεδο πόλη συνεργασίας. Γι' αυτό και για την στρατηγική για τον Δούναβη. Μόνο εκείνα τα θέματα μπορεί να καλύπτει και να εξετάζει που έχουν μια διασυνοριακή συνιστόσα στη συνεργασία και πρέπει να υποστηρίζονται. Για το θέμα της ποιότητας του νερού του Δούναβη και των ε, ποταμών που εκβάλλουν στον Δούναβη κατά τον Ρούτου. Δεν είναι δυνατόν μία χώρα ή μία περιφέρεια να επιλύσει όλα αυτά τα προβλήματα. Και για την οικονομική ανάπτυξη και τα λοιπά. Υπάρχουν διαφορετικοί τομείς, αλλά υπάρχουν και θέματα που εντάσσονται ή άλλα που δεν εντάσσονται σε μια μακροστρατηγική. Είναι σημαντικό να καθορίσουμε και να διαφοροποιήσουμε αυτά τα θέματα. Bottom-up στρατηγικές, εκ των κάτω προς τα άνω. Καμιά από αυτές τις στρατηγικές δεν εκπηγάζει, δεν ξεκινά από τις Βρυξέλλες. Επιτόπου από εκεί προέρχεται αυτή η στρατηγική και πρωτοβουλία. Και πρέπει να παραμείνει αυτό ως πραγματικότητα έτσι. Οι ίδιες οι περιφέρειες να δραστηριοποιούνται και για τον υψηλό βαθμό εξειδίκευσης σχεδίων και προγραμμάτων πάλι οι ίδιες οι περιφέρειες είναι αρμόδιες. Για τον συνάδελφο Βλάσακ και πάλι market level. Ε, γι' αυτό το έχουμε αναφέρει στο σχέδιο κανονισμού αυτό. Αυτό είναι ο λόγος. Πρώτα απ' όλα, από την άλλη βέβαια πλευρά πρέπει ξεκάθαρα και σταράτα να πω ότι φυσικά το συνταγματικό πλαίσιο και τους συνταγματικούς όρους πλαισίου μιας χώρας πρέπει να, το σεβό, να τους σεβόμαστε. Υπάρχουν κάποιες χώρες, π.χ. Γερμανία, που βρίσκονται πάνω-πάνω όσον αφορά την αρμοδιότητα των ομοσπονδιακών κρατηδίων και απορρέει η ανάγκη αυτόματα να εμπλέκονται και τα ομοσπονδιακά κρατήδια σε αυτές τις διεργασίες. Υπάρχουν άλλες χώρες όπου υπάρχει πολύ κεντρική δομή και εξειδικευμένη κεντροποίηση. Και εδώ πρέπει να διαφοροποιούμαστε. Πάλι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και να δεχόμαστε αυτές τις διαφορές και να τις σεβόμαστε. Δεν αλλάζει τίποτα και πάλι το επαναλαμβάνω εμείς στους κανονισμούς να εγγράψουμε και θα το εγγράψουμε και αυτή θα είναι η πρότασή μας ότι οι περιφέρειες και στο βαθμό του εφικτού και το περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και οι και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, οι ΜΚΟ, θα πρέπει όλες και όλοι να εμπλέκονται, ώστε με τον σωστό τρόπο να μπορούν να δράσουν. Ευχαριστώ για την επισήμανση, να μην χαλαρώσουμε και να συνεχίσουμε τις προσπάθειες. Οι περιφέρειες παραπονούνται ότι από το εθνικό επίπεδο αγνοούνται. Το τοπικό επίπεδο παραπονείται ότι αγνοείται από τις περιφέρειες. Λοιπόν, όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να είναι σεβαστοί και ο ένας να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες του άλλου και να ανταποκρίνεται σε αυτές. Τώρα, αυτό συμπεριλαμβάνει και τον τομέα της συγχρηματοδότησης. Αυτό επανειλημμένα και πολλαπλά είναι έλλειμμα ή έλλειψη πληροφόρησης για όσους δεν το γνωρίζουν και λιγότερο ένα θέμα της καθαρής συγχρηματοδότησης ή δυνατοτήτων συγχρηματοδότησης. Πολλές δυνατότητες υπάρχουν και μέσω πιστώσεων και δανείων που προσφέρονται. Υπάρχουν όμως, υπάρχει έλλειμμα στην πληροφόρηση και πρέπει να διαχέουμε πληροφορίες, να τις διαδίδουμε ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση όσον αφορά την ενημέρωση. Μεταβατικές ή προσωρινές ε, περιφέρειες. Είναι σημαντικό στο πλαίσιο του προϋπολογισμού να δράσουμε σωστά. Όταν μειώνεται ο αριθμός των περιοχών συνοχής είναι λογικό ότι απελευθερώνονται κονδύλια, αποδεσμεύονται κονδύλια Πρέπει να διαρωτηθούμε ποιος είναι ο πιο ευφυής τρόπος να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα αποδεσμευμένα, απελευθερωμένα κονδύλια, ώστε να αναπτυχθούν περαιτέρω και με τον καλύτερο τρόπο κάποιες περιφέρειες στην Ευρώπη. Και γι' αυτό καταλήγουμε σε αυτή την κλιμακούμενη προσέγγιση, βήμα προς βήμα σταδιακά σε κλιμάκωση. Ευχαριστώ. jetzt läuft uns die Zeit. Σε ευχαριστώ. Τώρα όμως πιέζει κάπως ο χρόνος, περισσότερο πιέζει όχι λόγω της κυρία Σρέτερ και το ομολογώ αυτό, όχι επειδή πρόκειται να παρέμβετε, αλλά παρόλα αυτά θα ήθελα και εγώ να πω σύντομα δύο λόγια για αυτά που ανέφερε ο Επίτροπος. Είναι σαφές όταν λιγότερες ε, περιφέρειες εντάσσονται σε μια κατηγορία, τότε υπάρχει ίσως και μεγαλύτερο δυναμικό. Πρέπει να δημιουργηθεί μια σαφής σταθερή δομή, σταθερή δομή και να υπάρχει και μια μεταβατική ενδιάμεση κατηγορία. Και όταν υπάρχει δεδομένο ποσό, και αυτό δεν μεγεθύνεται, θα πρέπει αυτή η κατηγορία σε ανταγωνισμό με άλλες, με στο στόχο 1, 2, να μπορούμε να δούμε από πού θα αντλήσει κονδύλια. Είναι λογικό συμπέρασμα αυτό και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Η κυρία Σουρέτερ παρακαλώ. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε που μου δίνετε τον λόγο. Κίνητρο ιδιαίτερο είναι αυτό, επιπρόσθετα να απαντήσω επί της ουσίας να υπάρξει τοποθέτηση σε κάποια θέματα παρατηρώ ότι εκμεταλλεύεστε κάθε δυνατότητα να έχετε την πλειοψηφία στο πλευρό σας. Όμως δεν υπάρχει αυτή η πλειοψηφία στο πλευρό σας. Είχαμε δύο ψηφοφορίες, μία στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή και μία στην Ολομέλεια και δύο τρίτα για την πρόταση αποδείχθηκε ότι υπήρχε σαφής πλειοψηφία, νομοθετική πλειοψηφία μπορούμε να πούμε ότι αυτή την πρόταση για μια ενδιάμεση κατηγορία την θεωρούμε σκόπιμη, ισορροπημένη πρόταση και έχει την σαφή πλειοψηφία των μελών του Ευρωκοινοβουλίου. Ακόμα και αν υπάρχουν κάποιοι που σε αυτό το σημείο θεωρούν ότι θα έπρεπε να αλλάξουν την κατάσταση και να ανατρέψουν την κατάσταση. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι κάποιες χώρες θέλουν να ανοίξουν την κάνουλα και να πάρουν περισσότερα κονδύλια, όμως θέλουν να δώσουν λιγότερα κονδύλια μέσω της αλληλεγγύης. Και παρότι υπάρχουν ιδιαίτερες ανάγκες από τις περιφερειές τους. Ένα άλλο θέμα θα ήθελα να θίξω, το οποίο σήμερα όμως δεν καλύφθηκε. Και αυτό είναι το θέμα των όρων και προϋποθέσεων. Η Επιτροπή από ό,τι κατάλαβα τουλάχιστον από το χαρτοφυλάκιό της υπέβαλε κάποιες προτάσεις. Υπάρχουν διαφορές, υπάρχουν προτάσεις δικές σας που λένε ότι πρέπει να υπάρχει μια ποιότητα που θα διασφαλίζεται στην παρέμβαση. Ποιοτικά αναβαθμισμένες προϋποθέσεις μέσω νομοθετικού έργου ή νομοθετικού πλαισίου και διαχείρισης, ώστε στοχοθετημένα τα, κονδύλια, τα διαθετικά κονδύλια να μπορούν να χρησιμοποιούνται σωστά. Το υποστηρίζουμε πολύ αυτό. Δεν είπατε όμως κάτι περισσότερο και το βρίσκω κρίμα. Για μας στην Επιτροπή μας είναι πολύ σημαντικό. Εμείς είμαστε κατά της ε, ε, πρότασης ε, όσον αφορά σε σχέση με την επιβολή των μακροοικονομικών όρων. Νομίζουμε ότι αυτές οι προτάσεις μακροοικονομικών όρων δεν την χάνουν πλειοψηφία. Πάει αυτό το θέμα λοιπόν σβήνει. Όμως αυτός ο όρος που προτάθηκε από εσά, δηλαδή να είμαστε προετοιμασμένοι κάποια πράγματα να τηρούνται οπωσδήποτε, βρίσκουμε ότι είναι πολύ καλή πρόταση εμείς και θα μα ενδιαφέρει, θα με ενδιαφέρει να δω πώς το προτείνεται αυτό, πόσο χειροπιαστό και εξειδικευμένο είναι. Ποια επιμέρους κριτήρια εξειδικευμένα θα δεσμεύσετε και θέλω να σας υποστηρίξω σε αυτό το εγχείρημα να παραμείνετε πιστός και να μην χαλαρώσετε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ συνάδελφε. <coughs> Ρίτα παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον Επίτροπο. Πολλά θέματα αναφέρθηκαν προηγούμενα και καλύφθηκαν. Ένα από αυτά θα ήθελα παρόλα αυτά εγώ ιδιαίτερα να το αναφέρω και να το τονίσω που συνδέεται με το άρθρο 74 βλέπετε ο Επίτροπος ε, στην παρέμβασή του απάντησε σχετικά και είπε ότι πρέπει να υπάρχει συντονισμός για τα κονδύλια. Και τώρα θέλουμε με το άρθρο 74 να μπορέσουμε να καταφέρουμε οι περιφέρειες εκείνες να καλυφθούν που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις ή πιέσεις. Και θα ήθελα σε σχέση με αυτό να ε, ε, επισημάνω στον Επίτροπο ότι αυτές οι περιφέρειες και στο μελλοντικό νομοθετικό έργο θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Έχουμε την έκθεση Πίπερ από το Ευρωκοινοβούλιο όπου ακριβώς υπέρ αυτών των περιφερειών υπάρχει τοποθέτηση και αναπτύσσονται επιχειρήματα. Και ακριβώς όσον αφορά την χρηματοδότηση των αναγκών αυτών των περιφερειών. Και δεύτερον, εκεί όπου θα είχα εγώ την ερώτησή μου προς τον Επίτροπο, συγκεκριμένα κιόλας όσον αφορά το σύστημα CBC, CBC, δηλαδή της ε, πολιτικής γυτνίασης ε, στην Ευρώπη. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Κάνουμε λόγο για την ανάπτυξη της δημοκρατίας, ιδιαίτερα στην ε, βόρεια όχθη της Αφρικής, αλλά να μην ξεχνάμε και τη Ρωσία σε όλα αυτά. Είναι το μόνο μέσο χρηματοδότησης το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας ώστε η δημοκρατία στη Ρωσία να μπορέσει να προαχθεί και να τονωθεί. Είναι κάτι το οποίο έχει μεγάλη σπουδαιότητα και πρέπει να μην το αγνοήσουμε. Αυτή τη στιγμή Πρόκειται, θα έλεγα, για μέσα ή εργαλεία για την ε, συνεργασία της ανάπτυξης, που πολλές φορές συνδέονται και με κάποια προβλήματα, όπως με τη Ρωσία εξειδικευμένα. Όμως ως γείτονες της Ρωσίας χρειαζόμαστε ένα εξειδικευμένο ή εξειδικευμένα προγράμματα για την προαγωγή της δημοκρατίας. Και αυτό σημαίνει μια εταιρική σχέση και συνεργασία και ανάπτυξη της εταιρική σχέσης και συνεργασίας με τους γείτονές μας Ρώσους. Θέλω να ρωτήσω τον Επίτροπο, η συζήτηση σε σχέση με αυτά τα θέματα έχει προαχθεί ότι αυτό το θέμα αυτή της συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο θα έπρεπε να ενταχθεί ώστε για παράδειγμα οι δυνατότητες διαχείρισης στις περιφέρειες θα πρέπει να είναι δεδομένες για να εκμεταλλευτούν τέτοιες ε, δυνατότητες, τέτοια μέσα, διότι αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν τα άλλα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. μας παρακαλώ. Köszönöm σας ευχαριστώ που μου δίνετε τον λόγο. Αξιότιμη Επίτροπε, θα είχα δύο ερωτήσεις και θα ήθελα σύντομα να τοποθετηθώ ώστε να έχουν και άλλοι συνάδελφοι τη δυνατότητα να παρέμβουν μετά από μένα και εκείνοι. Η πρώτη ερώτηση αφορά αυτή την ενδιάμεση προσωρινή μεταβατική κατηγορία. Αναφέρθηκαν κάποια πράγματα σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το θέμα σήμερα, αλλά και την Πέμπτη θα αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα όταν θα έρθει η ώρα να ψηφίσουμε. Έχω και εγώ τις προσωπικές μου απόψεις που είναι γνωστές μέσα στο πλαίσιο των μελών της κοινοβουλευτικής μας επιτροπής. Υποστηρίζω τον κύριο Πίπερ σημερινό προεδρεύοντα την ε, δική μας κοινοβουλευτική επιτροπή σήμερα. Υποστηρίζω τη γνωμοδότηση, την τοποθέτηση μια πολιτική, ε, ένα πολιτικό προβληματισμό θέλω να αναφέρω. Είναι σημαντικό το θέμα για τις περιφέρειες και τη συνεργασία τους. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το θέμα όμως αποτελεί μήλο της έρηδος. Και θα έλεγα για τις ενδιάμεσες περιφέρειες υπάρχουν θέματα που είναι πιο σημαντικά. Και παρόλα αυτά, κύριε Επίτροπε, και εδώ στην δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή, στις δικές μας αντικειμενικές συζητήσεις υπάρχουν άλλα θέματα που είναι πιο σημαντικά από το θέμα των ενδιάμεσων περιφερειών. Πιστεύω ότι πέφτουμε σε παγίδα που δημιουργούμε, με αυτή την παγίδα που δημιουργείται και συζητούμε αποκλειστικά αυτήν των ενδιάμεσων περιφερειών. Αυτά τα θέματα δηλαδή αναφέρθηκαν και θέματα ενδιάμεσων περιφερειών, υπάρχουν όμως άλλα θέματα τα οποία είναι πιο σημαντικά Συνεργασία μεταξύ των περιφερειών για παράδειγμα. Και αν δούμε την κατάσταση πώς έχει διαμορφωθεί σήμερα, αν τραβούσαμε μια διαχωριστική γραμμή και κάναμε έναν απολογισμό, θα έλεγα ότι ο περισσότερος χρόνος στις ερωτήσεις, στις απαντήσεις, στις ε, αναλύσεις, ο περισσότερος χρόνος δόθηκε σε αυτές τις ενδιάμεσες περιφέρειες. Θα έχουμε τις νέες δημοσιονομικές ε, προοπτικές, θα έχουμε την πολιτική συνοχή, χρειάζονται πολλά κονδύλια για όλες αυτές τις δράσεις. Εμείς ασχολούμαστε με θέματα πολιτικής συνοχής και εκεί εσείς κύριε Επίτροπε αρμόδιοι για αυτά τα θέματα κάνετε τα σωστά βήματα που είναι αναγκαία για την πολιτική συνοχής, όμως αν μια ιεράρχηση προτεραιοτήτων γίνει και υπάρχει μια σαφής πολιτική, θα ήθελα να κρούσω κόδωνα κινδύνου, να μην θέσετε τις ενδιάμε, την ενδιάμεση κατηγορία αυτών των προσωρινών περιφερειών ως πρώτη σας προτεραιότητα. Τώρα, τούτου λεχθέντος, όσον αφορά τις λύσεις, τις καλοχαιρετίζουμε τις προτάσεις ε, επίλυσης των προβλημάτων και λύσεων που προτείνεται. Τέλη Σεπτεμβρίου θα έχουμε αυτές τις προτάσεις που θα αντανακλώνται από πλευρά σας ε, μέσα στο πλαίσιο κανονισμών. Για την πολιτική όμως ε, δομή, κύριε Επίτροπε, το αναφέρατε αυτό, για αυτή την ανάπτυξη αυτών των στοιχείων θα ήθελα η εξή ε, σκέψη να ληφθεί υπόψη. Θεσμικά είναι πολύ σημαντικό να παραμείνουμε στο ΑΕΠ ως δίκτυ ή πύχη Δηλαδή, ε, σε εκείνες τις περιφέρειες που είναι χαμηλό το ΑΕΠ να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Είναι πολύ σημαντικό στις περιφέρειες όπου υπάρχουν προβλήματα και αντίθετα σε περιφέρειες που είναι πολύ υψηλό το ΑΕΠ, εκεί δεν επιτρέπεται να κάνουμε να αναλαμβάνουμε δράσεις όταν πρόκειται για περιφέρειες που ευημερούν Πρέπει να βοηθούμε και να υποστηρίζουμε εκείνες τις περιφέρειες και χώρες όπου είναι χαμηλότερο το ΑΕΠ τους. Μετάθεση πόρων. Μετάθεση πόρων είναι ο σωστός όρος. Η μετάθεση όμως κονδυλίων <coughs> από τις χαμηλότερες περιφέρειες προς τις υψηλότερες όσον αφορά το ποσοστό ΑΕΠ δεν είναι η σωστή πορεία. Είναι η λανθασμένη πορεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Τόμας Τόιτς. Κονίλια Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Λοιπόν, για το θέμα που συζητάμε, πρέπει να πω ότι η συζήτηση ε, δείχνει ότι διαμορφώνεται μια κάποια συμφωνία στην, ε, στην όλη ομάδα. Λοιπόν, εάν ακολουθήσουμε διαφορετικό σύστημα, ε, ίσως ένα διαφορετικό το αποτέλεσμα. Θα πρέπει όλοι να ακολουθήσουμε το σύστημα αυτό με το οποίο συμφωνούμε όλοι. Και ε, στην επόμενη φορά πρέπει αυτό να το λάβουμε υπόψη. Λοιπόν, ο προλαλής σας συνάδελφος έλεγε ότι μάθαμε πολλά από αυτή την ενδιάμεση κατηγορία και αυτό είναι σωστό. Από την άλλη πλευρά πρόκειται και περί καινοτομίας. Γι' αυτό υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, πολλά εκρεμή ζητήματα και αυτό που αναφέρθηκε ε, εκτενώς σαν θέμα. Υπάρχουν πολλά πράγματα λοιπόν τα οποία είναι ασαφή όσον αφορά την καινοτομία αυτή. Εγώ θα έλεγα το εξή. Αν δούμε τις διάφορες περιφέρειες που παραθέσατε εσείς κύριε Πρόεδρε, ε, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές οι περιφέρειες της σύγκλησης όπως αποκαλούνται, έχουμε τις περιφέρειες όπου αντιμετωπίζουν οικονομική κρίση και αρχίζουν να απομακρύνονται από τις περιοχές σύγκλησης. Περνάει όλη η Ένωση μια κρίση. Λοιπόν υπάρχουν αυτές τις διαφορές και θέτω το ερώτημα. Υπάρχουν αυτές οι διαφοροποίησεις λοιπόν. Υπάρχουν οι διαφοροποίησεις, λαμβάνονται υπόψη αυτές οι διαφορές στην ενδιάμεση κατηγορία. αυτές οι 51 περιφέρειες. Πώς έχουν προσμετρηθεί, με ποιες παραμέτρους, ποια διαδικασία χρησιμοποιήθηκε. Μπορώ να πω κάτι ακόμα. Μπορώ να πούμε κάτι πάνω σε αυτό. Λοιπόν, μετά τα ποσοστά υψηλότερη υποστήριξης, αυτό που αναφέρατε σε αυτές τις κατηγορίες, και αυτό είναι ερωτηματικό. Υπάρχει και άλλη προβληματική μετά. Η διασυνοριακή συνεργασία η οποία θα πρέπει να είναι ακόμα καλύτερη. Όπως έλεγε ο κύριος Βανίστελρο και έχει απόλυτα δίκιο σε αυτά που έλεγε. Ξέρω ότι στη δική μου περιοχή, στην Ανατολική Γερμανία, ακούγονται κάπως επικρίσεις όσον αφορά τη συμβατότητα που έχουν τα μέσα που διατίθενται και τα κίνητρα που δίνονται για την πρόσβαση στην α, βοήθεια. Ότι χρειάζονται απλουστεύσεις. Έχετε προτάσεις όσον αφορά τη διευκόλυνση αυτής της διασυνοριακής συνεργασίας. Ε, για να το πω προσεκτικά. Και θα ήθελα να ακούσω ποια είναι η θέση όσον αφορά αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν και άλλα σημαντικά θέματα και όχι μόνο ενδιάμεσες ε, περιφέρειες, όπως αναφέρθηκε. Η ποιότητα της βοήθειας έχει σημασία. Οι ενδιάμεσες λοιπόν περιφέρειες είναι ένα βασικό θέμα το οποίο συζητάμε εδώ σήμερα, αυτή η ενδιάμεση κατηγορία και βέβαια έγιναν διάφορες συμφορίες στο Κοινοβούλιο, διαμορφώθηκαν σαφείς πλειοψηφίες, όμως εξακολουθεί να είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί και να κουβεντιαστεί. Σε όλα τα άλλα ζητήματα νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε. Υπάρχει συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπής και Κοινοβουλίου, αλλά πρέπει να συζητήσουμε αυτή την ενδιάμεση κατηγορία των περιφερειών έτσι περαιτέρω. Είναι κάτι που προτείνουμε να εισαγάγουμε και θέλουμε να δούμε πώς θα πάει μετά την εφαρμογή του, να δούμε τι θα γίνει στο άμεσο μέλλον όταν εφαρμοστεί αυτή η προσέγγιση. Δεν είναι ότι παίρνουμε μία απόφαση για τον υπόλοιπο αιώνα τώρα. Απλώς συζητούμε τη νέα οικονομική περίοδο, τι θα κάνουμε, τι κανονισμούς θα χρειαστούμε, τι μέτρα θα χρειαστούμε. Άρα δεν λέμε ότι αλλάζουμε εντελώς κατεύθυνση με αυτά τα μέτρα. Αντιθέτως, εγώ βλέπω ότι αυτές οι αλλαγές δημιουργούν ευκαιρίες, δυνατότητες. Και ίσως τελικά δούμε ότι οι διάδοχοί μας θα πούν ότι αυτό το μέσο, αυτή η κατηγορία, των, η ενδιάμεση των περιοχών είναι κάτι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι το τέλος της νέας δημοσιονομικής περίοδου. Μετά μπορούμε να αποτιμήσουμε τα αποτελέσματα, να δούμε ποια είναι η ποιότητα των αποτελεσμάτων και τι κάνουμε από εκεί και πέρα. Θέλουμε να δούμε κάθε περιφέρεια, κάθε πρόγραμμα που εφαρμόζεται κάθε περιφέρεια, να θέσουμε ποσοτικοποιημένους στόχους και για τις ενδιάμεσες περιφέρειες και για τις περιφέρειες της σύγκλησης. Θέλουμε να θέσουμε στόχους, να στοχοθετήσουμε και να δούμε αν θα πετύχουμε τους στόχους. Εάν πετύχουμε τους στόχους, όλα καλά και άγια. Αν δεν πετύχουμε τους στόχους, θα πρέπει να αναλύσουμε για ποιο λόγο δεν πετύχαμε αυτούς τους στόχους. Βέβαια, άμα περάσει κάποιο χρονικό διάστημα και αν υπάρχουν περιοχές σύγκλησης, του τομέα σύγκλησης, που πάνε καλά θα κάνουμε την αποτίμηση. Θα δούμε αν υπάρχουν κενά, ποια είναι τα προβλήματα, ποια είναι τα προβλήματα του, των προγραμμάτων. Και όλα αυτά και πόσο απέχουν οι επιτυχίες των προγραμμάτων από τους στόχους που είχαμε θέσει. Να δούμε ποια απόκληση υπάρχει. Και θα δούμε τελικά μετά από ένα χρονικό διάστημα τι πετύχαμε, τι δεν πετύχαμε. Αν οι περιοχές σύγκλησης λοιπόν πετυχαίνουν τους στόχους, αν τα χρήματα που διατέθησαν χρησιμοποιούνται σωστά, με τον ευταίο τρόπο και όταν γίνει η αποτίμηση, η αξιολόγηση θα δούμε πώς μπορούμε να αποτιμήσουμε τη γενική ποιότητα των πεπραγμένων των αποτελεσμάτων. Θα δούμε λοιπόν τι καρπούς δίνουν αυτά τα μέτρα και αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε τι πρέπει να κάνουμε, πώς μπορούμε να αποτιμήσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα προγράμματα πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις παρεμβάσεις έτσι περαιτέρω για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Και ένα τελικό σχόλιο έχω πάνω σε αυτό που μας πηγαίνει λίγο πιο πέρα αυτό που θα πω. Ε, αλλά αναφέρομαι σε κάτι που είπε και ο κ. Ντόιτς. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να καταλάβουμε κάποια πράγματα να δούμε την περιφερειακή πολιτική πώς είναι, τι μορφή έχει. Δεν είναι μια πολιτική που εξυπηρετεί ιστορικούς στόχους αποκλειστικά, δηλαδή να ξεπεραστούν οι οικονομικές αντιθέσεις που υπάρχουν και μόνο, πρέπει να δούμε ότι έχουμε στα χέρια μας ένα εργαλείο που θέλει γενικά να προωθήσει ευρωπαϊκά προγράμματα σε σφαιρικό επίπεδο, σε γενικό επίπεδο. Και αυτό ε, θα πρέπει να επηρεάζει το πώς θα χρηματοδοτούνται τα διάφορα προγράμματα. Αυτή η έποψη. Τι θέλουμε να κάνουμε λοιπόν, θέλουμε να προσφέρουμε σε κάθε περιφέρεια οικονομικές δυνατότητες να μπορέσουν να γίνουν πιο αποδοτικές αφορά τη χρήση της ενέργειας, να μειώσουν την ανεργία, να καταπολεμήσουν τη φτώχεια, να πετύχουν διάφορους στόχους, να μπορούν οι περιφέρειες να κάνουν περισσότερη έρευνα. Αυτά πρέπει να προωθήσουμε και εδώ θα πρέπει να διαθέσουμε τα κατάλληλα μέσα, να δώσουμε τα κατάλληλα οικονομικά κίνητρα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι ε, συνεκτικό Νομίζω ότι τα κράτη-μέλη όσον αφορά τους στόχους για το 2020 με τα χρήματα που διαθέτουν, με τους προπολογισμού που διαθέτουν θα τα καταφέρνουν πολύ καλύτερα με τα ευρωπαϊκά κίνητρα βλέποντας ποια είναι η οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη σήμερα. Θα ήταν αφελές να πιστεύουμε κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό η Ευρώπη πρέπει να δώσει σε ένα πλαίσιο συμπροματικά ποσά για να πετύχουμε τους στόχους που όλοι έχουμε συμφωνήσει. Όλοι, από κοινού. Τώρα, έχουμε 51 περιφέρειες. Ο αριθμός των περιφερειών, ο αριθμός αυτός είναι προσωρινός. Θέσαμε ένα προσωρινό αρχικό αριθμό και ελπίζουμε να έχουμε πιο επικαιροποιημένα στοιχεία στο μέλλον για να χρησιμοποιήσουμε. Αν δούμε τις μέσες τιμές της τελευταίας τετραετίας, αυτό κάναμε, πήραμε αυτά τα στοιχεία, βγάλαμε μέσω όρους. Όταν έχουμε πιο πρόσφατα στοιχεία θα δούμε αν η κατάσταση διαμορφώνεται διαφορετικά. Τα στοιχεία που σας έδωσα είναι βασικά στοιχεία, είναι κάποιες ενδείξεις αυτές ε, παρουσιάζουν την παρούσα κατάσταση. Η κατάσταση θα αλλάξει αναφυσβήτητα σε κάποιες περιφέρειες. Όσον αφορά την ποιότητα των παρεμβάσεων που εφαρμόζουμε, την ποιότητα των στόχων που έχουμε θέσει, έχουμε την ιδέα της αιρεσιμότητας που εφαρμόζουμε. Ε, πιστεύουμε ότι τα κράτη-μέλη, εάν τους πούμε, εάν τους πούμε ότι πρέπει να ενταχθούν στη διαθωτική πολιτική θα δεχτούν κάποιους όρους, θα δεχτούν αυτούς τους όρους. Νομίζω ότι μάλλον έγινε άτυπο Συμβούλιο Υπουργών επί Ουγγρικής ε, Προεδρίας εδώ και μερικές εβδομάδες. Συζητήθηκε το θέμα, ήρθαμε και σε επαφή με την ομάδα υψηλού επίπεδου και μάθαμε ποια είναι τα συμπεράσματα της ομάδας και όταν λήξει η συζήτηση η οποία συνεχίζεται θα δούμε τι θα κάνουμε. Αυτό που μας προβληματίζει είναι ότι θέλουμε να αυξήσουμε, να βελτιώσουμε την ποιότητα των μέτρων που λαμβάνουμε, των αποτελεσμάτων που πετυχαίνουμε. Για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες. Θα πρέπει να μπορέσουμε να ακούσουμε τις προτάσεις που κάνουν τα διάφορα κρατημέλη, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν εκεί. Να δεχτούμε, να διαμορφώσουμε τα σωστά, σωστά πλαίσια, ούτως ώστε τα κράτη-μέλη να πάψουν να έχουν δισταγμούς όσον αφορά ε, τις προτινόμενες ε, ποσοστώσεις, τα διάφορα νούμερα προτείνουμε. Διαφορετικά ε, μπορούμε να προσαρμόσουμε δεόντως το νομικό πλαίσιο, τις, τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν όπου αυτό παραστεί αναγκαίο. Και ίσως θα μπορέσουμε να εισαγάγουμε κατά αποκοπήν ποσά, εάν αυτό παραστεί αναγκαίο βέβαια, ε, για τα διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Εάν περιφερειακοί οι κανόνες δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο, τα πλαίσια που υπάρχουν δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο και που, ή που είναι οι περιφέρειες ότι δεν χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο, εντάξει, έστω. Ίσως ε, διαφανεί ότι υπάρχουν κάποιες διατάξεις τοπικές για τις δημόσιες προμήθειες ή κάποιες τοπικές διατάξεις για το περιβάλλον ε, που δυσκολεύουν τα πράγματα και ίσω να μην ενσωματώνεται η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία το περιβάλλον στην Εθνική Νομοθεσία. Οπότε, εν αυτή περιπτώσει, κάποια προγράμματα δεν μπορούν να προχωρήσουν. Αυτέ είναι οι συνθήκε που πρέπει να αλλάξουν, ούτω ώστε αυτά που εγκρίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο να μπορούν να εφαρμόζονται και στο τοπικό επίπεδο. Λοιπόν, η κυρία Μάνα. Όσον αφορά το θέμα των περιφερειακών ζητημάτων, Ε, συζητήθηκε το θέμα για τις συνθήκες εργασίας στη Λαπωνία. Έγινε συζήτηση, είναι πιο, από τις πιο δύσκολες περιοχές στην Ευρώπη. Για περιοχές όπως είναι η Λαπωνία, υπό δύσκολες συνθήκες θα υπάρξει ειδική συζήτηση για αντιμετώπιση. Όσον αφορά τη συνορική συνεργασία, για να πάρουμε το παράδειγμα της Ρωσίας, ε, εδώ είναι πολιτικό θέμα και όχι διοικητικό θέμα που αφορά και την Κροατία, η Ρωσία θα δώσει τεράστια σημασία στην συνεργασία και την ε, σύμπραξη, αν θέλετε. Τη συνεργασία. Δίνει μεγάλη σημασία σε αυτό το θέμα. Και δεν θα πρέπει να αισθανθούν ότι δέχονται από εμά αναπτυξιακή ε, βοήθεια. Άρα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποια πολιτική σύνεση σε πολιτικά δέστητα ζητήματα αν θέλουμε να πετύχουμε αυτά που θέλουμε σε διασυνοριακή συνεργασία. Γι' αυτό θα χρειαστούμε διάφορα προγράμματα διασυνοριακού χαρακτήρα ε, θα πρέπει να επικρατεί, να ακολουθηθεί μια προσέγγιση για ισότιμη αντιμετώπιση. Αν δείτε ποια είναι η δομή των διαφόρων προγραμμάτων, η δομή των προγραμμάτων δεν ε, πρόκειται να αλλάξει. Κάποια προγράμματα θα βασίζονται επί σχεδίων, ε, κάποιες δράσεις θα βασίζονται επί συγκεκριμένων προγραμμάτων, αλλά ουσιαστικά, βασικά, πρέπει να δει κανείς ποιες είναι οι διοικητικές δυνατότητες που προσφέρονται και ποιες διοικητικές βελτιώσεις μπορούν να επιτευχθούν για την καλύτερη εφαρμογή των προγραμμάτων. Ελπίζω να κατάφερα να ικανοποιήσω αυτούς που έθεσαν τις ερωτήσεις. Έχουμε δύο ομάδες ε, τεσσάρων αγοριτών, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Εστέ σύντομη, ε, ο Σον Κέλλη. Και παρακαλώ και τον Επίτροπο να είναι σύντομο. Σε ευχαριστώ, λέει ο κ. Κέλλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναμφισβήτητα η περιφερειακή πολιτική υπήρξε πάρα πολύ επιτυχής εν γέννη σε όλη την Ευρώπη και φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει καμία χώρα που να είναι καλύτερο ε, παράδειγμα από την χώρα μου. Μπήκαμε το 1973 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΑΕΠ μας ήταν 40% ε, του μεσοόρου και τώρα είναι 120% του μεσοόρου. Αλλά μακροπρόθεσμα αν θέλουμε να πετύχει η πολιτική συνοχής, κάθε περιφέρεια θα πρέπει τελικά να βγει από τη σύγκληση και να γίνει ανταγωνιστική και τότε θα πετύχει η περιφερειακή πολιτική. Αναφέρθηκαν κάποιες δυνατότητες ενδιάμεσες κατηγορίες. Αναφέρθηκε σε μία από τις λύσεις για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της ε, πολιτικής. Και Νομίζω ότι είναι θετικό αυτό, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που θα πρέπει επίσης ε, να εξεταστούν. Δηλαδή, η κατηγοριοποίηση των περιφερειών αυτών καθ' αυτών. Εν γέννη είναι πολύ τεχνητή και αυθαίρετη κατηγοριοποίηση. Εντός περιφερειών υπάρχουν τεράστιες ε, διαφορές και αναφέρατε ο ίδιος το Λονδίνο που έχει ένα ΕΠ 380%. Ήμουν στο Λονδίνο την περασμένη εβδομάδα με την Κόνσταντς και τα άλλα μέλη της ε, Επιτροπής, Περιφερειακής Επιτροπής στην αντιπροσωπεία και είδαμε στην περιοχή των Docklands, του λιμανιού του Λονδίνου, μεγάλη φτώχεια που παίρνει χρηματοδότηση και χρειάζεται πολύ περισσότερη. Άρα, μήπως μακροπρόθεσμα αξίζει τον κόπο να έχουμε πολλές περιφέρειες εντός των περιφερειών, όπου είναι σαφές ότι είναι πολύ κάτω από το μέσο όρο της γενικότερης περιφέρειας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα και θα ήθελα να ρωτήσω να μας πει ο Επίτροπος ποια είναι η απόψή τους. Και το ΑΕΠ ήταν λίγο πολύ το αποκριστικό κριτήριο για την αξιολόγηση της θέσεως μιας περιφέρειας. Είναι κάτι αυτό που θα πρέπει να αλλάξει ριζικά. Επίσης, διότι αν πιστεύετε ότι 100 ευρώ αγοράζουν τα ίδια σε μια περιοχή όπως αγορές 200 ευρώ σε άλλη περιφέρεια. Πώς μπορείτε να πείτε ότι μια περιφέρεια είναι δύο φορές πιο πλούσια από την άλλη, ενώ σε πραγματικούς όρους ε, είναι ίσες. Την περσμένη εβδομάδα στον Ηνωμένο Βασίλειο ετέθη το θέμα της απλούστευσης. Ε, είναι απογοητευμένοι πολλοί, εκτιμούν τη χρηματοδότηση που τους δίνεται, αλλά είναι πολύ περίπλοκη η, πρόσβασή τους και καμιά φορά η γραφειοκρατία τόσο μεγάλη που δεν καν ασχολούνται να πάρουν τα χρήματα. Και τίθενται πολλοί όροι που πολύ συχνά είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμμορφωθούν αυτοί που θέλουν τα χρήματα, που θέλουν τα χρήματα να πάρουν τα χρήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τρία ερωτήματα θα ήθελα να θέσω. Πρώτα απ' όλα, κύριε Πίτροπε, οι ε, συμφωνίες ε, ανάπτυξης ε, επενδύσεων με τα κράτη-μέλη υπάρχει αυτό το πράγμα ακόμα, γιατί δεν αναφέρεται στην αναφορά σε ό,τι αφορά τις αγορές. Ε, εμένεται σε αυτή τη θέση ή όχι. Δεύτερον, η θέση της Επιτροπής δεν είναι να κατηγορία αριστερά και δεξιά, αλλά θα εμβαθύνουμε την ανάλυση. Γιατί δηλαδή χώρες που, ε, στις οποίες έχουν χορηγηθεί δυσανάλογα ε, μεγάλα κονδύλια από το Ταμείο Συνοχής, τώρα βρίσκονται στη μεγαλύτερη κρίση, στη βαθύτερη κρίση και ζητούν ε, περαιτέρω βοήθεια και στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν θέλω να τις κατανομάσω γιατί τις γνωρίζετε. Και τέλος, ε, στην έκθεση στο σημείο 97, ο Επίτροπος λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει πιο θετικό πνεύμα για να καταλήξουμε σε αποτελέσματα, σε αυτά αποτελέσματα, αυτός είναι ο στόχος. Και εγώ συμφωνώ μαζί σας, θέλουμε αυτά αποτελέσματα. Επομένω, στο μέλλον, ποια θα είναι τα κριτήρια, όχι μόνο για τα ε, ποσοστά απορροφητικότητας, αλλά ποια θα είναι τα, ποσοστά, τα αποτελέσματα που θα, θα απαιτείται από τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή γιατί, για να αποφύγουμε έτσι τις ε, ε, τρέχουσες καταστάσεις. Ευχαριστούμε. Μαρή Τερέζ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Δεν έχω πολύ χρόνο, αλλά και πάλι θα πρέπει να αναφερθούμε σε αυτή την ε, εδαφική συνεργασία, γιατί ε, θα ψηφιστεί και η έκθεση της Επιτροπής Ρέτζε για τον στόχο 3 και θα ήθελα να υπερθυμίσω ότι περίπου 200 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες βρίσκονται σε αυτές τις διασυνοριακές περιφέρειες, δηλαδή 40% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, εν συντομία να υπερθυμίσω ότι ε, επιφέρει προς τη θέμενη αξία αυτή η εδαφική συνεργασία ήθελα να ε, ρωτήσω ποια είναι η θέση σας ό,τι αφορά τις ε, ανάγκες που αναφέρθηκαν στη συζήτηση για το μέλλον της εδαφικής συνεργασίας. Πρώτον, για τους ε, δημοσιονομικούς στόχους, γιατί υπάρχει ουσιαστική αύξηση του προϋπολογισμού του στόχου 3 και μάλιστα διπλασιασμός του προϋπολογισμού, ακόμα και αν ε, δεν αναφερόμαστε πάντα σε αυτό το τομέα. Υπάρχουν ζητήματα κατανομής ε, των κονδυλίων αναπρόγραμμα. Αυτό ενδεχομένως να αποτελεί ένα πρόγραμμα, ένα ε, κριτήριο. Μετά σε αυτά τα διευρωπαϊκά προγράμματα απαιτείται βεβαίως συνεργασία. Και μετά υπάρχει περιθώριο βελτίωσης σε ό,τι αφορά την απλούστευση της εφαρμογής αυτής της συνεργασίας. Ε, για το μέλλον του GOCT ε, βλέπουμε ότι αποτελεί σημαντικό εργαλείο, αλλά απαιτείται βελτίωση μετά για την προβολή αυτής της εταιρική συνεργασίας. Αναφέρθηκε ορισμένες εταιρικές σχέσεις. Επομένω, ποιο ρόλο θα λάβει ο στόχο 3 στην πολιτική συνέχεια στο μέλλον, ποια θα είναι η συνέχεια και μετά για τις μεταβατικέ περιφέρειες το συζητήσαμε εκτενώς, αλλά θέλω να τονίσω το εξή. Ε, θα ήθελα να στηρίξω αυτή την πρόταση ε, να υπάρχει δηλαδή μια ισορροπία, μια ισότητα ε, στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις διάφορες περιφέρειες. Ε, στην έκθεση Γκαριντό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στήριξε αυτή την πτυχή. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε έμφαση σε αυτό το τομέα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα είμαι πολύ σύντομο από πλευρά μου. Θα ήθελα σε αυτή τη φάση στην οποία βρισκόμαστε στη συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής και για ένα νέο πλαίσιο πολιετές χρηματοδότησης, θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν θέματα τα οποία άμεσα θίγουν τις υπερπεριφερειακές περιφέρειες. Είχατε μία φράση που σημείωσα με την οποία συμφωνώ απόλυτα και είπατε το εξής. Πρέπει να υπάρξει σαφής διαφοροποίηση μεταξύ δημοσιονομικών πτυχών και πολιτικών στόχων. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να επενδύσουμε στο μέλλον των περιφερειών, άσχετα από κονδύλια προπολογισμού. Σημείωσα αυτή τη φράση ένα λόγο πολύ απλό. Υπάρχει μεγάλη τάση και συνέβη και σήμερα σε αυτή τη συζήτηση να συγχαίουμε αυτές που είναι οι λιγότερο ευνοημένες περιοχές και να αναφέρεται το άρθρο 174 της συνθήκης με τις υπερπεριφερειακές περιφέρειες. Αυτή η τάση να διαχέουμε και να συγχέουμε αυτές τις περιφέρειες σε σχέση με θέματα των εκθέσεων που εξετάζουμε και την έκθεση Πίπερ για το μέλλον της πολιτικής συνοχής και αυτή η διαφοροποίηση που γίνεται, γίνεται για ένα απλό λόγο. Οι υπερπεριφερειακές ε, περιφερειε έχουν συγκεκριμένο άρθρο στη συνθήκη. Και έχοντας συγκεκριμένο άρθρο στη συνθήκη, αυτό γίνεται επειδή η πραγματικότητα των υπερπεριφερειακών περιοχών και περιφερειών δεν ήταν, είναι τόσο διαφορετική που απαιτεί διαφορετικού όρου προσέγγιση. Διαφορετικά δεν θα είχαμε ξεχωριστό άρθρο. Και πρέπει να γίνεται αυτή η διαφοροποίηση. Σε περίοδο δημοσιονομικής ε, λιτότητας δεν μπορούμε απλά και μόνο να αγνοούμε τα προβλήματα αυτά. Πρέπει να είμαστε πολύ συνετοί στη χρήση των δυνατοτήτων και των κονδυλίων. Όμως αυτές οι υπερπεριφερειακές περιφέρειες έχουν ένα άρθρο στη συνθήκη επειδή έχουν μια διαφορετική πραγματικότητα που πρέπει να αντιμετωπίζεται. Έχουν διαρκείς περιορισμούς ε, μειονεξίας, η απόσταση που τις χωρίζει η ε, απόσταση από τις αγορές, όλα αυτά συνεπάγονται ότι πρέπει να έχουν διαφοροποιημένη αντιμετώπιση. Η ερώτηση που θέλω να θέσω είναι, δεν θεωρείτε ότι το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το συγκεκριμένο ξεχωριστό άρθρο της συνθήκης και αυτό το καθεστώς διαφορετικών περιφερειών δεν θέτει εδώ κάποιους όρους για την χρήση των κονδυλίων και αν δεν υπάρχει αυτή η θετική, αν δεν υπήρχε αυτή η θετική διακριτική μεταχείριση υπέρ αυτών των περιφερειών θα τις ισοπεδώναμε. Η δεύτερη ερώτηση αφορά τα ποσοστά συγχρηματοδότησης θεωρείτε ότι μπορεί να διατηρηθεί το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης στο 50% από πλευράς μας για αυτές τις υπερπεριφερειακές περιοχές ή θεωρείτε ότι θα είναι δύσκολο να διατηρηθεί αυτό το ποσοστό χρηματοδότηση, συγχρηματοδότηση όπως ισχύει σήμερα. Ευχαριστώ. Äh, ε, Επίτροπο σε σχέση με την ερώτηση του Επιτρόπου Κέλλη αν και πότε όσο θα υπάρχει η ε, περιοχή περιφερειών συνοχής ναι θα πρέπει σε σχέση με αυτό το οποίο προαναφέρθηκε ότι κάποτε πιστεύω ότι πρέπει να αναλύσουμε όταν πραγματικά και αν υπάρξουν περιφέρειες που πιθανώς δεν εξελίσσονται περαιτέρω, λέω φαινομενικά πιθανώς δεν μεταξελίσσονται. Γιατί και οι περιοχές ανταγων, ε, ανταγωνισμού ε, μεταξελίσσονται. Είναι μια διαδικασία ρευστό, όπου η πρόκληση υφίσταται στο ότι οι υπανάπτυκτες περιφέρειες ταχύτερα κινητοποιούνται και ταχύτερα καλύπτουν την απόσταση που τις χωρίζει και προσεγγίζουν τους, ε, τον μέσο όρο. Και αυτό ιδιαίτερα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το κίνδυνο να υπάρξει πάλι απόσταση που θα χωρίζει κάποιες περιφέρειες από τον μέσο όρο. Δεν έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία, δεν έχουν φτάσει όλες ε, στο τέρμα και σε σχέση με την ε, κατάσταση αυτή βρίσκεται στην ευθύνη και της αρχής της επικουρικότητας και την παίρνουμε σα σοβαρά αυτή την αρχή της επικουρικότητας. Οι ίδιες οι περιφέρειες θα πρέπει να καθορίζουν και να διαφοροποιούν αυτό το οποίο προανέφερα μέσα στην ίδια την περιφέρειά τους ποιο είναι θεματολογικά ή περιφερειακά το χαρακτηριστικό στο οποίο θα θέλουν να επικεντρώνονται. Αλλά θα ήταν και από πλευράς μας ε, αν λέγαμε θα σας επιβάλλουμε το να κάνετε κάτι να πάτε ακόμα ένα βήμα πιο πέρα. Εδώ έχουμε κυρίαρχα δικαιώματα των πολιτικών που εμπλέκονται στην περιφερειακή πολιτική. Πρέπει να υπάρξει και διαφάνεια. Όμως δεν έχουμε δυνατότητα εμείς, ούτε και είναι και ευκταίο πολιτικά να επιβάλλουμε κάτι σε άλλους, ούτε και έχει νόημα διοργανωτικά να πάμε ένα βήμα ακόμα πιο πέρα και να το επιβάλλουμε. Το θέμα της απλούστευσης, το ακούω πάντα αυτό, αυτή την αναφορά. Μόνο πολύ λίγες εξειδικευμένες χειροπιαστές προτάσεις υποβάλλονται. Εκτός από το να μην υπάρχουν λέει τόσοι πολλοί έλεγχοι. Ε, με αυτό δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε να μην υπάρχουν πολλοί έλεγχοι. Και εδώ, σε σχέση με την σωστή ε, κατεύθυνση, οι ε, εκπρόσωποι ενός κράτους μέλους οι ευρωβουλευτές πρέπει να δουν το θέμα του National Declaration και να το παρακολουθήσουν με ζήλο αυτό το θέμα, διότι όταν υπάρχουν εδώ εθνικές δηλώσεις ή αν είχαμε τέτοιες εθνικές τοποθετήσεις, αυτό θα είχε συγκεκριμένες επιπτώσεις για τον όγκο των ελεγκτικών δράσεων όμως θα συνεισφέρουμε εμείς από πλευράς μας στην απλούστευση. Για παράδειγμα, όσον αφορά τις ε, συμβάσεις ε, και την σύναψη συμβάσεων. Έχουμε και την πράσινη βίβλο, το πράσινο βιβλίο. Πολλές προτάσεις αντανακλώνται για την περιφερειακή πολιτική στο πράσινο βιβλίο. Θα δούμε τι γίνεται με την παγίωση στο τέλος αυτής της διαδικασίας τι γίνεται και πώς αυτά αντανακλώνται σε εθνική νομοθεσία. Αναμένουμε όμως από πλευράς μας μια απλούστευση που θα ε, επέρθει για τον κύριο Γκορμάλης ε, για την, ε, τον όγκο επενδύσεων σωστό blaming and shaming, το να κατονομάζουμε και να δημιουργούμε ενοχές σε εκείνους που κατονομάζονται και δεν προσαρμόζονται, δεν ευθυγραμμίζονται. Ο προσανατολισμός θα πρέπει να είναι στη συνολική στοχοθέτηση σε σχέση με τη στρατηγική της Ευρώπης 2020 και με ποσοστοποίηση σε σχέση με αριθμητικά μεγέθη. Είναι καλό να έχουμε σαφή πλαίσια και στόχους που να μπορούν να μετρηθούν και να αξιολογηθούν οι επιδόσεις για να μπορούμε χωρίς αμφιβολίες και αμφισημίες να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα. Περιφερειακή συνεργασία της κυρίας Σάντσες Σμιτ. Πρώτον, σίγουρα και δεύτερον, κατά πόσον το 7% μπορεί να υλοποιηθεί ή όχι. Αυτή ήταν η αναφορά σας. Από την άλλη πλευρά και δεν θέλω να νομίσετε ότι προσπαθώ να υπεκφύγω, αλλά αν στον τομέα της μακροπεριφερειακής συνεργασίας τα πράγματα έστω και κατά προσέγγιση μπορούσαν να λειτουργήσουν όπως το φανταζόμαστε, ε, τότε θα είχαμε μια διασυνοριακή περιφερειακή συνεργασία στο τέλος τέλος. Αυτό που είναι τελικός μας στόχος, και συμφέρον μας διαπεριφερειακά όχι μόνο να συνεργάζονται αλλά και να υπάρχει και κατανομή επιμερισμός κονδυλίων ε, και αυτό θα ήταν δεδομένο και αν όλα αυτά τα συνυπολογίσουμε στο τελικό αποτέλεσμα τότε το μέτρο της χρηματοοικονομικής, ας το πω έτσι, αποτελεσματικότητας κατά τη διάρκεια των ετών σημαντικά αυξάνεται. Και τον Αύγουστο σύμφωνα με την εντολή μας θα έχουμε και την έκθεση που θα παρουσιαστεί για την εκμετάλλευση και χρήση και το performance της επιδόσεις όσον αφορά τις ε, περιφέρειες αυτές και θα καταλήξουμε σε συμπεράσματα που θα δοθούν. Για τον συνάδελφο Τεσέρα εμείς πάντα, όπως πάντα, γνωρίζουμε και συνειδητοποιούμε την προβληματική των uttermost regions, των υπερπεριφερειακών απομακρυσμένων νησιωτικών περιφερειών. Και κατά τη διάρκεια της εκπόνησης αυτών των στοιχείων σε εκθέσεις για την εσωτερική αγορά και τις επιπτώσεις στις αυτόνομες αυτές περιφέρειες, όπου εμείς ως Ρέγγιο καταβάλουμε προσπάθειες μέσα στο γύρο των αρμόδιων ευρωβουλευτών που παρακολουθούν τα θέματα πρέπει να πω ότι λαμβάνουμε υπόψη την πολυμορφοποίηση των οικονομικών υποδομών στις υπερπεριφερειακές περιφέρειες και πρέπει σε αυτό να επικεντρωνόμαστε και αυτό θα είναι ένα κέντρο βάρους στην μελλοντική μας ε, ε, προγραμματική περίοδο, στον προγραμματισμό των εργασιών μας για τη συγχρηματοδότηση υπάρχουν εσωτερικές ακόμα συζητήσεις που διεξάγονται, δεν θέλω να προδικάσω τίποτα, δεν το αρνούμε ότι γίνονται αυτές οι συζητήσεις. Πολλοί θεωρούν ότι η συγχρηματοδότηση θα έπρεπε να μειωθεί κάπως, να συρρυκνωθεί, ώστε να αυξηθεί το ποσοστό των συμμετοχής των ίδιων των εμπλεκομένων. Αλλά περνάμε δύσκολες ε, περιόδους, δύσκολη συγκυρία και είναι δύσκολο να βρεθεί η συγχρηματοδότηση ακόμα σε πιο χαμηλά επίπεδα για τις υπερπεριφερειακές περιοχές. Ίσως θα υπήρχε μια διέξοδος τουλάχιστον με ένα χρονικό περιορισμό μιας χρονικής περίοδου, κατά τη διάρκεια μιας δημοσιονομικής περίοδου να έχουμε ένα υψηλότερο ποσοστό που θα διασφαλίζεται ώστε να υπάρχει ένα μέσο ελαστικότητα στο οποίο θα διασφαλιστεί για να μπορεί να λειτουργήσει. Δεν θα είναι αναγκαίο, αναγκαστικό, δεν θα είναι αναγκαστικό να επεκτείνεται καθ' όλη τη διάρκεια της ε, χρηματοοικονομικής περίοδου. Μπορεί κάτι το 2017 να χρειαστεί να γίνει, ε, θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα με αυτόν τον τρόπο ότι η περιφερειακή πολιτική πρέπει να είναι σε θέση με τέτοιου είδους ε, δράσεις ελαστικά και ε, άμεσα να αντιδρά σε συγκεκριμένα δεδομένα. Η βασική ουσιώδης φιλοσοφία μας είναι ότι πρέπει να διατηρηθεί η συγχρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Thank you. Ε, <clears throat> <clears throat> e- Ευχαριστώ. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι αυτή η συζήτηση για το μέλλον της ε, πολιτικής συνοχής είναι μια ιδιαίτερη συζήτηση. Επιτύχατε, Επίτροπε Χάν, να μας χωρίσετε ε, σε, διαφόρα, σε διάφορα τμήματα και κατηγορίες όλους μας στο Κοινοβούλιο. Όλοι έχουν πάρει ε, διαφορετικές μεριές ε, και έτσι έχουμε έχουν ανάψει τα αίματα, αν θέλετε, για την συζήτηση σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό. Μπορείτε λοιπόν να διασκεδάσετε τις ανησυχίε μας και τις αμφιβολίες μας αυτή τη στιγμή, κύριε Χάν. Υπάρχουν λοιπόν ε, αυτά τα προβλήματα και οι διαφορέ μεταξύ των ε, ε, συναδέλφων. Ορισμένοι πιστεύουν ότι τα κονδύλια για αυτές τις περιφέρειες θα αντιληφθούν από το στόχο 2, ενώ άλλοι θεωρούν ότι θα αντιληφθούν από το στόχο 1. Έτσι κάποιοι θεωρούν ότι θα έχουμε περισσότερα χρήματα για, τα, για τις περιφέρειες ε, ε, του στόχου 1, αν δεν υπάρχουν ενδιάμεσες ε, περιφέρειες. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε ξεκάθαρα εδώ και τώρα πώς θα γίνει η κατανομή αυτών των ε, κονδυλίων και ποια θα είναι η πηγή της χρηματοδότησης. Σύντομα θα έχουμε την ψηφοφορία και περαιτέρω συζητήσεις στο Κοινοβούλιο. Επομένως, είτε θα ψηφίσουμε στην τύχη, γιατί δεν έχουμε πληροφορίες από εσάς, ή θα είμαστε σωστά πληροφορημένοι. Μιλάμε για περιφέρειες που θα, χρηματοδο... Ε, που θα λαμβάνουν χρηματοδότηση που κανονικά θα πρέπει να πάει σε άλλες περιφέρειες. Εγώ εκπροσωπώ την Πολωνία. Και θα ήθελα να ρωτήσω, υπάρχουν αυτές οι ενδιάμεσες ε, μεταβατικές ε, περιφέρειες και αν έτσι αυτό ισχύει, τότε εμεί θα έχουμε λιγότερα χρήματα στη διάθεσή μα. Ξέρω ότι τα απλουστεύω τα πράγματα, αλλά περί αυτού πρόκειται. Γιατί δημιουργούνται κάποιοι φόβοι ε, για το ποιο θα έχει να κερδίσει και ποιο να χάσει από αυτή την ιστορία. Ένα άλλο ερώτημα. Αναφέρθηκε από την Κόνσταντς ότι πολύ σύντομα τα κράτη-μέλη θα προτείνουν μειώσεις ε, του προπολογισμού και ο Επίτροπος Χάν ε, το ανέφερε και αυτό, αλλά θέλω να το επαναλάβω. Γιατί τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Εάν αντί να, να αυξήσουμε, μειώσουμε τον προπολογισμό στην πολιτική συνοχή, θα έχουμε οριζόντιες ή κάθετες μειώσεις θα προτείνετε να μειωθεί ο στόχος 2 και αυτό τον ενδιάμεσο στόχο ή θα προτείνετε και τη, μείωση του στόχου 1. Αυτό είναι σημαντικό γιατί ξέρουμε πώς ε, θα συνεχιστεί αυτή η συζήτηση για τον, για τον προπολογισμό. Θα χάσουμε όλοι δηλαδή ή οι πλουσιότερες χώρες. Ζητώ την γνώμη σας, Επίτροπε Χάν. Χρειαζόμαστε ξεκάθαρες πληροφορίες από εσάς. Και το τελευταίο ζήτημα για την τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα. Η κατάσταση αυτή επηρεάζει την πολιτική συνοχή στην Ελλάδα. Έχουμε λοιπόν ε, αυτά τα προβλήματα τα οικονομικά. Έχουμε προβλήματα και στην συγχρηματοδότηση από πλευράς Ελλάδας ιδιαίτερα σημαντικό το ζήτημα αυτό για την ε, μελλοντική συζήτηση του, ε, της πολιτικής συνοχής. Γιατί αρκετοί πολιτικοί θεωρούν ότι αυτοί που αποφελούνται περισσότερο από την πολιτική συνοχή είναι αυτοί που βρίσκονται στις, ε, που έχουν αντιμετωπίσει τα μεγαλύτερα προβλήματα. Έχουμε, δηλαδή, υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στα προβλήματα που αντιμετωπίζει μια χώρα και στην πολιτική συνοχή. Και χθε στι Βρυξέλλε κάποιο είπε ότι η Ελλάδα έχει πρόβλημα, αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω τη πολιτική Λισαβόνα. Σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα άλλο πρόβλημα έχω, αλλά χρειάζομαι γενικότερα και όχι τόσο στοχοθετημένα. Εδώ συζητάμε, λέμε, θα έπρεπε, πρέπει να, θα πρέπει αν γινόταν δυνητικά και διατυπώνουμε ιδανικές προτάσεις ε, που σε πολιτικά πεδία, σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να δεσμεύουν τις δράσεις μας. Όμως από διαφορετικούς συναδέφους ήδη προαναφέρθηκε, το επίπεδο μετάθεσης και λειτουργίας είναι τελείως διαφορετικό. Και όσον αφορά τη μετάθεση και εφαρμογή της πολιτικής συνοχής, έχουμε την αρμοδιότητα των κρατών μελών. Είχα την ευκαιρία πέρυσι και φέτος να συμμετάσχω σε διάφορες αποστολές της κοινοβουλευτικής μας επιτροπής. Τα ταξίδια μορφώνουν τον άνθρωπο. Αυτά τα οποία παρουσιάστηκαν όσον αφορά απλούστευση διοικητικών διαδικασιών, αναφέρθηκαν ως στοιχεία και από εμά και κοιτάξτε, προσέξτε, η κριτική στόχευε κυρίως στα ίδια τα κράτη-μέλη που με την υλοποίηση των δικών μας προγραμμάτων, των ευρωπαϊκών προγραμμάτων είναι υπεύθυνα και δημιουργούσαν δυσκολίες. Ή για εκεί όπου είναι αρμόδιες οι περιφέρειες, οι περιφέρειες ε, πρέπει να είναι υπεύθυνε. Η ιδανική μας λοιπόν στοχοθέτηση αντιμετωπίζει την πραγματικότητα επιτόπου με ομό τρόπο. Τι γίνεται. Δύο παραδείγματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο για τη διασυνορική συνεργασία, για παράδειγμα, ε, δημιούργησαν το μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Περιφερειακής Συνεργασίας. Εκεί πόλεις, περιφερειακά κέντρα, παράδειγμα Γερμανία, Πολωνία, θέλουν να συνεργαστούν με βάση ένα τέτοιο περιφερειακό σχέδιο διασυνοριακής συνεργασίας και να συντονίσουν τις δράσεις τους διασυνοριακά και να τις διαδικτυώσουν καλύτερα μεταξύ τους. Γερμανία και Πολωνία βρίσκουν μεγάλες αντιστάσεις στις περιφερειακές κυβερνήσεις στη Γερμανία, περιφερειακή κυβέρνηση του αρμόδιου κρατηδίου στη Γερμανία ή της κεντρικής κυβέρνησης στην Πολωνία. Από την άλλη πλευρά μας λένε ότι σε σχέση με περιφέρειες ε, περιοχής, ε, κατηγορία συνοχής έχουμε ανακοινώσεις και πληροφορίες επιχειρήσεων από τρίτες χώρες που εγκαταστάθηκαν σε αυτές τις περιφέρειες για υλοποίηση προγραμμάτων και τώρα απειλείται η ύπαρξή τους επειδή αναμένουν και καθυστερούν πληρωμές και απο, ε, μας αποστέλουν κραυγή βοήθειας. Έχουν ανάγκη να υποστηριχθούν. Κανένας δεν θέλει να αναλάβει δράση η κραυγή βοήθειας προέρχεται από αυτές τις επιχειρήσεις σε αυτές τις περιφέρειες και στρέφεται προς εμάς. Βοηθήστε μας, λένε. Κάτι πρέπει να γίνει. Όταν λοιπόν έχουμε την υλοποίηση πολιτικών συνοχής και δεν υπάρχει δημιουργία μεγαλύτερης, ε, περισσότερης Ευρώπης, αν υπάρχουν τέτοιες δυσκολίες, τότε επιτόπου με τις καλές μας προθέσεις δεν είναι δυνατόν να, να προχωρούμε παραπέρα. Δεν σημειώνεται τίποτα το θετικό και για την επόμενη περίοδο πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη. Αυτά τα πράγματα να μην τα αγνοήσουμε. Και όσον αφορά τη νέα διατύπωση δια, ε, κανονιστικών διατάξεων και ε, όρων και προϋποθέσεων να υπάρχει δυνατότητα μετάθεσης περισσότερων αρμοδιοτήτων στο ευρωπαϊκό επίπεδο να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Σέσκοντε Άντζελης παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, δύο ερωτήσεις στα γρήγορα. Πρώτη, είναι μία που αναφέρθηκε για πολλούς συναδέλφους. Διότι πάνω σε αυτό το σημείο διεξήχθη συζήτηση πάρα πολύ ζωηρή και αφορά αυτή την ενδιάμεση διάμεση κατηγορία, αυτό το θεσμό. Επ' αυτού θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η δεμή θα παραμείνουν περιθώρια βεβαιότητας, αμφιβολιών, σύγχυσης. Άρα χρειάζεται να αποσαφινιστεί. Ποια η σχέση μεταξύ πολιτικής του προϋπολογισμού από τη μια πλευρά και της δημιουργίας αυτού του, αυτής της νέας κατηγορίας. Από πού θα βρεθούν οι πόροι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι η δημιουργία νέας ενδιάμεσης ε, κατηγορίας δεν θα πρέπει να αφαιρέσει από τις υφιστάμενες κατηγορίες, να αφαιρέσει πόρους. Αυτό είναι σημαντικότατο. Θα πρέπει να διατεθούν συμπληρωματικοί πόροι ουσιαστικά. Λοιπόν, δεύτερο ερώτημα. Πιο πολλοί πόροι στις μικρές και μεσές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις. Ε, το έχω το θέμα αυτό στην καρδιά, με ενδιαφέρει πολύ όσον αφορά την έρευνα. Είναι πάρα πολύ σημαντικές για την πολιτική της καινοτομίας επίσης. Ε, έχω το εξή ερώτημα. Ποια μέτρα θα υθετηθούν για να δοθεί μια προώθηση στη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα προγράμματα καινοτομίας και έρευνας Δηλαδή, σωστικά, ποια μέτρα μπορώ να διευκολύνουν την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. Η πραγματική δυσκολία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, είναι η πρόσβαση σε αυτή τη χρηματοδότηση. Πολύ συχνά είναι πολύ δύσκολο, πάρα πολύ περίπλοκο. Και άρα τίθεται και το θέμα της απλούστευσης και της επιτάχυνσης ε, των διαφόρων διαδικασιών για την χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τρεμόπουλος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ε, θα ήθελα να αξιοποιήσω την παρουσία σας εδώ για να σας ρωτήσω κάτι εξαιρετικά επίκαιρο. Γνωρίζετε προφανώς ότι η Ελλάδα ε, έχει, βρίσκεται σε μια κρίση χρέους και ελλείμματος, κάτι που απειλεί με αποσταθεροποίηση ολόκληρη την Ευρωζώνη. Πρέπει να τιμωρηθεί ή πρέπει να υπάρξουν χρηματοδοτικές πολιτικές που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη, που εμείς λέμε φυσικά ότι πρέπει να είναι βιώσιμη. Σας άκουσα για τη συγχρηματοδότηση. Η ελληνική υποχρεωτική συμμετοχή στα ευρωπαϊκά προγράμματα όμως αυτή τη στιγμή είναι 22 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2013. Είναι προφανές ότι είναι αδύνατο να ανταποκριθεί. Αυτό είναι και ο λόγος που ο πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Γιούγκερ, δήλωσε προχτές στη βελγική εφημερίδα Libre Belgique ότι η Ελλάδα χρειάζεται μία ανάσα και πρότεινε τη χρηματοδότηση των ελληνικών προγραμμάτων από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία να γίνει κατά 100%. Δηλαδή χωρίς ελληνική συμμετοχή. Κατά τη γνώμη σας, είναι αυτό εφικτό, ώστε να μην επηρεάσει την υπόλοιπη περιφερειακή πολιτική. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε αυτή τη συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής συνόχης, Έχω τρία πράγματα που θέλω να πω. Πρώτα απ' όλα σε σχέση με το στόχο 3 που θα αφορά περίπου 150 χιλιόμετρα απόσταση και σε σχέση με το Κοινοβούλιο θα πρέπει να επανεξεταστεί αυτό το θέμα γιατί περιοχές όπως αυτή που εκπροσωπώ τα, ε, οι Βαλεαρίδες νήσι ε, δεν θα είχαν δυνατότητα να έχουν σωστή πρόσβαση. Για την ενδιάμεση κατηγορία θέλω να υπενθυμίσω αυτό το οποίο αναφέρθηκε εδώ, ότι το Κοινοβούλιο τοποθετήθηκε στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο με την έκθεση Γκαρίγα και στην Περιφερειακή Επιτροπή να μελετηθεί αυτή η κατηγορία ώστε να μην χάσει καμιά κατηγορία και να μπορούν όλοι να βρίσκονται σε πεδίο ισότιμο και δίκαιο και μια σκέψη σε σχέση με τις ε, ζώνες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, μειονεκτικές ε, περιοχές, ορεινές περιοχές. Ε, σε σχέση με αυτές δεν, έχουμε, δεν έχει η δική μου περιφέρεια σχέση ή με τις υπερπεριφερειακές περιοχές, αλλά ένα συγκεκριμένο άρθρο στη συνθήκη της Λισαβόνας για την αντιμετώπιση αυτών των περιοχών με μειονεξίες όπως στα νησιά. Και τέλος, πώς θα κατανεμηθούν τα κονδύλια. Υπάρχει ανησυχία να μην μείνει κανείς εκτός από την κατανεμηθή κατανομή. Θα είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσουμε σε αυτές τις δημοσιονομικές προοπτικές σε μια Ευρώπη με 27 κρατημέλη, με ΑΕΠ πολύ διαφορετικά μεταξύ της μιας χώρας και της άλλης και κανείς να μην παραμένει εκτός. Πώς θα είναι δυνατόν ώστε τα ταμεία αυτά να μπορέσουν να καλύψουν όλες τις ανάγκες. Με ποιο τρόπο θα κατανεμηθούν τα κονδύλια και πολλές φορές διεξάγονται περιττές συζητήσει και χάνουμε πολύ χρόνο. Θα ήταν καλό να ξέραμε τι υπάρχει, με ποιο τρόπο θα προταθούν κάποια πράγματα και έτσι να λαμβάνουμε υπόψη την σύνθεση αυτών των περιφερειών χωρίς να χάνουμε χρόνο σε συζητήσεις, χωρίς να έχουμε συγκεκριμένα χειροπιαστά στοιχεία. Αν είχαμε στοιχεία, αν έχουμε στοιχεία είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί. Χάνουμε και χρόνο χωρίς στοιχεία περνάμε πολύ χρόνο κάνοντας λόγο για το ίδιο θέμα τα, με τις ίδιες παρεμβάσεις αλλά με φήμες που κυκλοφορούν λόγω φημολογίας χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Παρακαλώ Επίτροπε έχετε τον λόγο να απαντήσετε. Αξιότιμη Ευρωβουλευτά, κατανοώ την ανησυχία σας και την ανυπομονησία σας. Καλύπτεται και με τη δική μου ανυπομονησία, διότι στην τελική αξιολόγηση από αυτά θα εξαρτηθεί τι θα γίνει με τον προϋπολογισμό και γι' αυτό δεν μπορώ να σας δώσω αριθμητικά στοιχεία για κονδύλια και προϋπολογισμούς. Μπορώ να σας πω ποιες είναι οι προσεγγίσεις, οι σκέψεις και τα επιχειρήματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έρχομαι στην παρέμβαση του κυρίου Όλμπριχτ. Έχουμε ένα σύστημα, ένα πρότυπο πώς κατανέμονται τα κονδύλια σήμερα. Και αυτό το πάνω κάτω έχει το εξής, περίπου 51% πάνε στους ε, αποδέκτες και έχουμε την αναλογία αυτή μισό-μισό έστω μεταξύ ε, των, ε, ε, αυτών που καταβάλουν τα κονδύλια και σε σχέση με τους αποδέκτες. Και για την αναλογία θα πρέπει για πολιτικούς λόγους να υπάρχουν κάποια κριτήρια που θα λαμβάνονται υπόψη για τη μελλοντική δομή του προϋπολογισμού και να μην έχουμε μετάθεση από τη μία μέρα στην άλλη. Να υπάρχει μια αντιστάθμιση, ένας, μια εξισορρόπηση μεταξύ των καθαρών εισφορέων και των καθαρών αποδεκτών που εποφελούνται. Και γι' αυτό θα πρέπει να γυρίζουμε διαφορετικές ε, βίδες ή κάνουλες, να ρυθμίζουμε λεπτά με το σωστό τρόπο τα στοιχεία αυτά και αν στην επόμενη περίοδο θα έχουμε λιγότερες περιφέρειες ε, ε, συνοχής, ανάλογα θα προσθεθούν κάποιες άλλες ε, σε άλλη κατηγορία αν δεν αλλάζαμε τίποτα στο όλο σύστημα συνολικά, τότε η κατανομή των κονδυλίων δεν θα έβαινε καλώς. Θα είχαμε 65-35% αναλογία και αυτό δεν θα ήταν δίκαιο. Γι' αυτό πρέπει να προβληματιστούμε, να δούμε πώς μπορούμε πάλι να εξισορροπήσουμε τα πράγματα και να έχουμε μια σωστή ισορροπία στην κατανομή των κονδυλίων. Αυτή τη στοχοθέτηση ακολουθούμε, άσχετα από τα απόλυτα μεγέθη που στο τέλος τέλος θα έχουμε ως έκβαση. Διότι στόχος πρέπει να είναι να μην υπάρχουν ακραία εκείνοι που θα κερδίζουν υπερβολικά και ακραία εκείνοι που θα χάνουν υπερβολικά. Πρέπει να υπάρχει μια εξισορρόπηση και να είναι δίκαια τα πράγματα. Και αν ο προϋπολογισμός ε, θα είναι ε, εξίσου μεγάλος σε απόλυτα αριθμητικά μεγέθη, θα υπάρχουν κάποιες χώρες που σε απόλυτα μεγέθη θα αυξήσουν και κάποιες θα υπάρξουν που θα μειώσουν, θα μειωθούν τα κονδύλια για αυτές, διότι υπάρχουν εξελίξεις σε κάποιες χώρες. Τα πράγματα μετεξελίσσονται. Ξέρουμε ότι και η ίδια η Ισπανία, στην Ισπανία όσον αφορά την εξέλιξη των περιφερειών, είναι μια ιστορία μεγάλων επιτυχιών. Θα υπάρχει κάποια περιφέρεια που θα είναι περιφέρεια συνοχής. Πρέπει αυτό στην κατανομή των κονδυλίων να λαμβάνεται υπόψη και να εκφράζεται, να αντανακλάται διότι στα κράτη-μέλη σχεδόν όλες οι πρωτεύουσε των κρατών μελών δεν θα είναι πια περιφέρειες συνοχής. Αλλάζουν λοιπόν τα πράγματα. Κύριος στόχος όμως είναι να διασφαλιστεί μια ισορροπία στην κατανομή των κονδυλίων συνολικά πανευρωπαϊκά αλλά και μεταξύ των περιφερειών. Γι' αυτό είναι ανάγκη να ρυθμίσουμε με τέτοιο τρόπο την ροή των κονδυλίων ώστε να υπάρχει αυτή η ισορροπία και όταν υπάρχουν ε, ε, αλλαγές να έχουμε την μεταβατική κατηγορία προσωρινή ε, κατηγορία των προσωρινών περιφερειών ή μεταβατικών περιφερειών ώστε να λαμβάνονται υπόψη αυτές οι ενρευστό αλλαγές και να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες τους. Δεν μπορώ να σας δώσω αριθμητικά στοιχεία, δεν τα έχω ο ίδιος για να σας τα δώσω. Μπορώ όμως να σας επεξηγήσω την θεμελιώδη προσέγγιση ως θέμα ουσιώδες, θέμα αρχής, πώς το προσεγγίζουμε εμείς για να το αντιμετωπίσουμε. Ελλάδα τώρα. Ελλάδα. Μάλιστα είχαμε προβλήματα απορροφητικότητα σε σχέση με την Ελλάδα. Ιδιαίτερα επειδή τα διατεθέντα κονδύλια όσον αφορά και την ιδιωτική οικονομία αυτή τη στιγμή δεν δεν χρησιμοποιούνται. Προφανώς το κλίμα της αβεβαιότητας και ανασφάλειας είναι τόσο μεγάλο στην Ελλάδα που υπάρχει ιδιαίτερη επιφύλαξη, επιφυλακτικότητα. Δεν θα καταφέρουμε να το απαρακάμψουμε, να το αποφύγουμε, να κάτσουμε κάτω με κάθε επιμέρους περιφέρεια και να συζητήσουμε σε βάθος τι συμβαίνει, τι μπορεί να οδηγήσει σε μια βελτίωση και διεύρυνση της βάσης στην επιμέρους περιφέρεια μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Πρέπει να το κάνουμε αυτό, να δούμε σε σχέση για παράδειγμα και με την όχι μόνο γεωργία και τουρισμό αλλά κάθε περιφέρεια έχει τις δικές της ιδιομορφίες και ανάγκες. Θα πρέπει να τα αναλύσουμε όλα αυτά για παράδειγμα cluster building, ε, κατηγοριοποίηση και ομαδοποίηση, εξειδίκευση, ε, specialization. Δεν θα ε, πρέπει να αμελήσουμε αυτό το έργο και για την Ελλάδα, πρέπει να το δούμε. Και σε σχέση με την άλλη παρατήρηση, αυτό που είπατε, είναι και σωστό, αλλά μπορεί να μην είναι και σωστό. Σε σχέση με την συγχρηματοδότηση και σε ποιο ποσοστό θα ανάγεται. Διότι αν πιστεύει κανείς ε, στη σκέψη ότι πρέπει να ε, υπάρχει συμμετοχή από πλευράς των ενδιαφερομένων δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτό το γεγονός. Αν αυξηθεί το ποσοστό συγχρηματοδότησης, τότε φυσικά η δυνατότητα της δημιουργίας περισσότερων προγραμμάτων μειώνεται με την αύξηση των κονδυλίων που δίνονται και σε σχέση με την Ελλάδα η δυνατότητα να αυξηθεί η συγχρηματοδότηση μέχρι μέγιστο 85% κατά τη διάρκεια της ε, τρέχουσας ε, περίοδου θα πρέπει να ε, εξεταστεί ξεχωριστά. Το άλλο το ανέφερα για τον συνάδελφο Τσέλερ. Προσέξτε, οι δικές μας, τα δικά μας αιτήματα, η ιδανικά και η πραγματικότητα που διήστανται θα πρέπει να καταλάβουμε το τι γίνεται. Δεν είναι δυνατόν ένα προς ένα να είναι η αναλογία υλοποίηση των πολιτικών μας. Η πολιτική μας πρέπει να μπορεί να ασκεί την αναγκαία πίεση ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί στο μέτρο του εφικτού. Και στη διασυνοριακή συνεργασία βλέπουμε προόδους. Το ανέφερα όμως και σε άλλο σημείο στην παρέμβασή μου. Τα κράτη-μέλη τα ίδια δεν είναι πολλές φορές τόσο ικανοποιημένα για αυτή την, από αυτή την διασυνοριακή συνεργασία. Αληθεύει αυτό. Αλλά βήμα προς βήμα πρέπει να δούμε την υλοποίηση των δράσεων ώστε στο τέλος τέλος οι εθνικά υπεύθυνοι στα κράτη-μέλη να μην κλείνουν τα μάτια και να μπορούν και εκείνοι να συμπορεύονται. Τώρα, ο κομβικός ρόλος ε, για τις ε, καινοτομίες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την έρευνα είναι πολύ σημαντικό να δούμε την προαγωγή, την προώθηση της έρευνας. Είναι αποφασιστική σημασίας πώς τα κονδύλια για την έρευνα κατανέμονται. Είναι η εξαιρετική αποδοτικότητα, οι καλύτερες επιδόσεις, excellence, η αρχή που είναι η πιο σημαντική. Στην αρχή της περιφερειακής πολιτικής υπάρχει και η αρχή των περιφερειακών ε, κριτηρίων επιδόσεων σε τεχνολογική επίδοση, στην, στο marketing, στο διοικητικό επίπεδο, να βελτιωθεί αυτό το δυναμικό των περιφερειών. Όλα αυτά τα βλέπω ως καινοτομία συνολικά. Γι' αυτό είναι σημαντικό στην μελλοντική ε, περιφερειακή πολιτική τομεακά να ληφθούν υπόψη αυτά και να έχουμε κονδύλια για την υποστήριξή τους. Ειλικρινά, συνάδελφε Τρεμόπουλε, για να ολοκληρώσω είμαι πάντα επιφυλακτικός για μεθόδους κυρώσεων και προστήμων. Ελπίζω ότι το θέμα δεν θα τεθεί ποτέ και δεν θα πρέπει ποτέ να ληφθεί η μία ή η άλλη απόφαση. Ας το πω έτσι, υπάρχει η παρακολούθηση αυτών των τάσεων από τους hardliners, τους σκληροπολιτικούς όταν κάποια χώρα παραβιάζει κάτι. Δεν θέλω να δώσω συνέχεια σε αυτό. Υπάρχει σοβαρή αντιμετώπιση με τα υπέρ, τα κατά σε σχέση με μια κυβέρνηση ή την αντιπολίτευση. Αν τώρα μια χώρα τα όσα επιβάλλει ή ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αγνοεί και τα παραβιάζει είναι ίσως πολύ σκληρό να τοποθετηθώ έτσι είναι μια θεωρητική συζήτηση δεν θα ήθελα να επισέλθω σε αυτήν και για το αν θα υπάρξουν εκλογές ή αλλαγές με τέτοιο τρόπο ώστε στον τομέα της Μεσογείου να υπάρξει μια δυνατότητα συνεργασίας. Αυτό θα το δούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε συνάδελφοι και ευχαριστούμε και τον κύριο Επίτροπο για τη συμμετοχή σε αυτή τη συζήτηση. Κύριε Πετρόπα, ελπίζουμε να σας δούμε και αυτήν την εβδομάδα κατά τη διάρκεια της Ολομέλης. Ελπίζω να παραστείτε, γιατί θα υπάρξει εκτενή συζήτηση με αρκετέ εκθέσεις που δείχνει ότι η Επιτροπή προετοιμάζεται για την περίοδο διαπραγματεύσεων. Και προσδοκούμε να έχουμε τους κανονισμούς των συντομότερο δυνατόν. Ξέρετε ότι, ξέρουμε ότι υπάρχουν και ε, κανόνες στο ιστορικό της Επιτροπής που το αποφασίζουν. Ευχαριστούμε και πάλι. Ας περάσουμε στην ε, έκθεση Herman Winkler. Περνάμε, συνάδελφοι, στο επόμενο σημείο της μέσης διάταξης. Έχουμε μισή ώρα στη διάθεσή μας για δύο ζητήματα. Πρώτον, έχουμε το σχέδιο γνωμοδότησης ε, του Χέρμαν Βίνκλερ για την πράσινη βίβλο για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας. Ας συνεχίσουμε, συνάδελφοι να δώσω πρώτα το λόγο στον συντάκτη της νομοδότησης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, μόλις πιο πριν στο προηγούμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης το ακούσαμε. Το μέλλον της χρηματοδότησης για την έρευνα, όχι μόνο υπό το πρίσμα της Επιτροπής Ενέργειας, ε, με συγχωρείτε, ε, ε, είναι σημαντικό, αλλά αν δούμε και τους αριθμούς, στα αρχικά χρόνια ήταν 5% και σε σχέση με τις επενδύσεις που έγιναν έναντι της ε, πολιτικής ε, για την ε, καινοτομία. Σήμερα μετά από 10 είναι 25% δηλαδή για την τρέχουσα περίοδο κάνουμε λόγο για 86 δισεκατομμύρια ευρώ που θα έχουμε σε διάθεση για την καινοτομία, την έρευνα, για τις επιχειρήσεις και αυτό είναι παραπάνω από το πρόγραμμα έρευνας, το 7ο πρόγραμμα δράσης. Το ξέρουμε αυτό και υπάρχουν μεγάλες διαφορές όμως στις περιφέρειες όσον αφορά το δυναμικό και τις ικανότητες για την ε, ε, καινοτομία. Και πρέπει να σκεφτούμε εμείς ποιες ε, συστάσεις θα δώσουμε στην Επιτροπή Βιομηχανίας Πολλά έχει εξετάσει η Επιτροπή Βιομηχανίας και ελπίζω με τη δική σας συμμετοχή να καταλήξουμε με σαφή τοποθέτηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης να δώσουμε έτσι ένα σαφές μήνυμα στην Ολομέλεια για το τι πρέπει να γίνει. Αγαπητοί συνάδελφοι, να πω δύο λόγια διαδικαστικά. Αφενός γνωρίζετε ότι εμείς είμαστε για το ε, σχέδιο ε, γνωμοδότησης ε, θα καταθέσω και ο ίδιος κάποιες τροπολογίες, θα υπησέρθω σε αυτό και δεύτερον Έχουμε ένα πρόβλημα χρονικό. Δεν οφείλεται όμως σε δική μας καθυστέρηση, αλλά στο χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής Βιομηχανίας. Γνωρίζετε ότι αύριο 18.00 εκπνέει η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Γνωρίζω ότι πολλοί έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα και έχουν ε, προβεί σε ανταλλαγή απόψεων, ώστε όλοι πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε να διατυπώσουμε τα αιτήματά μας έγκαιρα. Επί της ουσίας πέντε σημεία θα ήθελα να αναφέρω. Πρώτον, θα ήθελα μια σαφής τοποθέτηση να υπάρξει υπέρ της υποστήριξης για την καινοτομία μέσω της πολιτικής συνοχής. Επίκαιρα ανταποκρίνεται αυτό σε σχέση με τις κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική συνοχή. Υπογραμμίζει και τη σημασία της περιφερειακής υποστήριξης για την έρευνα και την καινοτομία υπέρ των ε, μελλοντικών ε, προγραμμάτων. Καμία αποδυνάμωση δεν θέλουμε να γίνει δεκτή. Το αντίθετο, πιστεύουμε ότι το θέμα της καινοτομία είναι μια αναγκαστική προτεραιότητα για τις περιφέρειές μας και πρέπει να αντανακλάται στα κονδύλια που δημοσιονομικά διαθέτουμε. Αυτή η αναγκαία προτεραιότητα πρέπει να έχει τέτοιο εύρος, τέτοιο φάσμα, ώστε άλλες ε, προτεραιότητες, για παράδειγμα τα θέματα που αφορούν την ενεργειακή αποδοτικότητα ή ε, άλλα θέματα να εντάσσονται μέσα στα πλαίσια αυτά. Ποια κονδύλια θα πρέπει να διατεθούν για τη χρηματοδότηση. Κέντρο βάρους της υποστήριξης θα πρέπει να είναι η βέλτιστη αποδοτικότητα excellence. Αυτό το αναφέραμε και πιο πριν. Όμως ε, η προσέγγιση σε αυτό το φάσμα εντάσσει και την καινοτομία και την υποστήριξη της καινοτομίας στην περιφερειακή πολιτική. Μια περιφερειακή πολιτική στο αναγκαίο εύρος με την ενδυνάμωση της περιφερειακής συνιστώσας παντού. Καινοτομία που για όλες τις περιφέρειες είναι αποφασιστική σημασίας. Δυστυχώς εξακολουθούν και υπάρχουν πολλές και μεγάλες διαφορές μεταξύ των περιφερειών. Εδώ πρέπει να εξισώσουμε τα πράγματα. Είναι καθήκον μας. Και ζητούν και περιφέρειες κονδύλια να διατεθούν μέσα στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών ε, για την ε, πολιτική αυτή που δεν έχουν διατεθεί επαρκώς μέχρι σήμερα και πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις. Τώρα, αν ο στόχο θα είναι περιφερειακή βέλτιστη αποδοτικότητα, excellence, υποστήριξη του δυναμικού, ώστε η έρευνα και το δυναμικό και η καινοτομία να ενισχύονται, ώστε μελλοντικά και περισσότερες επιχειρήσεις να μπορούν να συμμετάσχουν σε τέτοια καινοτόμα προγράμματα για την έρευνα. Κάνουμε λόγο για την βέλτιστη αποδοτικότητα, excellence όπω προανέφερα, και για την δυνατότητα συγχρηματοδότηση και από τα διαθροτικά ταμεία ή αν κάποιε περιφέρειες θα έχουν ένα ευρύτερο, μια ευρύτερη έννοια σε σχέση με την καινοτομία και τις δράσεις μας. Σε πάση περιπτώσει όμως στην περιφερική πολιτική πρέπει να επικεντρωνόμαστε στους κυριότερους στόχους της πολιτικής συνοχής. Δέσμευση ε, κονδυλίων για την κάλυψη των διαθροτικών ε, χασμάτων και διαφορών. Προαγωγή της περιφερικής οικονομίας, προαγωγή έρευνας ε, και καινοτομίας. Έρχομαι στο τρίτο σημείο εξειδίκευση, ευφυής εξειδίκευση. Από το σχέδιό μου μπορείτε να δείτε ότι θεωρώ αυτό το σημείο ουσιοδέστατο, σπουδαιότατο, πώς η τεχνολογική ανάπτυξη μπορεί να συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη και μάλιστα στην περιφερειακή πολιτική με την εξειδίκευση, την ευφυή εξειδίκευση. Έχει μεγάλη σπουδαιότητα αυτό το θέμα. Οι περιφέρειες πρέπει εντάσσοντας ε, τους εμπλεκόμενους ε, σε αυτή την ανάπτυξη, τις επιχειρήσεις και την έρευνα να έχουν μια κομμένη και ραμμένη στα μέτρα τους πολιτική για την έρευνα και την καινοτομία αναλαμβάνοντας πάντα δράσεις, έχοντας αναλύσει προηγούμενα τα ευάλωτα τροτά σημεία τους και τα δυνατά χαρτιά τους, ώστε να μπορούν μέσα από αυτό το νέο πλαίσιο για την έρευνα και καινοτομία να αποκομίσουν τα μέγιστα ωφέλη κατά την ε, διάθεση των κονδυλίων. Επίσης, ενδυνάμωση. Πρέπει εδώ η ενδυνάμωση, η ενίσχυση να είναι όρος κλειδί και να μην έχουμε την αρχή του ποτιστηριού της κάνουλας που θα ισχύει. Άλλα σημεία ε, στήριξης στα λειτουργικά προγράμματα πρέπει πάντα να αντανακλώνται όπως είναι το σωστό. Ευφυής εξειδίκευση. Συνάδελφοι, αυτό πρέπει να βοηθήσει την διεθνή ανταγωνιστικότητα να προαγάγουμε και μάλιστα μέσα από την ομαδοποίηση επιχειρήσεων και πρωτοβουλειών στο clustering και παραδοσιακή τομής όπως ε, η βιοτεχνία, ε, το χειροτεχνικό τμήμα, η γεωργία να μπορούν στο μέλλον για την καινοτομία ενισχυμένα να καλύπτονται. Θα έλεγα ότι μια προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και που αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται σε μια πλατφόρμα ε, που θα μπορούσε να ε, δημιουργηθεί για να βοηθήσει ώστε να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών και να υπάρχει και η προσέγγιση της επικοινωνίας των διαφορετικών επιπέδων μεταξύ τους σε σχέση με αυτή την πλατφόρμα περνάω στο τέταρτο σημείο που είναι κάτι πολύ σπουδαίο και σημαντικό για μένα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό που αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η συμμετοχή στο πρόγραμμα έρευνας μπορεί να επεκταθεί και να ενδυναμωθεί. Συμφωνούμε σε αυτό. Δεν είναι πολλές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που να μπορούν να επενδύσουν στην έρευνά τους πολλά κονδύλια όπως το, τα Eurostars ή άλλες πρωτοβουλίες. Όμως, παρόλα αυτά, είναι καινοτόμες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το βλέπουμε αυτό. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραδοσιακής εμβέλειας που εργάζονται πολύ στενά παρακολουθώντας τις ανάγκες, καλύπτοντας τις ανάγκες των πελατών τους και έτσι συνδέουν τις περιφέρειες ε, με τους πελάτες και είναι χρήσιμες για αυτήν την πολιτική στις περιφέρειες ε, με την προσφορά εφικτών όρων, με εφικτές προϋποθέσεις και όρους ε, στην υποστήριξή τους για την μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας και ε, τομέα ανάπτυξης είναι κάτι θετικό. Επίσης, ε, για την ίδρυση πολλά υποσχόμενων επιχειρήσεων, το θέμα της ε, διαδικτύωσης και των δικτύων, δημιουργίας δικτύων μεταξύ αυτών των επιχειρήσεων. Μπορούν τα διαθροτικά ταμεία να συνεισφέρουν με την προσφορά τους για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να επεκτείνουν την προσφορά τους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εδώ θα πρέπει να μην έχουμε ε, συγχώνευση μεταξύ του ενός και του άλλου ε, προγράμματος ή περιορισμό ε, εύρους ή φάσματος ε, δυνατοτήτων. Είναι μεγάλη σημασία οι δράσεις αυτές και εδώ θα έπρεπε να δράσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε η προσφορά και οι δυνατότητες να διευρυνθούν και να διασφαλιστούν. Πέμπτον, διεθνή συνεργασία για, παράλληλα με, την, με το αίτημα της ε, προώθησης της, ε, των βέλτιστων επιδόσεων για την περιφερειακή πολιτική θα πρέπει να διασφαλίσουμε και την προοπτική της διαπεριφερειακής συνεργασίας. Με την διαπεριφερειακή συνεργασία οι περιφερειακοί εταίροι μπορούν να προωθηθούν στην ε, δικτύωση μέσω clusters, μέσω ομάδων επιχειρήσεων και έτσι θα μπορούσαμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Τέλος, θέλω να αναφέρω κάτι για τα μέσα χρηματοδότησης και για τους ε, κανόνες από πλευράς διοικητικής ε, τάξης για τα μέσα χρηματοδότησης όπως τα ανακυκλούμενα ή ε, σε ανακύκλωση κονδύλια θα πρέπει να καθορίσουμε κομβικά σημεία ώστε να υπάρχει δυνατότητα συνδυασμού μέσω κονδυλίων διαθωτικών ταμείων να μην υπάρχει ε, μόνο αυτή η προοπτική αλλά να υπάρχει και η δυνατότητα επέκτασης ώστε στα θέματα χρηματο, ε, χρηματοοικονομικών δράσεων να μπορεί να υπάρχει επέκταση στις υποδομές. Διασταυρούμενη χρηματοδότηση είναι κάτι το οποίο είναι σκόπιμο ώστε συνέργεια να διασφαλίζεται για την υποστήριξη προγραμμάτων για την έρευνα και την καινοτομία αφετέρου. Κατά τα άλλα, κάθε απλούστευση των διοικητικών ή κανόνων για τις διοικητικές ε, ε, διεργασίες είναι κάτι θετικό. Και σε σχέση και με μια κεντρική διαχείριση σε σχέση με το ΣΕΙΠΕ ή και την αποκεντρωμένη ακόμα προσέγγιση από πλευράς μας, παρόλα αυτά θεωρώ την αναγκαίοι κανόνες. Κανόνες και διατάξεις και ποσοστώσεις όσον αφορά τις διατάξεις για την υποστήριξη και αποκοπήν ποσά που πρέπει να εναρμονιστούν σε ένα ενιαίο πλαίσιο στο μέτρο του εφικτού ώστε στα χρονοδιαγράμματα και στη δυνατότητα δράσης να έχουμε απλούστερες διατάξεις για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτά είναι οι προτάσεις μου για την έκθεσή μου. Προσβλέπω στη συζήτηση επ' αυτών και ελπίζω ότι με τροπολογίες και με συμβιβαστικές τροπολογίες θα καταφέρουμε η παρέμβασή μας στην περιφερειακή κοινωνική πολιτική να διασφαλιστεί και να βελτιωθεί. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε στους σκιώτες. Η Μαρία Πέρες. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι είναι έξοχη η δουλειά. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόταση που μας παρουσιάζεται σήμερα. Και είναι, θα ήθελα να αναφερθώ και μάλλον περιλαμβάνει τα πιο σημαντικά στοιχεία. Συμφωνώ ότι είναι σημαντικό να υπάρχει καλύτερο συντονισμό μεταξύ περιφερειακή πολιτική και των κοινών στατικικών που ακολουθούμε για την έρευνα και την καινοτομία. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι αυτός ο συντονισμό θα πρέπει να περνά μεγαλύτερη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην σύλληψη και διαμόρφωση αυτών των πολιτικών. Θα πρέπει προτεραιότητες να καθοριστούν, ε, συναρτήσει των ιδιαιτεροτήτων της κάθε περιφέρειας. Δεύτερον, ε, συμμερίζομαι την αύξηση της ε, συμμετοχής των μικρομεσών επιχειρήσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων για την καινοτομία, διότι είναι οι βασικές πηγές απασχόλησης οι μικρομεσές επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Συμμερίζομαι λοιπόν από το στόχο να υποστηρίξουμε τις μικρομεσές επιχειρήσεις, την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και να μειωθεί το γραφειοκρατικό άχθος που τις πλήττει. Ε, θα ε, συμφωνώ με τον εισηγητή στο τρίτο σημείο θα πρέπει οι περιφέρειες να αναπτύξουν ειδικέ στρατηγικές καινοτομία με ευφυείς ε, εξειδικεύσεις είναι σημαντική έννοια αυτή θα πρέπει να επιμείνουμε το συντονισμό που πρέπει να υπάρξει μεταξύ των εθνωτικών ταμείων, των ταμείων συνοχής, των πόρων συνοχής και των μέτρων για την καινοτομία και το γενικό, για το γενικό πλαίσιο το δημοσιονομικό θα πρέπει να βελτιστοποιήσουμε τις χρηματοδοτήσεις. Θα πρέπει να θαρρύνουμε τη διεθνή χρηματοδότηση να ε, συμμετάσχουν οι εθνικοί και περιφερειακοί φορείς όσον αφορά την κατάρτιση ενός στατηγικού προγράμματος, όσον αφορά την έρευνα και την καινοτομία ε, και να συντονιστεί αυτή η προσπάθεια με τις προσπάθειες που καταβάλλονται στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και τέλος, το έγγραφο χρειάζεται μια αναφορά στο ρόλο βιώσιμης ανάπτυξης των πόλεων, αστικής ανάπτυξης, που θα βασίζεται στην καλή ζωή του, του πληθυσμού και στην βιωσιμότητα, την κοινωνική και την περιβαλλοντική χωρίς να ξεχνάμε και την ενέργεια. Δεν θα πρέπει να υπάρχει αύξηση μεγάλη του κόστους περιβαλλοντικού. Ευχαριστώ εκ νέου τον εισηγητή για την έξοχη δουλειά που έκανε. Και θα παρουσιάσω κάποιες τροπολογίες εν ονόματι της ομάδας μου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Πραγματικά είναι ένα εξαιρετικό έγγραφο αυτό της έκθεσης αυτής και αφορά ιδιαίτερα την συνεργασία υπέρ έρευνας και καινοτομίας. Τούτων λεχθέντων κάποιες παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω, να προσθέσω μάλλον η Σκιώδη εισηγήτρια είπε ότι χρειαζόμαστε ένα καλύτερο συντονισμό. Έχουμε το πρόγραμμα πλαίσιο, έχουμε όμως και την ανάγκη να υπάρχει διασύνδεση και αναφορά με τα διαθροτικά ταμεία. Και υπάρχει μια διαφορά εδώ σε σχέση με αυτά που αναφέρονται στο πρόγραμμα πλαίσιο και μπορούν να χρηματοδοτηθούν και αφορά τεχνολογία εχμής αυτή η πτυχή και έχουμε και τα διαθεωτικά ταμεία και κονδύλια όπου η πρακτική εφαρμογή, η καινοτομία ε, καλύπτεται με ε, τρόπο χειροπιαστό έχουμε ένα μεγάλο μέρος ε, της καινοτομίας που απορρέει και πηγάζει στην Ευρώπη και που καλύπτεται έτσι. Πρέπει όμως να υποστηρίξουμε και έρευνα που οδηγεί στην καινοτομία και που οι επιχειρήσεις που ε, εργάζονται σε αυτόν τον τομέα να πρέπει να μπορούν να δράσουν με τέτοιο τρόπο ώστε η καινοτομία να αυξηθεί και να δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης. Με άλλα λόγια, χρειαζόμαστε δηλαδή τη συνεργασία με αυτές τις επιχειρήσεις. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε αυτό και να διασφαλίσουμε αυτή την πτυχή. Διότι είναι δεδομένο το ενδιαφέρον και συμφέρον των επιχειρήσεων να συμμετάσχουν σε αυτή τη δράση. Και στον τομέα της έρευνας λοιπόν πρέπει να εντάσσεται αυτή η προσπάθεια στην στοχοθέτηση που ε, καταρτίζουμε. Και εδώ αρκετά μπορούμε να πετύχουμε. Και πρέπει, πρέπει επίσης να μας προβληματίσει πώς θα μπορούσαμε την καινοτομία αυτή να την διοχετεύσουμε στην αγορά. Να αποτελέσει αντικείμενο, ας το πω έτσι, εμπορική εκμετάλλευσης. Σίγουρα πολλά μπορούν να βελτιωθούν στην Ευρώπη. Αυτέ είναι σύντομα οι σκέψει μου και θα εκφράσουμε και εμεί τι απόψει μα με τροπολογίε. Ο Ζαν Πολ Μπεσέτ για του Πρασίνου. Voilà, merci. Ε, souhaiterions... Ευχαριστώ. Θα θέλαμε να εμπλουτίσουμε αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης. Μόνο αυτό καθορίζοντας το αντικείμενο της έρευνας και καινοτομίας. Για να το καθορίσουμε, για να βρούμε κάτι, πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώ ψάχνουμε. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, για να καταστεί η έρευνα η καινοτομία μια δυνατότητα και μια ευκαιρία ε, για τις περιφερειές μας, θα πρέπει να κατευθυνθούν προς ένα ε, πιο συγκεκριμένο και καθορισμένο αντικείμενο και περιεχόμενο. Συγκεκριμένα, θα ήθελα να κατευθυνθούμε προς την γενικότερη έννοια της αιφόρου ε, ανάπτυξης, της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτή η καινοτομία λοιπόν θα πρέπει να έχει αυτό το προσανατολισμό να αποτελέσει δηλαδή εργαλείο για την γενικότερη ε, αναπροσαρμογή όλων ε, των επιστημών και όλων των δραστηριοτήτων μας. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτόν τον προσανατολισμό και αυτή την κατεύθυνση και σε αυτό το πνεύμα θα υποβάλουμε μία τροπολογία για να καθορίσουμε μία πιο κατάλληλη ε, κατεύθυνση για, αυτή την, για αυτό το σχέδιο γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Εντάξει, ας περάσουμε τώρα στου συναδέλφου που, θέλουν, να πάρουν το λόγο. Ο Φραντσέσκο Ντάντζελη. Ευχαριστώ. Σημερίζομαι την τοποθέτηση του συναδέλφου Βίνκλερ, πιο συγκεκριμένα την ανάγκη να προωθήσουμε περισσότερο την έρευνα, την καινοτομία και να βασιστούμε πάνω απ' όλα ε, στις έξοχες επιδόσεις σε περιφερειακό επίπεδο, στην αριστεία. Εντάχει τέσσερα σημεία που θεωρώ ότι έχουν προτεραιότητα. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη συνοχή μεταξύ των στόχων που καθορίζονται στρατηγική για το 2020 και των στόχων για την έρευνα και την καινοτομία. Και είναι ευκταίο να υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή μεγατή των κάθετων νομοθεσιών και των τομεακών για την έγκριση ε, του μελλοντικού προγράμματος πλαισίου. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Δεύτερον, χρειάζεται μεγαλύτερη απλούστευση κυρίω όσον αφορά τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, εντοπίζοντα θέματα πιο προσβάσιμα ε, και δεν θα είναι κατακαιρματισμένα τα μέτρα σε αυτόν τον τομέα και θα είναι πιο εύκολη προσβάσιμα. Πρέπει να μειωθεί μετά και η ε, γραφειοκρατία για την πρόσβαση στα ποσά μέσω της ηλεκτρονικής υπογραφής, παραδείγματι. Και τέταρτο θέμα, πρέπει να ευνοηθεί η ανταλλαγή των βελτίστων πρακτικών και των ευφυών κριτηρίων στα πλαίσια των δημοσίων ε, προμηθειών. Αυτά λοιπόν είναι τα τέσσερα βασικά σημεία. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σμόκοβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Για αυτή την ε, ανταλλαγή απόψεων που διασφαλίζει αυτή την πτυχή, πώς η έρευνα, η ανάπτυξη, η καινοτομία έχουν επιπτώσεις ε, και είναι σημαντικές για την περιφερειακή ανάπτυξη. Και συμφωνώ προσωπικά με την άποψη αυτή και θέλω ακριβώς στο σημείο 5 να αναφερθώ, στο εδάφιο 5. Θα έπρεπε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ένταξή τους, η ενσωμάτωσή τους στην έρευνα και ανάπτυξη να υποστηριχθεί. Ανήκουν σε αυτό το πλαίσιο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να αποτελούν τμήμα της διασύνδεσης, μέρος της διασύνδεσης με το πρακτικό επίπεδο εφαρμογής και υλοποίησης των μέτρων. Μία ερώτηση θέλω να διατυπώσω. Κύριε Σιγητά, στο εδάφιο 2 αναφέρεται ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι καινοτομία για τις περιφέρειες. Και αυτή η καινοτομία πρέπει να είναι δεσμευτικού χαρακτήρα. Συμφωνώ. Ένας στόχος της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020 εντάσσει, εντάσσεται ακριβώς σε αυτό το σημείο. 3% αναφέρεται ποσοστό του ΑΕΠ που θέλουμε να είναι δεσμευτικού χαρακτήρα για να είμαστε αποτελεσματικοί στις δράσεις μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θεωρώ ότι πρόκειται για μια καλή γνωμοδότηση του συναδέλφου. Για ένα σημείο ε, είχαμε μία ε, συνεδρίαση ως ε, ΕΛΚ για τη σύνδεση μεταξύ του νέου στρατηγικού πλαισίου και τα σχετικά πεδία και εκεί κοιτάξαμε λεπτομερώς τι μπορεί να κάνει το Ταμείο Συνοχής για την δημιουργία υποδομών, ε, ερευνητικών υποδομών. Δεν... Ήδη το Ταμείο Συνοχής έχει αναλάβει σημαντικό μέρος των δαπανών, αλλά εμείς μιλάμε για το ίδιο το πρόγραμμα αυτό. 90% του, των προϋπολογισμών ε, του προπολογισμού αυτού ε, ξεκινά από τα κράτη-μέλη μας. Αυτό δεν έχει σχέση με τους ε, στόχους, με, το, με την πολιτική συνοχής. αυτό οφείλεται καθαρά και μόνο στο κριτήριο excellence της αριστείας. Και η γνωμοδότηση αυτή σωστά παρουσιάζει το ζήτημα. Ο στόχος δεν πρέπει να είναι αυτό που γίνεται και στην έκθεση Ρίγα ότι πρέπει να διπλασιάσουμε δηλαδή την έρευνα. Και έτσι θα επιλυθούν τα προβλήματα. Όχι, δεν γίνεται αυτή η σύνδεση, ε, ο λόγος 90-10, 90%-10% να επιληθεί με την ε, ε χορήγηση περαιτέρω κονδυλίων. θα πρέπει να υπάρχει ακριβή διατύπωση που να λέει ότι ακόμα και από την πλευρά του προγράμματος NLA να τίθεται προτεραιότητα εξέβρεση μια ισορροπία στην Ευρώπη σε αυτό το τομέα. Και μετά μπορούμε να εξετάσουμε αυτή τη διατύπωση δεν λέμε ότι πρέπει να υπάρχει περαιτέρω χρηματοδότηση, πρέπει να υπάρχει καλύτερη κατανομή των ε, κονδυλίων. Θα πρέπει λοιπόν να ε, επεκτείνουμε περαιτέρω σε ό,τι σε αυτό το σημείο. Για το Regions of Knowledge. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ε, συμπεριλαμβάνεται στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Είναι το μοναδικό περιφερειακό ζήτημα. Εδώ μιλάμε για smart specialization. Αυτά θα πρέπει να τα συνδυάσουμε. Στο πλαίσιο αυτής της ε, smart specialization, της εφηούς ε, εξειδίκευσης, ε, και υπάρχει αυτή την εβδομάδα μια διήμερη συνεδρίαση για αυτό το σημείο, να διατηρήσουμε και να εξασφαλίσουμε την τήρηση αυτή τη ε, διάσταση. Ε, τα έχω θέσει αυτά τα ζητήματα βεβαίω και στην Επιτροπή Ήτρε, αλλά και εδώ θα πρέπει να αναφερθούμε σε αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μπλάσακ. Ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι, συμφωνώ και είμαι ικανοποιημένο με αυτή την πρόταση που με θετικό τρόπο επικεντρώνεται στα ουσιοδέστερα προβλήματα. Σε αυτόν τον επιμερισμό βλέπω κάποιου τομεί, Ο πρώτο τομέα είναι τα κέντρα των επιδόσεων. Η δημιουργία ομαδοποιήσεων και κατηγοριοποιήσεων. International clusters και ο συντονισμός είναι σημαντική πτυχή. Απ' την άλλη πλευρά βλέπω υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και υποστήριξη μέσω κονδυλίων για την έρευνα και τις επιστήμες. Πιστεύω ότι αν θέλουμε πραγματικά να πετύχουμε αυτούς τους στόχους είναι αναγκαίο τα στοιχεία 1, 5 και 6 να διασυνδεθούν και να είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Η σκοπιμότητα αυτή πρέπει να είναι δεσμευτικού χαρακτήρα. Στα προγράμματα περιφερικής ανάπτυξης πρέπει να είναι δεδομένη η διαφοροποίηση αυτών των προτεραιοτήτων και η διαδικτύωσή τους, ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ενδιαφερθούν, να ζητήσουν, να τύχουν ε, να, να τους δοθούν αυτά τα κονδύλια ώστε να συμμετάσχουν. Και το cross-financing, η διασταυρούμενη χρηματοδότηση, είναι μια ενδιαφέρουσα προοπτική σε αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, χαιρετίζω την έκθεση αυτή. Νομίζω ότι ήταν πολύ αναγκαία και είναι κατάλληλη στιγμή να συζητήσουμε την ανάπτυξη στα πλαίσια της πολιτικής ε, συνοχής, η οικονομική ανάπτυξη ε, μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω ε, αύξησης αγοράς είτε μέσω της έρευνας της καινοτομίας και της ανάπτυξης. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ανάπτυξη της αγοράς, για επέκταση της αγοράς. Νομίζω ότι υπάρχουν περιορισμένα όρια όσον αφορά τις ευρωπαϊκές αγορές σε αυτή τη φάση. Γι' αυτό η έρευνα, η ανάπτυξη και η καινοτομία θα πρέπει να είναι ο δρόμος θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον για τις πολιτικές μας για να τονώσουμε την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει αυτό τον παράγοντα να τον λάβουμε υπόψη στη διαμόρφωση της πολιτικής συνοχής, δοθέντως ότι υπάρχουν τόσες πολλές ανισότητες μεταξύ των διαφόρων περιφερειών. Αυτό που θα ήθελα να υπογραμμίσω εδώ είναι το ότι κάποιες κυβερνήσεις τώρα δεν γνωρίζουν πολύ καλά τις συγκεκριμένες δράσεις που θα πρέπει να δρομολογήσουν τόσο ώστε να τονώσουν την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία στις χώρες τους μέσω φορολογικών μέτρων, μέσω εκστρατιών ενημερώσεως ή μέσω άλλων δημιουργικών τρόπων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ώστε να συμμετάσχουν ενεργά στην επίτευξη του στόχου αυτού. Και γι' αυτό το ερώτημά μου είναι το εξή. Εάν εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κάνουμε κάτι για να τονώσουμε, να σπρώξουμε τις κυβερνήσεις. Αν βρούμε κάποιο κατάλληλο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, ούτω ώστε μάλλον να ενθαρρύνουμε τις ιδιωτικές επιχειρήσεις να επενδύσουν περισσότερο στην έρευνα και την καινοτομία. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Υπάρχει και μια άλλη πτυχή που αναφέρθηκε και δεν θα πρέπει να την ε, λησμονούμε. Πρέπει να καθορίσουμε ξεκάθαρα τι είναι η καινοτομία σε αυτή τη φάση δεν γνωρίζουμε πραγματικά αν η καινοτομία ε, συμπεριλαμβάνει το κόστος έναρξης μιας επιχείρησης ή όχι. Και υπάρχουν προβλήματα με τον ορισμό, διότι ερμηνεύεται ποικιλότροπα από τα διάφορα κράτη-μέλη. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ο όρος αυτός και στο Κοινοβούλιο και εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Χέρμαν, θες να απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχήν να ευχαριστήσω πρώτα για τις τοποθετήσεις σας και για τα, τις προτάσεις σας. Από τα όσα είπατε και προαναγγείλατε, μπορώ να κατανοήσω ότι με τροπολογίες θα αντιμετωπιστεί το θέμα ώστε να καταφέρουμε στις διαβουλεύσεις που θα απομένουν να καταλήξουμε σε μια σαφή τοποθέτηση και να συνεισφέρουμε για την περιφερειακή ανάπτυξη με αυτόν τον τρόπο. Λόγω του ότι πιέζει ο χρόνος, δύο-τρία θέματα επιλέγω στα οποία θα υπησέλθω. Χαίρομαι αφενός ότι αυτός ο τομέας της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι κάτι που το συμμερίζονται όλοι. Είναι πολύ σημαντικό διότι διαδραματίζει μεγάλο ρόλο στις περιφέρειες Χρειαζόμαστε την αηφορία που πρέπει να διασφαλιστεί και η διασύνδεση των, επιμέρων, των επιμέρους σημείων είναι σημαντική για να πετύχουμε κάτι από αυτά που θέλουμε. Για τα 3% ποσοστό Πιστεύω ότι είναι σημαντικό η προτεραιότητα να καθορίζεται οι προτεραιότητες από πλευράς μας και έχουμε πολύ φιλόδοξους στόχους όπως 3% του προϋπολογισμού αλλά να αναγνωρίσουμε ότι αυτοί οι φιλόδοξοι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μόνο αν συνδράμουμε τις περιφέρειες και τις υποστηρίξουμε και αυτό μπορεί να γίνει με σαφή στοχοθέτηση προτεραιοτήτων και εμπλοκή όλων εκείνων που χρειάζονται ώστε να καταλήξουμε σε αυτό το αποτέλεσμα, ώστε να κάνουμε το σωστό βήμα προς τον τελικό στόχο για τη στρατηγική 2020 και να επιτευχθεί ο στόχος μας. Γι' αυτό χαίρομαι για αυτές τις συζητήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Uh, ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει εδώ πέρα να καθορίσουμε την προθεσμία για, τις, ε, για την υποβολή των απολογιών. Είναι πολύ σύντομη αυτή η προθεσμία, μέχρι αύριο δηλαδή στις 6 το απόγευμα. Έχετε περιθώριο. Θα περάσουμε στην γνωμοδότηση για Νόλ Όλμπριχτ. Δημοσιονομικοί κανόνε που εφαρμόζονται στον ετήσιο προπολογισμό τη Ένωση. Θα ψηφιστεί σήμερα το απόγευμα. Επομένω, να δώσω τώρα τη δυνατότητα στο Γιάν ε, να μας παρουσιάσει αν έχει οποιαδήποτε άλλα σχόλια. Ευχαριστώ. Ήθελα να σας παρουσιάσω αυτή την ε, γνωμοδότηση. Μιλάμε για τον ε, κανονισμό ε, για τον οποίο προετοιμάζεται μία έκθεση στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου. Ο εισηγητής πρέπει να ε, προετοιμάσει την ε, έκθεση που αποτελεί κατάλογο των τροπολογιών στο αρχικό σχέδιο που έχει προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε ένα επίσημο έγγραφο, το σχέδιο κανονισμού που προετοίμασε η Επιτροπή. Σε μεταγενέστερο στάδιο όμως έχουμε και την τροποποιημένη εκδοχή αλλά και την θέση του Συμβουλίου. Γνωρίζουμε και τη θέση του εισηγητή. Είχα τη δυνατότητα να συμμετάσχω στην λεγόμενη ομάδα εργασίας και ξέρω ότι και η θέση του εισηγητή αλλάζει. Εγώ πρότεινα να προετοιμάσουμε τον κατάλογο των τροπολογιών για το αρχικό κείμενο, παράλληλα όμως να βρισκόμαστε σε επαφή με τον εισηγητή και να του ζητήσουμε να συμπεριλάβει τις τροπολογίες που θα υιοθετηθούν από την Επιτροπή μας στην έκθεσή της. Ιδάλλως, η ε, τροπολογίες θα ψηφιστούν ε, ε, διαζευτικά. δηλαδή θα πρέπει να επιλέξουμε ή αυτές ε, της ε, εισηγήτριας είτε τις δικές μας. Σε μια γνωμοδότηση λοιπόν που προετοιμάζεται για την Επιτροπή Ρέτζι, εγώ εστίασα σε δύο παραγράφους. Η μία αφορά την έννοια του αποδεκτού ε, κινδύνου σφάλματος και υπάρχει μια συζήτηση που συνεχίζεται μεταξύ διαφόρων φορέων για το πώς να χρησιμοποιήσουμε ε, τον όρο του σφάλματος, του αποδεκτού κινδύνου σφάλματος ε, και καθεξής. Είναι περίπλοκο το ζήτημα ε, υπάρχει συζήτηση μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, αλλά δεν έχουν καταλήξει σε μια συμφωνία. Γι' αυτό το Συμβούλιο πρότεινε να χρησιμοποιήσουμε έναν άλλον όρο. Tolerable level of compliance, αποδεκτό ε, όριο συμμόρφωσης, που συμπεριλαμβάνει και το αποδεκτό όριο σφάλματος. Ε, δεν είναι μόνο μια τεχνική παρατήρηση, αυτό επηρεάζει και την αξιολόγηση της αποδοτικότητα, για παράδειγμα, της πολιτικής συνοχής. Γιατί στο τέλος του ελεγκτικού συνέδριου έχουμε την έκθεση για την πολιτική συνοχή και εκεί έχουμε πληροφορίες για το επίπεδο σφάλματος. Και τίθεται το ερώτημα ποιο επίπεδο ε, μπορούν να θεωρηθούν αποδεκτά. Αυτή είναι η παράγραφος στην οποία αναφέρθηκα στην ε, γνωμοδότησή μου, αλλά κυρίως και η παράγραφος 56 του ε, ε, χρηματοδοτικού κανονισμού για την επιμερισμένη διαχείριση. Στην γνωμοδότησή μου εγώ πρότεινα να αναδιαρθρώσουμε ολόκληρη την παράγραφο, γιατί δεν ήταν καθόλου ξεκάθαρο στην αρχή. Μάλλον δεν ήταν ξεκαθαρή διατύπωση. Θα πρέπει λοιπόν να δείξουμε αυτή την κατανομή ευθυνών και αρμοδιοτήτων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα κράτη-μέλη, στα, στον πιστοποιημένο φορέα που θα ορίσουν τα κράτη-μέλη και μετά τις αρμοδιότητες των πιστοποιημένων φορέων που σήμερα αποκαλούμε ε, αρχές διαχείρισης. Υπάρχει λοιπόν ξεκάθαρη διάκριση μεταξύ των ε, ρόλων του, της Επιτροπής των Κρατών Μελών, του ε, φορέα που χορηγεί την πιστοποίηση, του πιστοποιημένου φορέα και το καθεξής. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να, καταστεί όσο δυνατόν πιο σαφές και θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την εφαρμογή της ε, πολιτικής συνοχής. συνεχίζονται συζητήσεις και για την δήλωση ασφάλειας, Declaration of Assurance. Δύο στοιχεία αναφέρονται. Πρώτον, έχουμε την διαχειριστική δήλωση που θα προετοιμάσουν οι πιστοποιημένοι φορείς και μάλιστα οι διαχειριστικές αρχές, οι διοικητικές αρχές και μετά έχουμε και τον πολιτικό διάλογο για την εθνική δήλωση Και εδώ υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και στο Κοινοβούλιο. Γι' αυτό και εγώ δεν ε, εστίασα στην εθνική δήλωση. Ακόμα και η συγγήτρια στην ε, γνωμοδότησή της θα κάνει τις απαραίτητες αλλαγές για το μέλλον. Και δεν αναφέρεται στην απόφαση σήμερα. Ένα στοιχείο το οποίο λείπει στη δική μου γνωμοδότηση είναι ότι δεν ε, ανέφερα, το αποδεκτό επίπεδο σφάλματος, όχι αποδεκτό κίνδυνο, αλλά επίπεδο που ε, θα προταθεί από την εισηγήτρια και δεν είχε προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ακόμα περισσότερο δεν είχε προταθεί και από το Συμβούλιο. Η εισηγήτρια ε, χρησιμοποίησε το ε, επίπεδο το συντελεστή 2% ως αποτελεσ... αποδεκτό επίπεδο σφάλματος. Κατά τη γνώμη μου, ε, το ελεγκτικό συνέδριο έχει τους κανόνες του και είναι μάλιστα ιδιαίτερα αυστηροί και τα επίπεδα αυτά έχουν ε, καθοριστεί ε, με τόσο αυστηρό τρόπο που δεν δείχνουν την πολυπλοκότητα των διαφόρων μέτρων που συμπεριλαμβάνονται στην πολιτική συνοχή. Όταν αναφέραμε εμεί το συνελεστή 2% για αποδεκτό επίπεδο σφάλματο, τίθεται και το ζήτημα των κυρώσεων που θα έχουμε στο μέλλον στο Κοινοβούλιο. Δηλαδή, αν υπερβούμε το 2%, αυτό τι σημαίνει δεν θα δώσουμε αυτό το ρόλο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή θα έχουμε αρνητική γνωμοδότηση για κάτι. Αλλά στην πράξη δεν θα αλλάξει τίποτα γιατί το καθήκον αυτό είναι τόσο περίπλοκο. Γι' αυτό δεν έχω ε, καθορίσει συγκεκριμένο συντελεστή. Υπήρξαν αρκετέ τροπολογίε των συναδέλφων από την Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξη. Ορισμένε από αυτέ έγιναν ε, δεκτέ χωρί κάποιο πρόβλημα. Άλλε αφορούσαν τη δομή οι προτάσει των μέλων τη Επιτροπή αναφέρονταν σε κάποιο άλλο σημείο και εγώ επειδή πρότεινα την γενικότερη αναδιάρθρωση της ε, παραγράφου υπήρξε μια παρανόηση. Ε, έχουμε όμως δύο συμβαστικές τροπολογίες. Συμφωνήσαμε πάνω κάτω στο περιεχόμενο και ελπίζω ότι αν ψηφίσουμε σήμερα την ε, γνωμοδότηση αυτή θα ληφθεί υπόψη από την εισηγήτρια για να την έχει στο δικό της κείμενο. Βεβαίω και θα ψηφιστεί στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου ε, ως ε, τρο, γνωμοδότηση της Ρέτζη, αλλά δεν είμαι και ιδιαίτερα αισιόδοξο. Βρίσκομαι σε συνεχή επαφή με την εισηγήτρια και ελπίζω αν έχουμε μια συμφωνία εδώ πέρα να συμπεριληφθεί στην πρότασή της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Γκάιερ για τους σοσιαλιστές ε, του Σκιώδης. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Όλμπρεχτ, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για το έργο που επιτελέσατε για μια περιεκτική πλήρη γνωμοδότηση. Μια ολόκληρη σειρά τροπολογιών έχω για τις προτάσεις του συναδέφου Όλμπρεχτ. Όχι επειδή δεν συμφωνώ με την προσέγγιση του κυρίου Όλμπρεχτ ή δυσπιστώ εναντί αυτής, αλλά επειδή Ω συντονιστή των Σοσιαλδημοκρατών στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού, αντιμετωπίζω τη δυσκολία μια θέση να μην την εγκαταλείψω που στην Επιτροπή Ελέγχου του προπολογισμού θα πρέπει να την ξαναϊοθετήσω. Και γι' αυτό θα με ρωτούσαν οι συνάδελφοι στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού πώς εγκατέλειψε αυτή τη θέση στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξη. Γι' αυτό χαίρομαι για τη δυνατότητα συμβιβασμών που είναι ε, μια δυνατότητα που έχουμε στη διάθεσή μας και θα ήθελα να επισέλθω σε κάποια σημεία τα οποία ίσως εξηγούν πού και γιατί καταλήγω σε άλλη αξιολόγηση εγώ από πλευράς μου σε κάποια θέματα. Το ένα είναι η άτυχη έννοια, η προσέγγιση του ανεκτού επίπεδου σφάλματος. Θέλω να υπενθυμίσω ότι αυτή η έννοια, θα το υπενθυμίσω στους συναδέλφους, στο ευρωσκεπτιστικό τμήμα του σώματος έχει οδηγήσει σε κάποια πολεμική αντιμετώπιση, σε κάποια επίμαχα θέματα. Δηλαδή λένε, κοιτάξτε, εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι καν αποφασισμένο σε σχέση με την καταπολέμηση σφαλμάτων όσον αφορά την Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού. Το έχουν εγκαταλείψει το θέμα και σε σχέση με αυτή την προσπάθεια υπάρχουν ατέλειες και κένα τα οποία διατυπώνονται κάθε χρόνο και δεν τα καταπολεμούν. Πρώτον, αυτό είναι σφαλμένη θέση. Δεύτερον, δεν είναι αποδεκτό και γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε το περιφερειακό κεφάλαιο του προϋπολογισμού να το δούμε πραγματικά σε κυριολεκτικούς όρους. Δηλαδή είναι ο τομέας εκείνος που έχει το υψηλότερο ποσοστό σφαλμάτων στην υλοποίηση των δράσεων του προϋπολογισμού. Και γι' αυτό οι επαΐοντες που βρίσκονται εδώ γνωρίζουν ότι αυτά τα σφάλματα οφείλονται στα κράτη-μέλη. Εκείνα κάνουν αυτά τα σφάλματα. Αυτό συνδέεται με τον περίπλοκο χαρακτήρα των κανόνων και κανονισμών, αλλά συνδέεται επίσης και εδώ δεν είναι εξαίρεση η χώρα μου, με το γεγονός ότι στα κράτη-μέλη η αντιμετώπιση ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι χαλαρή, πώς να το πω. Πολλές φορές είναι λιγότερο προσεκτική από εκείνη που θα έπρεπε. Υπό αυτό το σκηνικό η έννοια του αποδεκτού επίπεδου σφάλματος είναι ήδη κάτι επικίνδυνο. Στην παρουσίαση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού διορθώνει ο μιλητής τις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου απορρέει ότι υπάρχουν οριακές τιμές που ξεπερνούν πολλές φορές το κόστος των ελέγχων. Μπορεί κανείς να εξηγεί σε κάποιον ελεγκτή ότι δεν έχει νόημα να γίνονται δαπάνες δεκάδων χιλιάδων ευρώ για να αποκαλυφθεί ε, μια παρατυπία μερικών δεκάδων ευρώ ή κάποιων ευρώ. Με αυτή τη βάση η καποιον ευρω με αυτη Επιτροπή συνέταξε σε έγγραφα εργασίας και προβληματισμού από τα οποία μπορεί να δει κανεί ποια είναι η οριακή τιμή σε σχέση με το όφελος όσον αφορά ελεγκτικές δράσεις. Και μέσω των τριών διαφορετικών εγγράφων που έχουμε στη διάθεσή μας για αυτό το θέμα καταλήγουμε σε διαφορετικά αριθμητικά μεγέθη. Ο συνάδελφος Όλμπρεχτ ανέφερε και πάλι το 2%. Είναι το ποσοστό αυτό ανεκτού σφάλματος που δέχεται το ελεκτικό συνέδριο. Λέει οι άνθρωποι σφάλουν και υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσοστό σφάλματος που πρέπει να γίνεται δεκτό. Όμως δεν μπορεί κανείς να πει για αυτόν τον λόγο ότι δεν είναι ακριβής η εκτέλεση του προϋπολογισμού, γι' αυτό το ανεκτό αυτό επίπεδο φτάνει στα 2% και έχει και ένα πράσινο μήνυμα το οποίο αποστέλλεται. Δηλαδή ότι δεν, δεν διαπιστώθηκαν άλλα σφάλματα. Η Επιτροπή πέρα από αυτό το 2% ανάλογα με τους τομείς που εξετάζονται ξεπερνά το όριο αυτό. Δεν θα κερδίσαμε τίποτα όμως ε, συνάδελφοι αν ακολουθούσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή την αξιολόγηση. Διότι δεν έχει καθόλου υπόψη το ελεγκτικό συνέδριο να ανυψώσει, να ε, αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο το αποδεκτό επίπεδο σφάλματος. Όταν λέει το ελεγκτικό συνέδριο ότι το επίπεδο σφάλματος θα βρίσκεται σε συγκεκριμένο επίπεδο, θα λένε άλλοι βρισκόμαστε κάτω από αυτό, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχουμε το δίλημα, θα συμφωνήσουμε με το Ελεγκτικό Συνέδριο ή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και δεν θα επιλύαμε, δεν θα αντιμετωπίζαμε σωστά αυτό το πρόβλημα αν λέγαμε υπάρχει ένα αποδεκτό επίπεδο σφάλματος και τότε θα λέγαμε ε, αυτό που είμαστε ε, πρόθυμοι να αποδεχτούμε είναι ε, το σφάλμα που διατυπώνεται βρίσκεται κάτω από αυτό. Φυσικά οι άνθρωποι σφάλουν, αλλά υπάρχουν σφάλματα τα οποία δεν μπορούν να γίνονται αποδεκτά. Θέλουμε στο μέτρο του εφικτού να έχουμε μια εκτέλεση προϋπολογισμού σχεδόν χωρίς σφάλματα ή προσεγγίζοντας την απάλληψη σφαλμάτων. Αυτό είναι ο στόχος και είπαμε το πεδίο των αποδεκτών επιπέδων πρέπει να τεθεί στο περιθώριο και να πούμε ότι πρόκειται για μια διαφορετική έννοια, δηλαδή για την πιθανότητα σφάλματος υποστατιστικό πρίσμα. Αυτό είναι το ένα σημείο διαφοροποίησης. Το ένα σημείο όπου στην προσέγγιση του κυρίου Όλμπριχτ ακολουθώ μια άλλη προσέγγιση. Αιτιολογείται όμως αυτή η διαφορετική προσέγγιση από την δράση μου στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού σε σχέση με την προσέγγιση του κυρίου Όλμπρεχτ. Γι' αυτό διαφοροποιούμε από αυτόν. Το δεύτερο σημείο είναι το θέμα της εθνικής δήλωσης, διαχείρισης ή δήλωσης αξιοπιστίας. Αυτό είναι ένα από τα θέματα στην αντιπαράθεση με τη νέα δημοσιονομική τάξη πραγμάτων. Δίνουμε μάχη εδώ και χρόνια ώστε από τα κράτη-μέλη να υπάρχει μια δήλωση, διακήρυξη διαχείρισης από πλευρά τους που να προσυπογράφεται και να δεσμεύει τους πολιτικά υπεύθυνους και να πιστοποιείται από το Εθνικό Ελεγκτικό Συνέδριο. Και αυτό όχι επειδή είμαστε βιτσιόζοι ή έχουμε κάποιες αιμονές όσον αφορά τους ελέγχους, αλλά επειδή κάτι τέτοιο μια ολόκληρη σειρά ελέγχων θα, τους, θα την καθιστούσε, μια ολόκληρη δράση με ελέγχους θα την καθιστούσε περιττή. Αν είχαμε στην εκτέλεση των δράσεων των διαθροτικών ταμείων με νόμιμη διεργασία αυτά τα πιστοποιητικά από, τους, από τα Εθνικά Ελεγκτικά Συνέδρια, συνέδρια πιστοποιούμενα από τους πολιτικά υπεύθυνους θα είχαμε ένα μέσο μέσω του οποίου στα κράτη-μέλη θα μπορούσαμε να παρέμβουμε. Και έτσι θα μπορούσαμε, ας το πούμε έτσι, να απόσχουμε σε μεγάλο βαθμό από περαιτέρω ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό θα ήταν μεγάλη ελάφνηση μεγάλη ανακούφιση, αλλά καθιστά αναγκαίο αυτό όχι ένας ε, υπάλληλο μεσαίου επίπεδου να δρά και να πιστοποιεί αυτά, αλλά ένας υψηλά ιστάμενος αξιωματούχος σε πολιτικό επίπεδο που θα είναι υπεύθυνο πολιτικά και θα έχει κάτι να χάσει αν κάτι πάει στραβά. Και γι' αυτό η συνάδελφο Γκρέσλε που στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού και στην Επιτροπή Προπολογισμών μετά από πολλέ διαπραγματεύσει πιστεύει ότι το επίπεδο το υπουργικό είναι το σωστό επίπεδο πιστοποίηση. Και εγώ το βρίσκω σωστό αυτό. Και γι' αυτό στι τροπολογίε που έχω καταθέσει αυτή τη θέση υποστηρίζω και εγώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μάνα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ εκ μέρου τη ομάδα μου, λέει η κυρία Μάνερ, τον κύριο Όλμπρεχτ. Έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τι προτάσει που μα κάνετε. Ήθελα απλώ να αναφερθώ σε δύο ζητήματα και μόνο, τα οποία αφορούν την ομάδα μα, προβληματίζουν την ομάδα μα. Πρώτα απ' όλα, το θέμα του ε, φορέα πιστοποίησης, του γεκριμένου φορέα. Πώς αλλάζει ε, πώς μπορεί να αλλάξει το διοικητικό άχθος αυτό ο φορέας. Δεν θέλουμε να αυξήσουμε το διοικητικό άχθος στα κράτη-μέλη, αντιθέτως. Οι τροπολογίες δείχνουν ότι αυτός ο φορέας θα έχει σαφέστατο, σαφέστατες ευθύνες ελέγχου, διότι θα αυξήσει τους ε, ελέγχους. Στη Φιλανδία τουλάχιστον η έλεγχη όσον αφορά τα διεθνωτικά ταμεία ε, ίσως να οδηγήσουν σε συμπληρωματικούς ελέγχους, αύξηση αριθμού ελέγχων. Δεύτερον, ε, εντός του κανονισμού ε, μπαίνουμε σε πάρα πολλές λεπτομέρειες όσον αφορά διαφόρους τομείς πολιτικής. Αυτός ο κανονισμός μήπως γίνεται πάρα πολύ άκαμπτος, γίνει πολύ άκαμπτος στο μέλλον. Εν συντομία αυτές είναι οι δύο ερωτήσεις που είχα να θέσω. Ευχαριστώ. Θέλει κάποιος άλλος να πάρει το λόγο. Ιδεμή, Γιάν, μπορείς να απαντήσεις. Ευχαριστώ για τα σχόλια. Θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι. Συμφωνώ απόλυτα ότι η Εθνική Δήλωση Αξιοπιστίας θα πρέπει να συντάσσεται από κάποιον σε υπουργικό επίπεδο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το θέμα είναι αν τα κράτη-μέλη θα εγκρίνουν την εθνική δήλωση αξιοπιστίας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όσον αφορά την δήλωση διαχείρισης, αυτές οι δηλώσεις θα συνδέονται άμεσα με τους εγκεκριμένους φορείς, τους πιστοποιημένους φορείς. Αυτή θα είναι οι διοικητικές αρχές που αποκαλούμε, οι αρχές διαχείρισης όπως υποκαλούμε σήμερα. δεν προσθέτουμε διοικητικό βάρος. Έχουμε διαχειριστικές αρχές σήμερα. Οι διοικητικές αρχές μπορούν να ασχολούνται με πολλά επιχειρησιακά προγράμματα. Ποια είναι η αλλαγή. Πρώτον, σήμερα γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η, ε, α, δίνονται τα διαπιστευτήρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η έγκριση. Η διαφορά είναι ότι θα γίνεται από τον φορέα πιστοποίηση στον εθνικό, αλλά θα έχουμε τον ίδιο αριθμό φορέων διαχείρισης όπως σήμερα. Το θέμα είναι αν ο φορέας πιστοποίησης, έγκρισης θα είναι κάτι καινούριο. Δεν νομίζω. Θα είναι ένας από τους ισχύοντες φορείς του κράτους μέλους, των κρατών μελών, που θα εγκρίνει τις ε, αρχές διαχείρισης και αυτή, αυτός ο φορέας που θα εγκρίνει ένας για κάθε κράτος μέλος θα είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία των φορέων που εγκρίνει. Άρα δεν αυξάνεται το διοικητικό άκθος, αλλά είναι τα κράτη-μέλη εγκρίνουν και πιστοποιούν. Πρώτον. Και δεύτερον, ότι η δήλωση διαχείρισης που προτείνεται θα συντάσσεται από τους συγκεκριμένους φορείς. και θα γίνει του χρόνου το Μάρτιο όπως προτείνεται. Το θέμα ε, είναι κατά πόσο αυτή η αλλαγή θα μειώσει τη διάρκεια για τη χορήγηση της απαλλαγής. Η απάντηση είναι όχι, ίσως κατά ένα μήνα να μειωθεί η διάρκεια τη της διαδικασίας απαλλαγής. Δυστυχώς είναι δύσκολο η απαλλαγή να γίνει μετά το, το χρόνο μετά το χρόνο που ελήφθη υπόψη. Δηλαδή η απαλλαγή το 2010 να γίνει το 2011. Έχουμε απαλλαγή του 2010 που γίνει το 2012. Και η αλλαγή του κανονισμού δεν θα βραχύνει την όλη διαδικασία. Είναι αδύνατον λόγω των αιτήσεων εκθήσεων, λόγω του ελεκτικού συνεδρίου κλπ. κλπ. Αυτές οι αλλαγές πρέπει να πλουστεύσουν τη διαδικασία εντός των κρατών μελών, θα δοθούν σαφείς ευθύνες στους φορείς πιστοποίησης και στους εγκρινόμενους φορείς, αλλά δεν, ε, δεν αλλάζει την κατάσταση την απόφαση για την έγκριση της εθνικής δήλωσης. Η κυβέρνηση ή το Υπουργείο πρέπει να υπογράψει τη δήλωση. Δεν είναι η ίδια η δήλωση. Θα έχουμε τη δήλωση διαχείρισης από τη μία σε επίπεδο των φορέων των εγκεκριμένων και ενδεχομένως εθνική δήλωση σε επίπεδο κυβερνητικό. Αυτό δεν έχει αποφασιστεί ακόμα όμως. Ευχαριστώ. Δεν, αν δεν υπάρχουν άλλες χώρες, υπενθυμίσω ότι σήμερα το απόγευμα θα ψηφίσουμε και αυτή την έκθεση και εδώ κλείνουμε τη συνεδρίαση και θα ήθελα να ζητήσω από τους συντονιστές να παραμείνουν. Όλοι οι άλλοι συνάδελφοι παρακαλώ το ταχύτερο δυνατόν να αποχωρήσετε για να ξεκινήσει η συνεδρίαση των συντονιστών γιατί έχουμε καθυστερήσει πολύ.